Sí, sí, pasa nada. Okay. Let's start again. Excuse me. We are starting. Ας ε, ξεκινήσουμε λοιπόν. Παρακαλώ, καθίστε. Το πρώτο σημείο για σήμερα το απόγευμα είναι οι σημερινές αποφάσεις των συντονιστών. Ο Πρόεδρος ε, θα μιλήσει με τους Προέδρους ε, της ΕΜΒΗ και ΑΓΡΙ για να βρεθεί μια λύση σχετικά με την ακρόαση, απανακτήμηση των ε, πληθυσμών των λύκων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Επίση, εγκρίθηκε το σχέδιο ημερήσιας διάταξη ε, για τη συνάντησή μας τον Νοέμβρη. Η διαδικασία επίγοντος ε, θα εφαρμοστεί στην αναφορά 084 του 2019. Οι αναφορέ 0271 του 2019 και 0386 του 2018 και 0174 του 2018 και η 194 του 17 θα προσθεθούν στην ημερήσια διάταξη του Νοεμβρίου. Άνταμ Κόσα και Άλεξ Σαλίμπα είναι αυτοί που ορίστηκαν ως εκπρόσωποι της ΠΕΤΗ ε, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο ε, ε, του, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία. Μασιμιλιάνος Μερίλιο είναι ο εκπρόσωπος για το δίκτυο ισότητας των φύλων. Επίσης, ε, εγκρίθηκε ο σχεδιασμός για τις συναντήσεις του 2020. Επίσης, θα συντάξουμε γνωμοδότηση στην έκθεση της Γιούρη «Παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού ε, του Ευρωπαϊκού Δικαίου με εισηγητή από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Τρεις ακροάσεις θα λάβουν μέρος στο ε, χώρα, συγγνώμη, το πρώτο εξάμεινο του 2020, η πρώτη για τα πλαστικά και διαχείριση αποβλήτων, η δεύτερη για τα δικαιώματα των καταναλωτών στον τομέα της αεροπλοείας και σε περίπτωση που ε, γίνει το Δεκέμβριο του 19 η ακρόαση για τους λύκους, θα γίνει και μία τρίτη ακρόαση για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τους ε, αγρότες ε, με δίκαιο και ισότιμο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Δύο επισκέψεις, το πρώτο ήμιση του 2020, Βουλγαρία την εβδομάδα 24-28 Φεβρουαρίου, Πολωνία την εβδομάδα 18-22 Μαΐου. Επίσης, ε, τρίτη ε, επίσκεψη στη Σλοβακία εγκρίθηκε, ενώ άλλες δύο όχι. Τα σημεία 10 και 11 της μερίσιας διάταξης ε, θα, τα, ε, θα τα κάνουμε με τη γραπτή διαδικασία. Ωραία, πάμε στο επόμενο θέμα. Αλλάζω και θα μιλήσω ισπανικά. We are... Περνάμε στο σημείο 12. Έχουμε διάφορες αναφορές εδώ. Η 545-2015, η 629-2016, η 1068 του 17, 1141 του 17, 1188 του 17, 1231 του 17, 0011 του 18, 0149 του 18, 0412 του 18, 1064 του 18, 0256 του 19. Όλες αυτές για την μεταφορά των ζώων που προορίζονται για σφαγή. Προστασία των ζώων σε συνδεόμενες ε, ε, μεταφορές και παρόμοια θέματα. Εξαγωγή ζώων των ζώων. Όλα αυτά έχουν σχέση με την μεταφορά ζώων που προορίζονται για σφαγή. Η κυρία Μανουέλα Τζακομίν είναι εδώ, είναι μία από τις αναφέρουσες, της 12.31 ε, του 17 συγκεκριμένα, εκπροσωπεί ε, την Animal Welfare Foundation. Καλ, την καλωσορίζω, θα σας δώσουμε πέντε λεπτά για να μας εξηγήσετε την αναφορά σας. Eh, eh, Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. όπω γνωρίζετε, την τελευταία φορά που συζητήθηκε η αναφορά μου τον Ιούλιο του 2018 η Επιτροπή αποφάσισε να την κρατήσει ανοιχτή στην Επιτροπή ε, και έγινε ένας έλεγχος στη Σλοβενία, Κροατία και Ισπανία ώστε να διαπιστωθεί πόσο καλά εφαρμόζεται ο κανονισμός 1205. Έγιναν λοιπόν οι έλεγχοι, εκδόθηκε η σχετική έκθεση και πρέπει να τονίσουμε τα αποτελέσματα, τα οποία είναι ιδιαίτερα, θορυ... ε, μας θορυβούν ιδιαίτερα. Σύμφωνα λοιπόν με την έκθεση που θέσαμε στην Επιτροπή τον Δεκέμβρη του 2017 υπήρχαν σημαντικές ε, παραβιάσεις όχι μόνο του κανονισμού 12 25 ε, αλλά και τον 882 του 2004 που ορίζει τους επίσημους ελέγχους. Είχαμε δύο επίσημα έγγραφα τα οποία στην ουσία δείχνουν ε, ποιοι είναι οι αρμόδιοι κτηνίατροι για τα σημεία εξόδου και ε, λένε επίσης ε, πως ε, θα έπρεπε να γίνουν έλεγχοι για να εγκριθούν τα σκάφη, όμως από ό,τι φαίνεται τελικά δεν συνάδουν με αυτά που ορίζονται στον κανονισμό 1205. Δεν γίνεται σεβαστό αυτό που ορίζεται σχετικά με το περιβάλλον και την ευζοία των ζώων. Και αυτά δεν είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, αυτές οι πρακτικές φαίνεται ότι είναι παγιωμένες. Μπορείτε να δείτε ακριβώς, να εξακριβώσετε πώς γίνεται αυτό. Το έχει εξακριβώσει η Επιτροπή, ε, διότι ε, στην ουσία αυτό που ε, φάνηκε από τους ελέγχους είναι ότι δεν γίνονται αρμόδιοι έλεγχοι. Και αυτό και για τα ταξίδια στη θάλασσα, αλλά και έτσι λοιπόν δεν μπορέσαμε να δούμε ποιος είναι υπεύθυνο ε, για την ευζοία των ζώων και για τη μεταφορά τους στη θάλασσα. Επίσης αυτό που εξακριβώθηκε με τους ελέγχους της Επιτροπής ε, σε πολλές περιπτώσεις ήταν ότι ο τελικός προορισμός Ε, που εγγράφεται είναι το λιμάνι της αναχώρησης. Αυτό φυσικά δεν συνάδει με την απόφαση του δικαστηρίου. Έτσι λοιπόν τα ζώα δεν προστατεύονται και οι κτηνίατροι στα σημεία εξόδου δεν έχουν ούτε την τεχνική γνώση ούτε την κατάρτιση για να επιθεωρήσουν ορθά τα σκάφη. Ε, είδαμε ε, σε κάποιες περιπτώσεις μια επιθεώρηση η οποία διήρκησε μόνο μία ώρα. Στη Σλοβενία και στην Κροατία δεν είχαμε ε, ταξινόμηση για τους διαρθρωτικούς ελέγχους των ε, σκαφών και στα κεντρικά γραφεία δεν υπάρχει καν άποψη και γνώση για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η έλεγχη. Αυτό λοιπόν δεν έχει να κάνει μόνο με την ευζοία των ζώων, αλλά και είναι και στρέβλωση του ανταγωνισμού, γιατί οι μεταφορείς ε, προτιμούν τα κράτη-μέλη που είναι πιο χαλαρά ως προς την εφαρμογή του κανονισμού. Αυτό που επίσης είναι ε, πολύ ε, Ενδεικτικό είναι ότι στην Ρουμανία 70.000 πρόβατα ε, εξήχθησαν και υπήρχαν ε, εκατοντάδες ε, από αυτά που μπλοκαρίστηκαν στα σύνορα και πέθαναν από τη ζέστη. Αυτό δείχνει ακριβώς ότι δεν εφαρμόζονται σωστά οι ευρωπαϊκοί κανόνες που έχουν να κάνουν με τη μεταφορά των ζώων και υπάρχουν και αποδείξεις που μας δείχνουν ότι ε, υπάρχει μια πολύ δεινή κατάσταση. Ε, τώρα να περιμένεις ε, σε ένα σκάφος μια, από μια τρίτη χώρα και να είσαι σε συνθήκες καταστροφικές, ε, πραγματικά αυτό δεν είναι αυτό που θέλουμε ε, ε, να δούμε για να πείσουμε την Επιτροπή πόσο επίγον είναι το θέμα και να ξεκινήσει η διαδικασία επί παραβάση. Φαίνεται ότι η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για την Ευζωία των Ζώων κατά τη μεταφορά πρέπει να γίνεται σεβαστή και με όσα είδαμε φοβάμαι ότι η Επιτροπή θα πρέπει να ξεκινήσει τη διαδικασία επί παραβάση εναντί αυτών των κρατών μελών για να μπορέσουμε να εγγυηθούμε ότι η νομοθεσία για την προστασία των ζώων και την ευζοία των ζώων εφαρμόζεται. Ο λόγος στην Κομισιόν. Άννα Ραμίρεθ Βέλα. Θα σας ε, ενημερώσω ε, χωρίζοντας, διαχωρίζοντας τις οδικές μεταφορές από θάλασσες μεταφορές ε, για τις ε, πιο πρόσφατες δράσεις που έχουμε αναλάβει. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, έτσι. Ήταν μία από τις προτεραιότητες της επιμερίας των ζώων. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια δουλέψαμε πάρα πολύ σε αυτό το ζήτημα. Όπως είπε η αναφέρουσα, ολοκληρώσαμε το εισερασίας μας και στις θάλασσες και τις οδικές μεταφορές αποφασίσαμε να προσθέσουμε και άλλες ε, επιθεωρήσεις την Ρουμανία και τη Γαλλία τον επόμενο χρόνο για τις θαλάσσιες μεταφορές. Ε, δύο αναφορές εκδόθηκαν ήδη, μία για τις θαλάσσιες, μία για τις οδικές μεταφορές. Ε, θα δημοσιευθούν έτοιμε και θα δημοσιευθούν τώρα που θα αναλάβει τα καθηκόντα της Νέα Κομισιόν. Τουλάχιστον 13 κράτη-μέλη ανέφεραν δράσεις για την απαγόρευση, κοινοποίηση της απαγόρευσης ε, μεταφορά ζώων όταν η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς. Ε, βλέπουμε μείωση της εξαγωγής ζών των ζώων μεταξύ Βουλγαρίας και Τουρκίας τα τελευταία χρόνια. Η περίοδος μεγιστο μέγιστου κινδύνου, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, το 2017 είχαμε πάνω από 160 φορτία Αυτά μειώθηκαν σε 965 το 2018 και το 2019 μόνο 556. Πολύ σημαντική μείωση του στερινούς ζεστούς μήνες. Επίσης έχουμε αυξήσει τον αριθμό, ε, ε, έχει μειωθεί ο αριθμός των κρατών μέλων που εξάγουν ζώα. Ε, Επίσης τώρα οι δευτερεύοντες ε, δρόμοι ε, που παλιότερα χρησιμοποιούνται για λίγες ώρες την ε, μέρα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ανοίγουν 24 ώρες έτσι ώστε να μπορέσουν να διακινούνται γρήγορα τα ζώα χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν στα σύνορα. Ε, οι μη κυβερνητικέ οργανώσει που ασχολούνται με αυτά τα θέματα μα ανέφεραν ότι φέτο στα βούλγαρο-τουρκικά σύνορα δεν είχαμε σημαντικά προβλήματα σε ό,τι αφορά τη μεταφορά των ζώων. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη δουλειά που έχουν κάνει όλοι. Ε, το ποσοστό συμμόρφωση μετριέται ω 97% αυτή τη στιγμή για τον κανονισμό. Μιλώ για, για την ε, οδική μεταφορά, χερσαίες μεταφορές ε, και είναι ε, υψηλότερο από ό,τι στο παρελθόν. Σε ό,τι αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, Τι θαλάσσιε μεταφορές όπως εξήγησε η ε, αναφέρουσα, ε, κάναμε και εδώ πολλέ επιθεωρήσεις. Ε, βρήκαμε παρατυπίες, έχουμε αναλάβει δράση. Ε, ήρθαμε σε επαφή με την Υπηρεσία Ασφάλεια στη Θάλασσα, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλεια στη Θάλασσα, που είναι στη Λισαβόνα ήδη κάνουν επιθεωρήσεις για περιβαλλοντικά θέματα και για θέματα ασφάλειας θάλασσα. Θα κάνουμε επιθεωρήσεις και για τη μεταφορά των ζώων, έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα, τα κράτη-μέλη να βελτιώσουν την κατάσταση. Θα τους παράσχουμε αρρωγή και βοήθεια. Η Ευρωπαϊκή Πρίση Θάλασσα στην ασφάλεια στη θάλασσα μας αναφέρει επίσης και εκεί βελτίωση της κατάστασης με βελτίωση των προδιαγραφών για τα σκάφη τα σκάφη δεν θα μπορούν στο μέλλον να διαλέξουν το κράτος μέλος το οποίο έχει την πιο χαλαρή εφαρμογή της νομοθεσίας προκειμένου να πάρουν άδεια. Θα απαγορεύσουμε δηλαδή αυτού του είδους τον ανταγωνισμό προς τα κάτω. Ήδη έχουμε προβλέψει οικονομικές διατάξεις για, την, για το επόμενο έτος με την υπηρεσία ασφάλεια θάλασσα θα ε, συζητάμε αυτή τη στιγμή τα τεχνικά μέτρα που θα ληφθούν από αρχέ του 2020. Είμαστε σε επαφή με τρίτε χώρε επίση που λαμβάνουν, εισάγουν ε, ζώντα ζώα μέσω θαλάσση. Έχουμε μια συμφωνία με το Ισραήλ, το οποίο δέχεται περίπου 6, κατά μέσο όρο μάλλον, 6 σκάφη τη βδομάδα. Ε, έχουν αρχίσει και μα στέλνουν πληροφορίε, feedback. Αυτό βοηθάει να βελτιώσουμε το σύστημα της Πορτογαλίας που εφαρμόζεται από την υπηρεσία στην Πορτογαλία, στη Λισαβόνα, γιατί με αυτόν τον ε, τρόπο εντοπίζουμε ακριβώς που είναι το πρόβλημα. Είναι η διανομή των ζώων, είναι ο καπετάνιος, είναι οι διαδικασίες. Αυτά. Πρόεδρος, θέλω να δώσω το λόγο στις πολιτικές ομάδες. Η κυρία Κίρτον. Thank you very much and, um, thank you. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και την αναφέρουσα, τους αναφέροντες που ήρθαν και πάλι σήμερα εδώ για να συζητήσουμε αυτό το σημαντικό θέμα. Το ζήτημα της μεταφοράς των ζών των ζών είναι κάτι που απασχολεί το Ευρωκοινοβούλιο εδώ και πάρα πολύ καιρό και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων αυτό το ζήτημα εγέρθη αμέσως μετά τις ευρωεκλογέ στην Ολομέλεια ως ζήτημα προτεραιότητας. Επομένως θεωρώ ότι είναι πεποίθηση του Ευρωκοινοβουλίου να επιμείνει στην πρόοδο αυτού του ζητήματος. Επίσης καλωσορίζουμε την έκθεση από την Επιτροπή σε ό,τι αφορά τις δράσεις που έχουν αναλάβει από την τελευταία φορά που εξετάσαμε τις αναφορές αυτές. Πιστεύω βεβαίως ότι υπάρχουν ακόμη ευρύτατες ανησυχίες ό,τι αφορά την καλή μεταχείριση των ζώων κατά την μεταφορά τους. Προσωπικά θα ήθελα να δω να τελειώσουν, να πάυσουν εντελώς οι μεταφορές ζών των ζώων και θεωρώ ότι ως αποτέλεσμα είναι σημαντικό να παραμείνουν ανοιχτέ οι αναφορές αυτές ώστε να εξακολουθήσουμε να πιέζουμε για περαιτέρω δράση. Ε, σε ένα πιο τοπικό, τώρα σε μια πιο τοπική διάσταση πιστεύω ότι είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε αυτό το ζήτημα για το οποίο αγωνιζόμαστε στο Ευρωκοινοβούλιο εδώ και πάρα πολλά χρόνια να χρησιμοποιείται με έναν πολύ κοινικό τρόπο από τον Πρωθυπουργό μας σήμερα στο Manchester στην ομιλία του στο συνέδριο των συντηρητικών όπου με ένα κοινικό τρόπο μίλησε για την μεταφορά των ζώων ως ένα καλό παράδειγμα για το πώς θα είναι να ζει κανείς στο Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς ένα deal. Επιστεύω ότι ως μέρος του Ευρωκοινοβουλίου προσωπικά και στην ομάδα καλής μεταχείρισης των ζώων ποτέ δεν με προσέγγισε κανείς από την κυβέρνηση της χώρας μου για να συζητήσουμε την απαγόρευση της μεταφοράς των ζώων και θεωρώ ότι πραγματικά είναι ιδιαίτερα κοινικό να αναμειγνύουμε αυτή την πολύ σημαντική εκστρατεία πραγματικά σε τακτικές που αφορούν στο Brexit και πραγματικά με θλίβει ότι αυτή ήταν μια επιλογή του Boris Johnson σήμερα. Τέλος, αν θέλουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση των ζών των ζών στην Ευρώπη, πρέπει να έχουμε πιο α, ισχυρούς κανονισμούς ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και η ιδέα ότι αν ε, αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο θα καταφέρουν να βελτιωθούν στον τομέα αυτό θεωρώ ότι είναι ε, εντελώς ψευδής και πραγματικά χωρίς καμία κεραιότητα. Πιστεύω ότι πρέπει να επιμείνω σε αυτό το θέμα γιατί ο Μπόρις Τζόνσον μόλις το είπε τρεις ώρες πριν στο Μάντσεστερ και θεωρώ ότι πρέπει να το θίξουμε σήμερα εδώ στο Ευρωκοινοβούλιο χρειαζόμαστε να έχουμε ισχυρού κανονισμούς σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυξημένου ελέγχου από την Επιτροπή, ώστε να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την κατάσταση για τα ζώντα ζώα όπου και αν βρίσκονται. Η ε, κυρία ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και στην αναφέρουσα για τις αναφορές που εξακολουθούν να, να προκύπτουν για μια εκ νέου ακρόαση. Δεν είναι νέο. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, μετά από πολλά χρόνια βρισκόμαστε σε αυτό το σημείο που να πρέπει να επαναλάβουμε το ίδιο επιχείρημα γιατί το ζήτημα δεν έχει επιληθεί παρά τις προσπάθειές μας. Οι πρωτοβουλίες που έχουν αναλυφθεί με σκοπό να βελτιώσουν τους ελέγχους και το σύστημα ελέγχου γενικότερα η πολιτική του Επιτρόπου, του αρμόδιου Επιτρόπου και επίσης το γεγονός μη συμμόρφωσης με τον ανάλογο κανονισμό είναι γεγονότα και είναι γεγονός ότι σήμερα οι αποτυχημένες προσπάθειες του Κοινοβουλίου να επιλύσουν αυτό το ζήτημα οφείλονται σε όλα αυτά. Θεωρούμε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να συζητήσουμε το ζήτημα αυτό εκτενώς, γιατί θεωρούμε ότι το, το κοινοβούλιο αυτό έχει επικρίνει την α, ολιγορία αρκετών κρατών μελών σε ό,τι αφορά το ζήτημα της μεταφοράς των ζώων. Σε, αυτό το, σε αυτή την καινούρια λοιπόν Ευρωβουλή είναι ύψης της σημασίας το ζήτημα αυτό. και της συγκεκριμένη επιτροπής. Έχουμε ασχοληθεί με ζητήματα πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τη διάρκεια του ταξιδιού, για παράδειγμα, τις συνθήκες του ταξιδιού και τις μεταφορές σε τρίτες χώρες. Ε, επομένως, οι κανονισμοί δεν θα πρέπει να αποτυγχάνουν να εφαρμόζονται. Δεν θα πρέπει αυτό να είναι μια επιλογή αποτυχία εφαρμογής των κανονισμών η εφαρμογή των κανονισμών σε τρίτες χώρες είναι κάτι το οποίο θα πρέπει εμείς να εξασφαλίσουμε. Θα πρέπει να δώσουμε το, το καλό παράδειγμα, θα πρέπει εμείς οι ίδιοι πρώτα απ' όλα να σεβόμαστε τα δικαιώματα των ζώων. Έχουμε έναν νέο επιτροπό τώρα και ελπίζουμε ότι πραγματικά θα κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζουμε ότι θα λάβει υπόψη τις αναφορές αυτές ο νέος Επίτροπος και θα παραμείνουν ανοιχτές οι αναφορές και οι εκθέσεις θα ρυθμιστούν, θα έρθουν στην προσοχή του υποψηφίου Επίτροπου. Κύριε κύριος ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ για την αναφορά, ευχαριστώ όλους τους αναφέροντες. Σε, ευρωπαϊκή, ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπάρχει ένα συγκεκριμένος κανονισμός ε, που βασίζεται στη θέση της, Επιτροπής, ε, της Επιστημονικής Επιτροπής για την προστασία του ζώνα και φαίνεται ότι αγνοείται μια βασική αρχή. Υπάρχει ένα βασανιστήριο στο οποίο υποβάλλονται τα φορτωμένα ζώα ε, και σε χώρες όπως και η Γερμανία για παράδειγμα μόνο το 1% των ζώων ελέγχονται και όταν υπάρχει κάποια παραβίαση τότε γίνονται γελίες ε, κυρώσεις, επιβάλλονται γελίες κυρώσεις ακόμα και όταν έχουμε μεταφορές μεταξύ των κρατών μελών ε, πρέπει να υπάρχει ένα μέγιστο 8 ωρών ε, στη μεταφορά και αυτό ε, δεν τηρείται πάντοτε. Ε, προτείνω λοιπόν να μείνει ανοιχτή η αναφορά και να συνεχιστεί η έρευνα, όπως ήδη ε, είπαν και οι συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Άουκεν. Ναι, ευχαριστώ. Σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα που έχουμε στο τραπέζι όλα τα χρόνια, από τότε που είμαι εγώ εδώ. Και πάντοτε ζητούμε να τεθούν ε, σε εφαρμογή οι κανόνες ε, για τις παραβιάσεις. Φαίνεται ότι δεν εφαρμόζονται οι κανόνες και ειδικά πραγματικά μετά από όλα όσα έχουμε ζήσει, πόσος καιρός ε, χρειάζεται, πόσες ώρες μπορεί ένα ζώο να περιμένει στα σύνορα, 8 ώρες για έναν έλεγχο, τι να πω, δεν είμαι σίγουρη για όλα αυτά. Και η Επιτροπή ε, θα πρέπει να επιμείνει. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι αυτό δεν παραβιάζεται. Ότι τα ζώα δεν βασανίζονται. Πρέπει να δούμε πραγματικά τι ισχύει, γιατί όταν βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν όταν φεύγουν τα ζώα από την Δανία και πάνε στη Γερμανία και μέχρι το, ε, να φτάσουν εκεί έχουν γίνει ακόμα και πεθαίνουν. Πραγματικά δεν το έχετε δει ποτέ. Τυχεροί είστε. Λοιπόν, ε, φεύγουν και πάνε σε φθηνά σφαγεία. Υπάρχουν πολλά, πολλές άσχημες εικόνες και όχι μόνο για τα ζώα. Δεν έχω πιστεί ότι το θέμα έχει επιληθεί και θέλω σίγουρα να είμαι σίγουρη ότι συμβαίνουν, ε, ότι αυτά που συμβαίνουν ελέγχονται. Γιατί πόσες ώρες έχουμε στο νόμο. Δεν είναι ότι όλα αυτά συμβαίνουν όταν βγαίνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βασικό πρόβλημα είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και για τους χείρους, ε, και για τα μοσχάρια, και για τα άλογα. Για όλα ισχύει. Πραγματικά μπορεί η Επιτροπή να μας διαβεβαιώσει ότι οι ανησυχίες μας ε, δεν ε, έχουν βάση και ότι είμαστε στη σωστό δρόμο και δεν χρειάζεται πια να ανησυχούμε και οι αναφέροντες μπορούν ε, να φύγουν και να πάνε στο σπιτάκι τους και ότι είναι ασφαλή τα ζώα μας. Κοιτάξτε, προσπάθω να το πιστέψω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορώ. Ο ε, Χούμπερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Επιτροπή. Η μεταφορά των ζώων στην Ευρώπη θα πρέπει να γίνεται με τα ύψιστα στάνταρ. Θα πρέπει να υπάρχουν οι βελτιστοί έλεγχοι όπως ε, ε, ορίζει η Κομισιόν και η Κομισιόν βασικά με βάση όλα αυτά ε, θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τις αναφορές που γίνονται προς, αυτό το, προς αυτή την κατεύθυνση. Ε, θα ήθελα λοιπόν ε, πραγματικά να έχουμε πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές των ζώων, διότι οι άνθρωποι που εργάζονται με τα ζώα δεν μιλούν για τα ζώα, εργάζονται με τα ζώα, προσπαθούν να κάνουν ό,τι καλύτερο είναι για τα ζώα ε, μιλάνε για τρίτα κράτη, για αναπτυξιακή βοήθεια σε τρίτα κράτη. Ε, μιλάμε για ε, ζώα τα οποία εκτρέφονται. Πραγματικά ε, στέλνουμε αυτή τη βοήθεια με σκοπό το καλύτερο να γίνει για τα ζώα. Αν υπάρχουν προβλήματα στη μεταφορά μέχρι κανείς να, να φτάσει σε αυτές τις χώρες και αν δεν ξέρει κανείς που βρίσκεται το ζώο κάθε στιγμή, πραγματικά ε, δεν ξέρω αν ε, έχει νόημα, γιατί υπάρχουν οι τεχνικές, υπάρχουν τα στάνταρ για να δούμε ακριβώς που βρίσκεται κάθε φορά το ζώο και να μπορούμε να ορίζουμε ακριβώς ε, ε, ποιες είναι οι συνθήκες. Εγώ θα έλεγα να κλείσει αυτή η Επιτροπή. Η 1680 ε, του 2017 έχει αντιμετωπιστεί και με γνωμοδότηση από την ΕΒΒ και την ΑΦΕΤ. Αυτή μπορεί να μείνει ανοιχτή. 11-18 από τη Γερμανία δεν έχει πάρει κάποια θέση από την Κομισιόν και υπάρχουν κα... αυτές οι δύο μπορούν να μείνουν ανοιχτές. Όλες οι υπόλοιπε μπορούν να κλείσουν λόγω της επαρκούς απάντησης της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο λόγος του κύριο Ράντου. Ράδε, συγγνώμη, λέει πρόεδρος. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε το πρόβλημα με τη μεταφορά των ζώων είναι υπαρκτό και είναι σοβαρό. Δεν ξέρω αν έχετε δει στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης τι γίνεται με τα ζώντα ζώα. Ένα τμήμα αυτών των ζώων χάνουν τη ζωή τους, πεθαίνουν ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που έχει ζέστη. Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι δεν είναι θέμα ελέγχου και ελληματικού ελέγχου. Χρειάζεται καλύτερη νομοθεσία και περισσότερη καλύτερη έλεγχη για τη μεταφορά των ζώων. Ειλικρινά, κάθε χρόνο χάνουμε πολλά ζώα εξαιτία τη ζέστης και μάλιστα υποφέρουν κιόλα. Κυρία Άουκεν. η παραγωγή χείρων στην Γερμανία μπορεί να αλλά όχι στη Δανία. Εγώ έχω δει βιομηχανική παραγωγή χείρων στη Δανία και δεν μπορώ να μιλήσω για ευζοία. Και δεν μπορώ να πω ότι η μεταφορά είναι καλύτερη από ότι η εκτροφή. Παραβιάζουν ένα σωρό ευρωπαϊκών νόμων. και χρειαζόμαστε να βεβαιωθούμε ότι οι κανόνες θα εφαρμόζονται. Δεν είμαι τόσο σίγουρος ότι η εκτροφή στη Γερμανία είναι τόσο καλή, αλλά σε κάθε περίπτωση. Στη Δανία το έχω δει και το έχω δει και σε πολλές άλλες χώρες ότι η κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Εντάξει, μακάρι η Γερμανία να είναι έτσι τόσο καλή. Αλλά θα πρέπει να κρατήσουμε ανοιχτές αναφορές αυτές και να εξασφαλίσουμε ότι εφαρμόζεται η νομοθεσία. Μπορεί να είμαι παραπληροφορημένη, αλλά πάντως πεπιπισμένη δεν είμαι. Also be Κυρία Τόμ, και εγώ λέω να κρατήσουμε ανοιχτέ αναφορέ. Δεν έχω πιστεί ότι το πρόβλημα έχει λυθεί κατά κάποιο τρόπο. ΟΚ. Ωραία. Άρα τώρα για δύο λεπτά ο λόγο στην κυρία Τζακομίνη, την αναφέρουσα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του Κοινοβουλίου που στηρίζουν την αναφορά και θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Επιτροπή που μας κατέδειξε τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει. Για μένα βεβαίως δεν είναι επαρκής. Από το 2016 ήδη βλέπουμε τα ίδια έγγραφα και τις ίδιες αποδείξεις του τι συμβαίνει παρά τις συστάσεις που έχουν γίνει σε κράτη-μέλη, το τι συμβαίνει στη Σλοβενία για παράδειγμα, οι συστάσεις δεν έχει γίνει follow-up. Βλέπουμε τι συνέβη το καλοκαίρι στη Ρουμανία παρά το γεγονός ότι οι επίτροποι εξέθεσαν τις απόψεις τους δημοσίους, παρόλα αυτά δεν είχαμε κανένα αποτέλεσμα πέρα από αυτά τα 70.000 ζώα που έφυγαν από τη χώρα σχετικά με τον κανονισμό του 2005. Γνωρίζω ότι κρατημέλη πραγματικά πρέπει να εφαρμόσουν τους κανονισμούς αυτούς, αλλά ε, τουλάχιστον τα τελευταία τρία χρόνια δεν έχουμε δει την επιβολή των κανονισμών. Επομένως δεν μπορούμε να μελήσουμε αυτά τα πολύ σοβαρά περιστατικά γιατί η ίδια η συνθήκη της Λισαβόνας το άρθρο 13 ορίζει ότι τα ζώα δεν είναι αντικείμενα, αλλά ζώντες οργανισμοί. Επομένως θέλω να ενθαρρύνω την Επιτροπή να δείξει πραγματικά πυγμή και θέληση, ούτω ώστε να μπορέσουν να ξεκινήσουν και συγκεκριμένες κυρώσεις απέναντι σε κάποια κράτη-μέλη. Και πάλι ακούσαμε στοιχεία σε ό,τι αφορά τεχνική πρόοδο και αυτό πραγματικά είναι φανταστικό. Θα ήταν όμως πολύ καλύτερα αν η τεχνική αυτή πρόοδος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί. Είναι λυπηρό ότι πολύ συχνά ακόμη και η Επιτροπή ε, διαπιστώνουν ότι τι στα σκάφη ανοίγουν το, τη θέρμανση, την ψήξη όποτε χρειάζεται. Πολύ λίγο χρησιμοποιούνται οι τεχνολογίες αυτές παρά την προοδό τους. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ και μας εξηγήσατε την αφορά σας. Ακούσαμε τα, την Κομισιόν, τα, τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων. Προτείνω να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά Περιμένουμε την αξιολόγηση της και τη δημοσίευση της γενικής έκθεσης ε, του 2019 και ζητούμε την Κομισιόν να μας ενημερώσει όταν ολοκληρωθεί αυτή η ενημέρωση και οι εκθέσεις της. Περνάμε στο σημείο 13. Αναφορά 1344-2012 της Ρομπέρτα Φορνασάρη, Ιταλική Σταγένεια, σχετικά με την κατάργηση της ζωοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, αναφορά 1581 του 13 του Ντανιέλ Μπέουκλερ, Μπεκλέ, Ντανιέλ Γαλλική Σταγέννη, σχετικά με την απαγόρευση των πειραμάτων σε ζώα. Αναφορά 0947 το 17 τη Τζούλια Μπέιν, Βρετανική Σταγένεια, εκ μέρου Τη ε, οργάνωσης ΠΕΤΑ φέρουσα 109.802 υπογραφέ σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωση τη καταλληλότητα και τη αποδοτικότητα του κανονιστικού πλαισίου του κανονισμού REACH και την απαγόρευση δοκιμών σε ζώα για την εφαρμογή του ε, κανονισμού REACH. Αν δεν κάνω λάθο, δύο από του αναφέροντε είναι εδώ, η κυρία Ρομπέρτα Φορνασάρη και η κυρία Τζούλια Μπέιν. Δίνω το λόγο για πέντε λεπτά σε κάθε μία από τις δύο αναφέρουσες, τις οποίες και καλωσορίζω. Κυρία Φορνασάρη στην αρχικά. Ευχαριστώ. Μου δίνετε το λόγο. Είναι δύσκολο να σας παρουσιάσω όλα τα στοιχεία τα που έχουμε συλλέξει σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Θα σας πω όμως ποια είναι τα βασικά προβλήματα. Τοξικότητα και έλλειψη αποτελεσματικότητα των φαρμάκων είναι ένα από αυτά. Ένα άλλο είναι η λανθασμένη επιλογή των ουσιών που συμπεριλαμβάνονται σε φάρμακα τα οποία τελικά δεν χρησιμεύουν. Οι κλινικές δοκιμές που είναι πάρα πολύ μακρόχρονες και καθυστερούν πάρα πολύ την κυκλοφορία των φαρμάκων. Μια σειρά ουσιών που έχουν αφαιρεθεί, όπως για παράδειγμα η περίπτωση του Γκλίβεκ για την γλυκαιμία. Μετά, κατάσταση των ζώων και φαρμακολογικού τύπου επεισόδια εξαιτία της έλλειψης γνώσης του μηχανισμού λειτουργίας των φαρμάκων. Αποτυχία των φαρμάκων που οδηγεί σε αύξηση των δημοσίων δαπανών και αύξηση του δείκτη θνησιμότητας. Υπάρχουν αρρώστιες οι οποίες πραγματικά θερίζουν. Οι στόχοι της ζωοτομίας δεν έχουν επιτευχθεί. Και μάλιστα δεν τίθεται καν το θέμα της ε, θεραπείας τίθεται μόνο το θέμα της επιμήκυνσης της ζωής. Μετά από έναν αιώνα ε, πειραμάτων με ζώα, η ζημιά που έχουν προκαλέσει είναι τεράστια και βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολύ περίπλοκης κατάστασης, υγειονομικής κατάστασης. Ε, πολλοί γιατροί και επαγγελματίες έχουν Υποβάλλει καταγγελίες και δεν εφαρμόζεται ο μηχανισμός της, η αρχή της πρόληψης. Θα έπρεπε η ζωοτομία τουλάχιστον να ανασταλεί. Πέραν αυτού υπάρχουν τοξικές ουσίες σε υψηλή συγκέντρωση, μια μόλυνση που σχετίζεται με τις ασθένειες. Εκτιθέμεθα σε μια σειρά ουσιών των οποίων το αποτέλεσμα δεν γνωρίζουμε. Ο κανονισμός REACH επιτρέπει να χρησιμοποιούμε τα στοιχεία των, που προκύπτουν από ε, επιράματα σε ζώα αλλά και πάλι δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε τις ζημιές όπως για παράδειγμα με τον άσβεστο. Χρειάζεται να βρούμε εναλλακτικέ λύσεις. Η ζωοτομία είναι άχρηστη, η ζωοτομία είναι άχρηστη και μεθοδολογικό σφάλμα. Η χρήση της έχει καταστροφικές συνέπειες. Θέλω να σας δείξω μερικές εικόνες για να καταλάβετε γιατί μιλάμε. Δεν, δεν μπορούμε να μιλάμε για ευζοία όταν χρησιμοποιούμε αυτή την τεχνική. Η ζωοτομία προκαλεί πόνο και ασθένειες. Σύμφωνα με τις συνθήκες μας, σύμφωνα με τους κανόνες μας, κάτι τέτοιο δεν θα ήταν δυνατό αν δεν αποδειχθεί ότι είναι απολύτως απαραίτητη. Μία από τις αιτιολογίες όμως είναι ε, ότι η ζωοτομία γίνεται μεταξύ άλλων για να προβλεφθούν αντιδράσεις των ανθρώπων. Όμως, παρόλα τα ε, πειράματα στα ζώα, τελικά δεν καταλήγουμε να γνωρίζουμε ποιος είναι ο κίνδυνος για τους ανθρώπους. Επίσης δεν ξέρουμε τι γίνεται με το θυλασμό. οι μηχανισμοί εξακολουθούν να είναι άγνωστοι, ε, παρόλο ότι ε, τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για πολλά χρόνια. Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η διαφορά μεταξύ των ειδών, ε, η, ο πολυπαραγοντισμός των ασθενειών δεν είναι απλές καταστάσεις. Δεν μπορώ να σας δείξω τα εξοικολογικά στοιχεία βέβαια, αλλά οι απαντήσεις για τους ανθρώπους είναι άγνωστες. Άρα ο λόγος στην κυρία Τζούλια Μπέιντς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη. Ο κανονισμός ΡΙΤΣΕ ε, περιλαμβάνει την αξιολόγηση και βασικές ε, προϋποθέσεις που θα μειώνουν τις επιπτώσεις στα ζώα. Οι δοκιμές στα ζώα πρέπει να γίνονται μόνο ως τελευταία λύση και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται τέτοιες μέθοδοι όποτε είναι δυνατόν. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται μια αξιολόγηση του κίνδυνου. Παρ' όλα αυτά όμως η ΕΚΑ αναφέρει ότι πάνω από ένα εκατομμύρια ζώα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για δοκιμές σύμφωνα με το ΡΙΤΣ και περισσότερα περιμένουμε να χρησιμοποιηθούν στα επόμενα χρόνια και το ανησυχητικό είναι πολλές από τις δοκιμές ε, θα μπορούσαν να αποφευχθούν. Επίσης, ε, υπήρξε αναφορά προς τα κράτη-μέλη ότι τα ζώα συνεχίζουν ε, να χρησιμοποιούνται στις δοκιμές χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη έγκριση ή έχουν χρησιμοποιηθεί σε δοκιμές δέρματος και ματιών χωρίς να έχουν υπάρξει εγκεκριμένες μέθοδοι ε, να έχουν χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένοι μέθοδοι που δεν περιλαμβάνουν ζώα. Έτσι λοιπόν, 100.000 πολίτες υπέγραψαν μια ανοιχτή επιστολή που ζητά από την Επιτροπή και την ΕΚΑ να σταματήσει αυτή την αναθεώρηση του ΡΙΤΣ, ε, να πάρει μάλλον, ε, να μετράξει αυτή την ευκαιρία για να χρησιμοποιήσει την αναθεώρηση του ΡΙΤΣ για να αλλάξει η κατάσταση με τα ζώα. Έχει ήδη ε, δημοσιευτεί η έκθεση REACH ε, ε, και έχουν βρεθεί ευκαιρίες που θα μπορέσουν να μας οδηγήσουν σε πιο συγκεκριμένη ομαδοποίηση των προσεγγίσεων και στο να εξετάσουμε τα στοιχεία ώστε να αποφύγουμε τα ζώα. Επενδύσεις σε νέες προσεγγίσεις και έγκριση νέων μεθόδων in vitro. Ε, περισσότερα λοιπόν μπορούν να γίνουν για να επιταχυνθεί η ρυθμιστική αποδοχή αυτών των μεθόδων. Όμως, από τις 16 δράσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση για την αναθεώρηση του REACH ε, για να βελτιωθεί ε, η κανονιστική ορθότητα του ΡΙΤΣ, ε, καμία από αυτές δεν μιλάει για την ε, ελαχιστοποίηση των δοκιμών στα ζώα. Μάλιστα υπάρχει ένα πολύ επικίνδυνο προηγούμενο, γιατί αναφέρεται ότι παρόλο που έχει βελτιωθεί η ανάπτυξη μεθόδων που δεν περιλαμβάνουν ζώα, αυτό τελικά ε, μάλλον βλάπτει την παροχή πληροφοριών περί του κινδύνου. Φαίνεται λοιπόν ότι ε, μόνο με τα ζώα ε, έχουμε ανώτερα στοιχεία σε, ε, έτσι θεωρεί η αναθεώρηση του ΦΙΤ, όμως αυτό δεν ισχύει. Επίσης, η ερμηνεία του Ρίτσα από την Κομισιόν στην ουσία παραφιάζει και τον κανονισμό για τα καλλιτικά. Το 2014 η ΕΚΟ και η Κομισιόν δημοσίευσαν κοινή δήλωση όπου λέγεται ότι μπορούν να γίνουν υπό συγκεκριμένε συνθήκες δοκιμές σε ζώα για καλλιντικά για τους σκοπούς του ΡΙΤΣ. Επίσης υπάρχουν ε, κάποιες ε, τέτοιες ε, προσεγγίσεις που είναι κατά της απαγόρευσης σύμφωνα με το ΡΙΤΣ. Πρέπει να... Και, και αυτός είναι ο λόγος που έγινε η καταγγελία στον Ομπούτσμαν από την ΠΙΤΑ. Υπάρχει ένα έγγραφο εργασίας ε, στο οποίο η Κομισιόν ε, θεωρεί ότι η κοινή ε, δήλωση αυτή δεν αντιτίθεται στις απογορεύσεις δοκιμών. Αυτό είναι κατηγορηματικά ανακριβές η διαμεσολαβήτρια δεν ε, συμφώνησε με την Κομισιόν, μάλιστα κράτησε επιφύλαξη και είπε ότι η κοινή δήλωση δεν είναι νομικά δεσμευτική και το γεγονός ότι η Κομισιόν και η, ΕΚΟ, η ΕΚΑ ε, στέλνουν τέτοιες οδηγίες, αυτό δεν προ, προϋποθέτει ότι είναι σωστή η καθοδήγηση αυτή. Θεωρώ λοιπόν ότι η αναθεώρηση του Ρίτζ είναι μια χαμένη ευκαιρία. Θα ήθελα λοιπόν να μην χαθούν τρεις χρυσές ευκαιρίες. Ε, σας ζητώ να συστήσετε στην Κομισιόν να ε, ε, συνεργαστεί με την Επιτροπή Περιβάλλοντος για να ενισχυθούν οι μηχανισμοί που έχουν σχεδιαστεί για να ελαχιστοποιήσουν τις δοκιμές στα ζώα και να συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη για να εφαρμοστούν σημαντικές ποινές για δοκιμές που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί σε ζώα. Δεύτερον, Καθώς ε, τα παρατήματα του ΡΙΤΣ ε, θα αναθεωρηθούν, είναι σημαντικό η Κομισιόν να αναπτύξει μια, ένα στρατηγικό σχέδιο για σιγά σιγά να σταματήσουν οι ρυθμιστικές δοκιμές στα ζώα και να γίνουν πιο εξελιγμένες ε, δοκιμές οι οποίες σχετίζονται περισσότερο με την ανθρώπινη επιστήμη. Τέλος, ε, είναι σημαντικό η Κομισιόν και η ΕΚΑ να επανεξετάσουν την αλληλεπίδραση μεταξύ του ΡΙΤΣ και των κανονισμών για τα καλλιντικά και να ε, σταματήσουν οι λανθασμένες ερμηνείες αυτών των δύο κανονισμών. Σημαντικό λοιπόν είναι να προωθήσουμε την επιστημονική και ανατομία, να ενισχύσουμε την ανθρώπινη υγεία και να βελτιώσουμε την ε, ευζοή των ζώων. Απλώς χρειάζεται να έχουμε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονται με τρόπο καινοτόμο. Τώρα ο λόγος στην Κάτριν Σούτεκ, εκ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τις επεξηγήσεις σας σχετικά με τις αναφορές σας. Από την πλευρά της Επιτροπής θα ήθελα να ενισχύσω την οπτική μας γωνία, την οποία έχουμε μοιραστεί μαζί σας και γραπτός, ότι όντως η Επιτροπή στηρίζει απόλυτα την πρόοδο σε ένα καινούριο επιστημονικό μοντέλο, μακριά από πειράματα σε ζώα, όπου αυτό είναι δυνατό και όπου υπάρχει εναλλακτική μεθοδολογία, η οποία έχει αναπτυχθεί επιτυχώς και μπορεί να αντιμετωπίσει τα επιστημονικά ζητήματα. Σε πολλές περιοχές έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή μέσω της Γενικής Διεύθυνσης RTD, της ΕΝΒ και της ΣΑΝΤΕ στηρίζουν την ανάπτυξη νέων μεθόδων με σοβαρές χρηματοδοτή, χρηματοδοτήσεις ερευνητικά προγράμματα σε ό,τι φορά τον ορίζοντα 2020 και για το 2019 υπήρξαν νέες εκκλήσεις για την επαλήθευση μεθοδολογιών σε ό,τι αφορά νέες ε, επιστημονικές μεθόδους που θα καταλήξουν, ε, ελπίζουμε, στην χρηματοδότηση 6 με 10 νέων επιστημονικών προγραμμάτων. Επομένως, η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων συνεχίζεται με τεράστια ταχύτητα. Οφείλω να ομολογήσω ότι οι παρουσιάσεις των ατόμων που έκαναν τις αναφορές φαίνονται κάπως μονομερείς γιατί κατά κάποιο τρόπο δείχνουν ότι εναλλακτικέ μέθοδοι υπάρχουν για όλους τους τομείς ασφαλών δοκιμών. Δυστυχώς πράγμα το οποίο θλίβει ιδιαίτερα την Κομισιόν, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα σε πάμπολους τομείς και γι' αυτό το λόγο σε πολλές περιπτώσεις χρησιμοποιούμε μια ελεγχόμενη, χρησιμοποιούμε ελεγχόμενα πειράματα σε ζώα όπου αυτό είναι υποχρεωτικό. Στους τομείς αυτούς επαναλαμβάνω όπου δεν υπάρχουν εναλλακτικέ μέθοδοι. Σε ό,τι αφορά την Οδηγία 2010-63, ρυθμίζει την χρήση των πειραμάτων σε ζώα με πολύ αυστηρό τρόπο. Η Επιτροπή ετοιμάζεται να δημοσιεύσει δύο εκθέσεις υπό το φως της οδηγίας αυτής το Νοέμβριο αυτής της χρονιάς, η μία αφορά στην εφαρμογή της οδηγίας στα διάφορα κρατημέλη και η αναφορά θα δίνει πληροφορίες για τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιούνται για επιστημονικούς λόγους. Επομένως έχετε ε, το νου σας για τις εκθέσεις αυτές που πιστεύω ότι θα δείξουν τις ε, θετικές εξελίξεις και ε, επίσης θα υποδείξουν και πού μπορούμε να κάνουμε ακόμη πρόοδο σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Οι αναφέροντες αναφέρθηκαν επίσης στην τελευταία έκθεση της ΕΚΑ ό,τι αφορά την αξιοπιστία των πειραμάτων σε ζώα και το περιεχόμενο των πειραμάτων της Ριτς και πάλι έχω την εντύπωση ότι η παρουσίαση των πορισμάτων της ΕΚΑ ήταν κατά κάποιο τρόπο μονομερής γιατί η έκθεση της ΕΚΑ έδειξε με λεπτομέρειες και πολύ συγκεκριμένα σε πόσες περιπτώσεις οι εταιρείε απέφυγαν την χρήση ζώων προσπαθώντας να χρησιμοποιήσουν άλλου τύπου εργαλεία μετρήσεων και in vitro τεχνολογίες αλλά και άλλες εναλλακτικές τεχνολογίες. Επομένως, για το 2018 το συμπέρασμα ήταν ότι τέλος μέχρι σήμερα η REACH έχει χρησιμοποιήσει πολύ πολύ λιγότερα ζώα από ό,τι είχε προβλεφθεί όταν ε, πρώτο εισήχθη η οδηγία REACH. Η Επιτροπή εξακολουθεί να δεσμεύεται στην υποχρέωσή της να ανανεώνει τα παρατήματα τα επιστημονικά, όταν υπάρξουν επιστημονικές μέθοδοι και είναι διαθέσιμε. Αυτή τη στιγμή διεξάγουμε μία έρευνα σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ε, σε ό,τι αφορά την, τις εναλλακτικής μεθόδους αλλά και τις δοκιμές για την αναπαραγωγική τοξικότητα. Και για αυτές τις εκθέσεις παρακαλώ έχετε το νου σας στο μέλλον. Έχοντας όλα αυτά κατά νου, λοιπόν, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι οι διατάξεις του κανονισμού REACH είναι πάρα πολύ σύγχρονες ό,τι αφορά τη χημική νομοθεσία με στόχο να ελαχιστοποιήσουν όσο το δυνατόν γίνεται τη χρήση ζώων και η Επιτροπή εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες προς την κατεύθυνση αυτή με όλες τις δυνάμεις της, μέσω των γενικών διευθύνσεων, των αρμόδιων γενικών διευθύνσεων, αλλά και μέσω της κοινή έρευνας και της ομάδας ΕΚΠΑΜ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε. Ο λόγος στην κυρία Εύη για τις πολιτικές ομάδες πλέον. Κύριε Εύη, ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες. Για μία ακόμα φορά έχουμε ένα θέμα πολύ σημαντικό. Έχουμε χάσει χρόνο, έχουμε μείνει πίσω. και η αρχή της ε, πρόληψης, η αρχή της προφύλαξης μάλλον, θα έπρεπε να, είναι, να θεωρείται δεδομένη. Υπάρχει στην, εθνική, στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, αλλά δεν την χάνει σεβασμού. Η νομοθεσία λέει ότι σταδιακά θα καταργηθεί η χρήση των ζώων στο εργαστήριο. Πότε θα γίνει όμως τελικά. Αυτό το ακούμε εδώ και χρόνια. Δεν έχουμε ακόμα όμως τα απαραίτητα εργαλεία προκειμένου να εγκαταλείψουμε αυτή την βάρβαρη και απάνθρωπη πράξη. Τα νούμερα είναι εκεί, τα ξέρουμε όλοι. Το 90% των φαρμάκων δεν ξεπερνούν το στάδιο των κλινικών δοκιμών, δεν διατίθενται λοιπόν στο, στο εμπόριο, διότι αποδεικνύονται αναποτελεσματικά. αλλά με τον τόσο χρόνο που χάνουμε για να τα δοκιμάσουμε, καθυστερούμε με φάρμακο που πραγματικά είναι χρήσιμα και σώζουν ζωές. Για το Alzheimer, για παράδειγμα, έχουμε επενδύσει τρομακτικά ποσά με πολύ φτωχά αποτελέσματα. Γιατί, γιατί εξακολουθούμε να πειραματιζόμαστε με ζώα, ενώ υπάρχουν πλέον τεχνολογίες που θα μας βοηθήσουν να πάμε πολύ πιο γρήγορα με άλλο τρόπο. Οπότε έχει φτιάξει, φτάσει πια η ώρα να κάνουμε αυτό το άλμα. Να εγκαταλείψουμε οριστικά την μεθοδολογία αυτή που είναι άχρηστη και βασανιστική. Αυτό γίνεται και στον υπόλοιπο κόσμο. Η περιβαλλοντική υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε χτες ότι το, από το 2025 και μετά η χρήση των θηλαστικών σε πειράματα θα μειωθεί πάρα πολύ και θα καταρριφθεί από το 2035 και μετά. Αυτό κάνει και ο υπόλοιπο πλανήτη λοιπόν. Εμεί τι κάνουμε, περιμένουμε. Θα πρέπει να γίνονται περισσότεροι έλεγχοι. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε ζώα ενώ υπάρχουν εναλλακτικές μέθοδοι. που δεν χρησιμοποιούνται όμως για εξαιτία πολλών πολλών λόγων. Θέλω να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά, να συνεχίσουμε να μεριμνούμε για αυτό το ζήτημα. Και όλες οι πληροφορίες που μας δίνουν οι αναφέροντες πρέπει να αποσταλούν στην καινούρια Κομισιόν και στην καινούρια Πρόεδρό της. Ευχαριστώ ως Φλόρε. Ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τη Ρομπέρτα Φωνασάρη που σήμερα βρίσκεται εδώ μαζί μας γιατί αυτό το θέμα που έθιξε πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ήθελα να συμφωνήσω με τη Σνάλφα να την ευχαριστήσω και για την δουλειά της ε, ως τον τομέα της προστασίας των ζώων. Πραγματικά η κατάργηση της ζωοτομίας δεν είναι ένα θέμα καινούριο για την Κομισιόν. Αυτό ε, συνάδει και με αυτά που θέλουν οι πολίτες. Θέλουν περισσότερη προστασία των ζώων. Είχαμε τον ε, κανονισμό το 2010. Ήδη από το 2007 είχαμε μιλήσει για εναλλακτικά μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μείωση των δοκιμών σε ζώα, των δοκιμασιών σε ζώα. Στο μεταξύ, ε, παρατηρήθηκαν οι αρνητικές συνέπειες ε, στους ανθρώπους ε, και στο περιβάλλον. Πραγματικά είδαμε πόσο Φρικαλές είναι αυτές οι μέθοδοι για τα ζώα, οι επιστημονικές ε, μέθοδοι οι οποίες ε, θα προστατεύουν το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Ε, είναι ένα επιχείρημα διεθνές και εθνικό που πάντοτε πραγματικά ισχύει. Θα ζήταγα λοιπόν και θα έκανα έκκληση η Κομισιόν χωρίς άλλη καθυστέρηση να προχωρήσει σε αυτό σε διευθέτηση αυτού του θέματος. Η κυρία Άουκεν, θα μιλήσω δανέζικα. Θα κάνω δηλαδή μια εξαίρεση στον κανόνα μου, γιατί αυτό εδώ το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Ευχαριστώ την Επιτροπή, κατανοώ την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω και τους αναφέροντες. Είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να εξετάζουμε αυτό το θέμα. Πριν από μερικά χρόνια ήμουν μέλος ε, ενός ε, γραφείου για τις δοκιμές στα ζώα. Εκπροσωπούσα τα ζώα συγκεκριμένα. Τελικά είδα ότι τα ζώα που χρησιμοποιούνται στις ε, ιατρικές δοκιμασίες προστατεύονται πολύ καλύτερα από ότι τα βιομηχανικά ζώα. Δηλαδή αυτά που γίνονται στα βιομηχανικά ζώα δεν γίνονται στα ζώα εργαστηρίου. Υπάρχουν λοιπόν κάποιες απαιτήσει ε, οι οποίες ε, έχουν μετατραπεί σε νομοθεσία σε πολλές χώρες ε, και τελικά γίνονται σεβαστές. Και τελικά έχει γίνει πολύ δαπανηρό να χρησιμοποιήσεις ζώα για το εργαστήριό σου. Έχει ενεργό ενδιαφέρον λοιπόν η βιομηχανία να απαλλαγεί από τις δοκιμές στα ζώα. Έχουν ξεκάθαρο συμφέρον να αποφύγουν τις δοκιμές στα ζώα, όχι χάρη των ζώων, αλλά χάρη της δικής τους ε, τσέπης. Στα Ηνωμένε Πολιτείε επίσης έχουν μια νομοθεσία που αφορά στην ευθύνη των προϊόντων. Ε, δεν το έχουμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν μια εταιρεία δηλαδή παράγει κάτι που βλάπτει τους ανθρώπους θα έρθει ένα ολόκληρο jumbo jet με δικηγόρους και θα προσγειωθεί στην αυλή σου και θα προσπαθήσει να σε ε, ε, διώξει. Ε, έτσι λοιπόν, ακόμα και το να χρησιμοποιήσεις μια σύριγγα στο ζώο σημαίνει ότι προκαλείς πόνο στο ζώο. Δεν επιτρέπεται. για την αρθρίτιδα για παράδειγμα. Δεν πρέπει να προκαλέσεις πόνο στα ζώα και γι' αυτό χρησιμοποιούν περισσότερα ζώα. Αυτό τελικά ε, δεν ξέρω κατά πόσο σημαίνει ότι είναι χειρότερο για τα ζώα, ε, μάλλον έχουν καλύτερη μεταχείριση. Το θέμα είναι ε, πώς θα φυλάσσουν βέβαια μεταξύ ε, ή πριν ή μετά από αυτές τις δοκιμασίες είναι σε στάβλους, πού τα, ε, τα φυλούν τα ζώα. Γενικά από ό,τι βλέπω όμως, ε, επειδή έχω παρακολουθήσει αυτό το θέμα για χρόνια, η βιομηχανία θεωρεί ότι είναι πολύ δαπανηρή αυτή την χρήση των ζώων. Ε, παρόλα αυτά δεν μπορεί να την αποφύγει τελείως, ε, ε, γιατί με τα in vitro πειράματα δεν φτάνει. Πρέπει να υπάρχουν και δοκιμές σε ζωντανούς οργανισμούς. Βέβαια, όπως είπα, τα ζώα είναι πάρα πολύ δαπανηρή μέθοδος ε, για αυτούς. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί σε αυτά που λέμε. Δεν ελπίζω φυσικά ότι έχουν επιδεινωθεί τα πράγματα από τότε που εγώ έχω να ασχοληθώ. Με αυτά που λένε οι Ιταλοί συνάδελφοι φαίνεται σαν να πήγαμε προς τα πίσω. Έχω εργαστεί από αυτού του θέματος και δεν νομίζω ότι πλέον ε, ασχολούμαστε με τα ζώα με χειρότερο τρόπο, είναι πολύ σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, να υποστηρίξουμε αυτό το υψηλό επίπεδο προστασίας για τα ζώα του εργαστηρίου και κάποια από αυτά τα στοιχεία να τα περάσουμε και στα ζώα ε, της κτηνοτροφίας, της βιομηχανίας. Ε, γιατί αν είχαμε τα ίδια επίπεδα, τότε η Ευρωπαϊκή Στάβλη για, τα χείρο, για τους χείρους και τα βοηδή θα ήταν πολύ διαφορετική από αυτό που έχουμε σήμερα. Ε, δεν επιτρέπεται τα ζώα του εργαστηρίου να τα αντιμετωπίζεις όπως ε, αντιμετωπίζονται ε, τα ζώα της βιομηχανίας. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Όλα τα ίδια λένε, παιδιά. Ευχαριστώ ο τον κύριο Μπούχμαν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εδώ ευχαριστώ τους αναφέροντες ε, και ε, που υποστηρίζουν αυτή την αναφορά. Το 2011 είχαμε 11.000 ε, ζώα που χρησιμοποιήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για δοκιμές. Αυτά λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτό σημαίνει ότι τα βασάνισαν και τα ε, εκμεταλλεύτηκαν, τα μεταχειρίστηκαν ε, βάναυσα και τα σκότωσαν για επιστημονικούς λόγους. Είχαμε ε, και σκύλους και γάτες, ποντίκια, κάποιους πυθίκους, όλα αυτά μόνο και μόνο στη Γερμανία ήταν σε μεγάλους αριθμούς. Όλα αυτά με βάση και είχαν ως αιτιολογία την προστασία των ανθρώπων. Δυστυχώς τα ζώα δεν έχουν φωνή στην κοινωνία και γι' αυτό δεν μπορούν να προστατευτούν. Ε, δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε όταν μιλάμε για την ασφάλεια των ανθρώπων λιγότερο από το 1% των μελετών που γίνονται στα ζώα τελικά έχουν κάποια αξία για τους ανθρώπους. Ε, ε, πολλές φορές γίνονται δύο και τρεις φορές οι δοκιμές, ε, γιατί δεν υπάρχει κάποια βάση δεδομένων και δεν ανταλλάσσονται τα στοιχεία. Έτσι λοιπόν χωρίς νόημα για την ίδια ουσία βασανίζονται πολλές φορές τα ζώα. Ούτε ηθικά λοιπόν αυτό ε, μπορεί κανείς ε, να το υπερασπιστεί. Εδώ είμαστε για να υπερασπιστούμε την ευμερία των ζώων. Υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικέ ε, μέθοδοι, μικρά όργανα με τη μορφή chip, organ on a chip. Αυτά μπορούν να αναγνωρίσουν καλύτερα τις επιδράσεις των φαρμάκων και να έχουμε και λιγότερες δοκιμασίες ζώα. Επίσης μπορούν να γίνουν προσωμιώσεις σε υπολογιστές. Αυτές οι εναλλακτικέ ε, ε, μέθοδοι λοιπόν πρέπει να υποστηριχθούν οικονομικά για να μην υπάρχει πλέον η ανάγκη να χρησιμοποιούνται ζώα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να αφήσουμε ανοιχτή και να προωθήσουμε την αναφορά στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος ε, Παρανικούμφεν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους αναφέροντες. Όπως είπαν και οι συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να τονίσω ότι όπως είπε και η Κομισιόν, υπάρχουν πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια που ισχύουν. Ε, πολλές φορές ε, υπάρχουν κάποιες ε, τέτοιες δοκιμασίες οι οποίες οδηγούν σε μεγάλες ιατρικές ε, καινοτομίες. Υπάρχουν εναλλακτικέ, ε, αλλά είναι δύσκολο κανείς να τις βρει. Αυτές οι αναφορές δείχνουν ότι υπάρχουν πολύ καλές απαντήσεις από την Κομισιόν για το πώς μπορεί να προχωρήσει το θέμα στην Κομισιόν. Υπάρχουν συνεχώς βελτιώσεις, υπάρχει καθοδήγηση ως προς το τι πρέπει να γίνει. Θεωρώ λοιπόν ότι επειδή πρέπει να έχουμε όσο λιγότερες αναφορές γίνεται και φόρτο λόγω αυτών και εφόσον η Κομισιόν έχει επεξεργαστεί πολύ καλά το θέμα, προτείνω να κλείσει αυτή η αναφορά. Ευχαριστώ Υπάρχουν πολλά ηθικά ζητήματα σχετικά με το, τα πειράματα στα ζώα και η τάση είναι και πρέπει να είναι μια τάση μείωσης της χρήσης των ζώων και προς πειράματα τα θα είναι πιο γρήγορα, πιο οικονομικά και πιο αποτελεσματικά. Όμως θα πρέπει να είμαστε και ρεαλιστικοί. Εξακολουθεί να υφίσταται ανάγκη χρήση ζώων στα πειράματα σε πολύ, πολύ συγκεκριμένους τομείς, πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις με πολύ περιοριστικό τρόπο. Η αναφορά της ε, ΠΕΤΑ δεν έλαβε μια πλήρη απάντηση από τους ομιλητές. Όταν υιοθετήσαμε το REACH το 2006 ήταν ε, πολύ ε, πρωτότυπο νομοθέτημα και επαναστατικό. Θα πρέπει να είμαστε περήφανοι. Με το ΡΙΤΣ ε, καθορίζεται ότι η χρήση των ζώων για πειράματα είναι το τελευταίο καταφύγιο και είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρακολουθούν το κατά πόσον αυτό υλοποιείται και οι μη κυβερνητικέ οργανώσει και ιδιώτες, άτομα. Χρειάζεται να εξασφαλίζουμε την ασφάλεια και την υγεία όχι μόνο στη ζωή μας και στην εργασία, στον χώρο εργασίας, αλλά και στη ζωή των ζώων. Είναι σημαντικό εμείς ως ευρωβουλευτές να εξασφαλίζουμε ότι ο κανονισμός REACH εφαρμόζεται σωστά. Η κατοπινή απαγόρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χρήση ζώων σε πειράματα για καλλιντικά ήταν πολύ συνεπής ε, με τη λογική του Ρίτς, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίζουμε, επαναλαμβάνω, ότι πράγματι εφαρμόζονται αυτές οι, αυτά τα νομοθετικά κείμενα. Πιστεύω ότι θα πρέπει να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά της Julian Baines και να είμαστε σε εγρήγορση Αυτή είναι η διαφορά του δικού μας ρόλου σήμερα σε σχέση με το ρόλο των ευρωβουλευτών σε προηγούμενες θητείες. Εμείς πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση να παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις. Και θα πρέπει να είμαστε πολύ δυναμικοί και στον υπόλοιπο κόσμο έτσι ώστε να καταλήξουμε σε μια σε εισαγωγικά εξοειδαφική εφαρμογή του κανονισμού REACH. Να οθήσουμε και άλλες χώρες για αντίστοιχες απαγορεύσεις ε, η Νέα Ζηλανδία, το Ισραήλ, η Ινδία και άλλες χώρες είναι χώρες που πραγματικά θα μπορούσαν να μπουν σε αυτό το δρόμο. Και θα έπρεπε να το προσπαθήσουμε. Εκεί, επαναλαμβάνω, σε αυτό το πράγμα διαφέρει ο ρόλος μας σήμερα από το ρόλο των ευρωβουλευτών σε προηγούμενες θετίες. και θα πρέπει στο μέτρο που μπορούμε να χρησιμοποιούμε μεθόδους ε, ανάλυσης των φαρμάκων που δεν χρησιμοποιούν ζώα. Ευχαριστώ πολύ. Κλείνοντας, θα δώσουμε ένα ενάμιση λεπτό σε κάθε μία από τις αναφέρουσες. Καταρχήν ο λόγος στην κυρία Φορνασάρη. Ευχαριστώ πολύ για όλες τις νόμες που εκφράστηκαν. Το πρόβλημα είναι το εξής. Αν η χρήση των ζώων δεν είναι απολύτως απαραίτητη, κάνουμε ένα μεθοδολογικό λάθος. Υπάρχουν χιλιάδες γιατροί τις τελευταίες δεκαετίες που έχουν καταγγείλει την ζωοτομία ως το βασικό πρόβλημα για την ευζοία των ζώων. Ο Κλοντ Μπράιντ που ήταν για πολλά χρόνια ε, διευθυντής του Τμήματος Έρευνας του CNR στη Γαλλία έχει πει ότι μεταξύ όλων αυτών που έχουν, μετά από όλα όσα έχουν ακουστεί είναι απίστευτο το ότι δεν έχει δοθεί τέλος σε αυτό το σύστημα. Η, ο ρόλος της ζωοτομίας είναι καταστροφικός. Κάποια στιγμή θα εγκαταλειφθεί όπως και η η δουλεία όπως και το apartheid. Η απόλυτη και οριστική κατάργηση της ε, ζωοτομίας είναι απολύτως απαραίτητη και πρέπει να γίνει αμέσως, εδώ και τώρα. Και θα πρέπει να εγκαταλειφθούν τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν ζώα στα πειράματά τους. Το 1910 ε, από το 1910 οι γιατροί και οι κτηνίατροι ζητούν κατάργηση αυτής της μεθόδου. Έχει περάσει πάνω από ένα αιώνα και ακόμα δεν έχει συμβεί. Έχουμε 83 εκατομμύρια ημέρες νοσοκομιακής περίθαλψης εξαιτίας της ανικανότητάς μας να σχεδιάσουμε τα φάρμακα σωστά και αποτελεσματικά. Και αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούμε ζώα στα πειράματά μας και όχι εναλλακτικές μεθόδους. Είναι τρομακτικός αυτός ο αριθμός και επηρεάζει πάρα πολύ προφανώς βαθιά και την οικονομία μας. Η χρήση των ζώων μας δίνει μια ψευδεπίγραφη ασφάλεια. Στην πραγματικότητα το κόστος είναι τεράστιο. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο στην άλλη αναφέρουσα. Ευχαριστώ πολύ. Με δεδομένο ότι εξακολουθούμε να βλέπουμε που και που τη χρήση μη απαραίτητων πειραμάτων σε ζώα και με δεδομένο ότι η ίδια η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι κάποια πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν στην εφαρμογή και στην ανάπτυξη μεθόδων που δεν αφορούν ζώα. Α, και με δεδομένο ότι αρκετές εταιρείες κοσμημάτων εξακολουθούν να κάνουν πειράματα σε ζώα, είναι σαφές ότι ο κανονισμός REACH δεν λειτουργεί έτσι όπως θα έπρεπε και είναι ανάγκη να αλλάξουμε το μοντέλο μας πέρα από τα πειράματα στα ζώα. Χρειαζόμαστε ένα στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα εξασφαλίσει τη βελτίωση της καλής μεταχείρισης των ζώων. Επομένως, ας θέσουμε μία προθεσμία και ας δουλέψουμε πάνω σε αυτό και ας μη χρησιμοποιούμε τον κανονισμό REACH για να επιτρέπουμε στην βιομηχανία κοσμημάτων να παραβιάζει διαρκώς τους όρους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους ανα... τις αναφέρουσες που ήρθαν εδώ έχοντας ακούσει την Κομισιόν και τις κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης και τις αναφερόμενες. Θα διατηρήσουμε ανοιχτή, ανοιχτές και τις τρεις αναφορές και θα παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις, τις βελτιώσεις που θα γίνονται από την Κομισιόν και περιμένω από την Κομισιόν να μας ενημερώσει ε, στο μέλλον για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται αυτέ τι αναφορέ. Περνάμε στο επόμενο σημείο τη ημερησία διάταξη, το 14, αναφορά 0439 του 12, του Αντρέα Ρουτιλιάνο, Ιταλική Ιθαγένεια, εξ ονόματο τη Επιτροπή κατά τη Θανάτωση Πτηνών. Σχετικά με τη μία εφαρμογή από την Κυπριακή Δημοκρατία τη Οδηγία 2009-147 σχετικά με την προστασία των άγριων πτηνών. Ο αναφέρον δεν είναι παρόν, αλλά ε, μας παρακολουθεί μέσω του ίντερνετ και μας έστειλε επικαιροποιημένα έγγραφα. Θα δώσω καταρχήν το λόγο στην Κομισιόν, στον κύριο Πολ Σπέιθ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή συμφωνεί ότι η παράνομη παγίδευση πουλιών εξακολουθεί να, να παραμένει ζήτημα ανησυχία στην Κύπρο τόσο εξαιτίας του μεγάλου δικτύπου που έχει στον πληθυσμό των πουλιών, αλλά και λόγω των κινήτρων, η κατανάλωση των πουλιών αυτών σε εστιατόρια, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχει εξαλειφθεί. Θα ήθελα να ενημερώσω την Επιτροπή σας ότι η Κυπριακή νομοθεσία εξακολουθεί να συμμορφούνται με τον Ευρωπαϊκό νόμο. Δεν υπάρχει ζήτημα επομένως συμμόρφωσης. Επίσης, είχαμε κάποια θετικά βήματα από τις Κυπριακές Αρχές που περιλαμβάνουν κυρίως την ανέβρεση επιτόπου των παγίδων, κάτι το οποίο είχε θετικές επιπτώσεις στις περιόδους παγίδευσης, στις τελευταίες περιόδους παγίδευσης. Αν ε, ελέγξουμε τις τελευταίες αναφορές βλέπουμε μια κάπως πολύπλοκη εικόνα. Σε κάποιες περιοχές έχει μειωθεί, κάποιου είδους μέθοδοι παγιδεύσεως έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχει και μια μικρή άνοδο σε άλλους τομείς. Βλέπουμε ότι η επιβολή είχε αποτελέσματα αποτελέσματα απονθάρρυνσης. Έναν συμπεράσματος λοιπόν η Επιτροπή σημειώνει ότι οι Κυπριακές Αρχές και οι προσπάθειες επιβολής του κανονισμού τον τελευταίο καιρό είναι σημαντικέ. Εξακολουθεί να ανησυχεί όμω για τα υψηλά νούμερα και θα εξακολουθούμε να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυ στην δράση των κυπριαρχών αρχών σε ό,τι αφορά την παράνομη παγίδευση πουλιών οι προσπάθειές μας είναι να δώσουμε προτεραιότητα σε δύο πράγματα επί της ουσίας. Πρώτα απ' όλα να αντιμετωπίσουμε την πηγή του προβλήματος αυτός, με άλλα λόγια δηλαδή να μειώσουμε την κατανάλωση οδικών πτηνών στα εστιατόρια. Εξετάζουμε και εναλλακτικού τρόπους. Ένα παράδειγμα ας πούμε είναι ότι διοργανώσαμε ένα σεμινάριο στην Κύπρο για Κύπριους δικαστές, ούτως ώστε να αυξήσουμε την γνώση τους πάνω στο ζήτημα αυτό. Προς το παρόν υπάρχει πολύ μικρή χρήση του, της κυπριακής νομοθεσίας είτε από μη κυβερνητικούς οργανισμούς είτε από τους πολίτες για να αναλάβουν τις σωστές δράσεις. Αυτά είναι λοιπόν τα συμπεράσματά μας. Εξακολουθούμε να παρακολουθούμε από κοντά επιτόπου την υπόθεση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Θέλει κανείς το λόγο εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Όχι. Έχοντας ακουστεί κομισιόν και έχοντας μελετήσει το φάκελο, διατηρούμε ανοιχτή και αυτή την αναφορά. Ωραία. Περνάμε στο σημείο 15 της ημερήσιας διάταξης ανταλλαγή απόψεων με την διευθύνουσα ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το Brexit. Τα μέλη της διευθύνουσας ομάδας είναι έξι. Ο κ. Φερχόφστατ, κ. Χούμπνερ, Σίλβια Περέιρα, Λάμπερς, Σιρδεουάν και ο κ. Σταγιάννη. Είναι εδώ τέσσερις από τους έξι. Οπότε θα ξεκινήσουμε δίνοντας τον λόγο καταρχήν στον κύριο Φερχόφστατ, αλλά πιο πριν θα ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους της μόνιμης αντιπροσωπείας του Ηνωμένου Βασιλείου που βρίσκονται επίσης εδώ ε, παρόντες. Ο λόγος του κύριο Φερχόφστατ. Ευχαριστώ που με καλέσατε μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της διευθύνουσα Ομάδας. Θα ήθελα να σας πω ότι η Διευθύνουσα Ομάδα θα συναντηθεί μία ακόμα φορά σήμερα για να εξετάσει τις ενδεχόμενες νέες προτάσεις για το backstop που υποτίθεται ότι θα λάβουμε σε ένα λεπτό, στις 4 η ώρα το απόγευμα. Εικάζεται. Δεν είναι η πρώτη φορά που η ΠΕΤΗ έχει λάβει αναφορές σχετικές με τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και τον Brexit. Και πέρσι είχε λάβει αναφορές για την ακρίβεια από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε την εργασία της Διεθνής Ομάδα για τον Brexit και μπορώ να σας πω ότι πολύ προσεκτικά τις έχουμε εξετάσει στο παρελθόν. Τα δικαιώματα των πολιτών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρώτη στην προτεραιότητα, το γνωρίζετε εσείς πολύ καλά και εξακολουθούν να είναι πρώτη προτεραιότητα και σήμερα όλα τα δυόμιση τελευταία χρόνια έχουμε συζητήσει επανειλημμένως με τον επικεφαλής διαπραγματευτή τον κύριο Μπαρνιέ το πώς είναι δυνατόν να χειριστούμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούνται και από τις δύο μεριές της μάχης. Γιατί συζητούμε για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά ταυτόχρονα και για τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών που ζουν, διαμένουν μόνιμα στην υπηρετική Ευρώπη. Μιλάμε για παραπάνω από 4 εκατομμύρια άτομα. Πάνω από 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και πάνω από 1 εκατομμύριο Βρετανοί ζουν στην υπηρετική Ευρώπη. Έχουμε, εξετάσει, έχουμε εξηγήσει στον κύριο Μπαρνιέ τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί τα περασμένα χρόνια στην Επιτροπή Πέτη, αλλά όχι μόνο στην Επιτροπή Πέτη, διότι έχουμε συναντηθεί και με την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και άλλες επιτροπές. Ορισμένοι από τους αδέρφους μπορεί να το, θυμά, να το θυμούνται. Ο κ. Μωράης σίγουρα το θυμάται. Ε, η Επιτροπή Πέτη ε, έχει διοργανώσει σε κοινέ συναντήσεις, συνεδριάσεις με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ προκειμένου να συζητηθεί το θέμα αυτό με παρουσία των ε, υπαλλήλων του, Ευρωπα... του Υπουργείου Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου. Η... Ε, οι Βρετανοί το ονομάζουν αυτό το πρόβλημα το καθεστώς ε, των ε, μονίμως διαμενόντων, το settlers status και όπως σας λέω το έχουμε συζητήσει επανειλημμένως ε, προκειμένου να βρούμε μια λύση. Αν μου επιτρέπετε θα ήθελα να σας παραθέσω τα διάφορα σενάρια στα οποία καταλήξαμε. Γιατί ε, αν υπογραφεί μια συμφωνία αποχώρησης, ε, έχουμε ένα σενάριο. Το πώς θα εφαρμόσει τα δικαιώματα αυτά, τα οποία θα έχουν κατοχυρωθεί μέσω της συμφωνίας αποχώρησης, ε, είναι άλλο θέμα και άλλο σενάριο. Μετά Θέλω να δούμε, πρέπει να δούμε τι έχουν κάνει τα κράτη-μέλη για τους Βρετανούς πολίτες ως τρίτο στοιχείο. Και το τελευταίο έχει σχέση με το τι θα γίνει αν η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου γίνει χωρίς συμφωνία. Κατά τη διαπραγμάτευση της συμφωνίας ε, αποχώρησης, Η διευθύνουσα ομάδα για το Brexit προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση των δικαιωμάτων τα οποία θα προβλεπόντουσαν στην Συμφωνία Αποχώρησης. Η δική μας θέση από την πρώτη μέρα ήταν ότι δεν θα έπρεπε να γίνει κανένας είδους αλλαγή τροποποίηση των δικαιωμάτων. Τα δικαιώματα τα οποία εφίστανται σήμερα θα πρέπει, θα έπρεπε να συνεχίσουν να εφίστανται και στην και μετά την συμφωνία αποχώρησης. Βέβαια, η Βρετανική κυβέρνηση είχε άλλη προσέγγιση. Ήθελε κάτι λιγότερο από μια απλή επέκταση, χρονική παράταση των δικαιωμάτων. Ε, οπότε έγινε προσπάθεια να γίνει βελτίωση της αρχικής πρότασης Ε, θέλαμε, χρειάστηκε να προσθέσουμε ρήτρε για την επανένωση των οικογενειών, εγκατάσταση παιδιών, κάτι που είναι προφανές για μα, αλλά είχε παραλυφθεί, είχε παραλυφθεί στην αρχή τη συζήτηση. Δεύτερον, συμπερίληψη όλων των ε, κοινωνικών επιδομάτων. Τρίτον, η συμφωνία αποχώρησης να έχει άμεση ισχύ να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιηθεί ε, ενώπιον των δικαστηρίων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τέταρτον, εξασφαλίσαμε τον ρόλο του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την εφαρμογή και την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών των πολιτών. Και πέμπτον, καθόρισαμε τις ε, λεπτομέρειες ε, έτσι ώστε μια ανεξάρτητη αρχή να μπορεί να δράσει εξ ονόματος των πολιτών. Προβλέπεται λοιπόν μια ανεξάρτητη αρχή πλέον στην Συμφωνία Αποχώρησης. Έγινε μια διπλή μάχη για το καθεστώς εγκατάστασης της Συμφωνίας ε, Αποχώρησης, ε, έτσι ώστε το καθεστώς αυτό ε, να μην κοστίζει ε, στους πολίτες που θα το ζητήσουν. Μετά, ε, η, η, η, η οριστική, η τελική ημερομηνία για τους πολίτες για τα δικαιώματά τους να είναι η ημερομηνία στο τέλος μεταβατικής περιπτώσης, ε, περίοδου δεν ξέρουμε πόσο μακρά θα είναι αυτή η μεταβατική περίοδος, αλλά αυτή θα είναι η καταληκτική ημερομηνία για τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών και των Βρετανών πολιτών από την άλλη μεριά. Και τέλος, ελευθερία κυκλοφορία κατά τη διάρκεια τη μεταβατική περίοδου. Οπότε κατά τη διάρκεια τη μεταβατικής περίοδου ε, δεν θα τροποποιηθεί καθόλου η ελευθερία κυκλοφορία που ήδη υφίσταται. Αυτέ είναι οι αλλαγέ τι οποίε καταφέραμε να εντάξουμε στην Συμφωνία Αποχώρησης. Η τελική συμφωνία δεν ήταν 100% ικανοποιητική βέβαια. Ε, δηλαδή δικαιώματα ψήφου και το δικαίωμα επιστροφής καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής των πολιτών δεν έγιναν δεκτά ως αιτήματα, αλλά το 85% τουλάχιστον των αιτημάτων μας έγιναν δεκτά ε, και μιλώ πλεπάντα για τα δικαιώματα των ατόμων. 85% δεν είναι και λίγο. Ποτέ δεν έχω καταφέρει 85% σε μια διαπραγμάτευση στη ζωή μου εγώ. Οπότε δεν θα έλεγα ότι είναι και σημείο αναφοράς. Να σας υπενθυμίσω ότι πολλά από αυτά που μόλις ανέφερα τα έχουν διεκδικήσει και μέσω αναφορών οι Ευρωπαίοι πολίτες. Όχι όλα. Για... Δεν τα καταφέραμε όλα. Σας ε, μίλησα για το δικαίωμα ψήφου σε τοπικές εκλογές. Από την άλλη μεριά δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Εμείς μόνο εκφράζουμε επιθυμίες. Τα δικαιώματα ψήφου στι τοπικέ εκλογέ έχουν σχέση με την εθνική νομοθεσία κάθε φορά. Αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να οθήσουμε, να πιέσουμε τα κράτη-μέλη ε, έτσι ώστε να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται και να συντονίσουν τις διεκδικήσεις τους, τη διαπραγματευτική τους τεχνική και τα συστήματά τους. Αυτά σε ό,τι αφορά την συμφωνία αποχώρησης. Η οποία <laughs> δεν είναι προς εφαρμογή αυτή τη στιγμή βέβαια, έτσι, διότι φύσταται μια μεγάλη ασάφεια για το κατά πόσον θα εφαρμοστεί αυτή, κάποια άλλη, καμία. Το δεύτερο θέμα έχει σχέση με το πώς θα εφαρμοστεί η συμφωνία αποχώρησης. Διότι άλλο είναι τα δικαιώματα τα οποία κατοχυρώνονται με συμφωνίες και άλλο το πώς αυτά θα υλοποιηθούν, θα εφαρμοστούν και θα ασκηθούν. Έγιναν πολλές συνεδριάσεις με το Υπουργείο Εσωτερικών το, για το μέσο των οποίων πιέσαμε το σύστημα είναι όσο πιο φιλικό προς το χρήστη γίνεται. Ε, να μπορεί να γίνει όλες οι οι διαδικασίε να μπορούν να γίνουν ψηφιακά, αλλά όχι μόνο ψηφιακά μέσω του ίντερνετ. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το ίντερνετ, αυτοί θα πρέπει να μπορούν να ε, ασκήσουν τα δικαιώματά τους με μη ηλεκτρονικό τρόπο, ιδιαίτερα για τις πιο ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού. Επίσης, ζητήσαμε μια πραγματικά ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης που θα παρακολουθεί πραγματικά το κατά πόσον εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες και με ποιο τρόπο. Βέβαια, οι Βρετανικές αρχές λένε ότι ήδη έχουν έναν επιθεωρητή που εργάζεται στο Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά εμείς ζητήσαμε ανεξάρτητη αρχή και πραγματικά ανεξάρτητη αρχή. Να μην εξαρτάται από το Υπουργείο Εσωτερικών. Ε, ακόμα και ο ίδιος ο επιθεωρητής, ε, επικεφαλής επιθεωρητής του Νομού Βασιλείου, στο 2, στις 2 Μαΐου 2019 στην έκθεσή του έγραψε ότι εξακολουθούν να υφίστανται ανησυχίες τεχνικής και επικοινωνιακής φύσης Οπότε δεν έχει ολοκληρωθεί αυτή η διαπραγμάτευση και εμείς το ίδιο πιστεύουμε. Ε, αυτό που είναι πραγματικά ενισχυτικό είναι ότι τελευταία βλέπουμε σχόλια ε, που δεν αναφέρονται απλώ στο καθεστώς της ε, κατάστασης αλλά μόνο για ανθρώπους οι οποίοι το δικαιούνται Δηλαδή όχι για όλους. Ακούμε τέτοιου είδους αναφορές. Ε, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάνω από δύο δεκαετίες στη Βρετανία και ε, αντί να πάρουν το οριστικό καθεστώς έχουν ένα, τους προσφέρθηκε ένα προσωρινό καθεστώς. Ε, κανονικά θα έπρεπε μετά από πέντε χρόνια να παίρνουν το οριστικό καθεστώς που δικαιούνται. έχουμε ακούμε και τέτοιου είδου καταγγελίες. Τώρα, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο προσωρινό και το μόνιμο καθεστώ. Ε, στο προσωρινό καθεστώ έχει λιγότερα δικαιώματα, λιγότερη ασφάλεια σε σχέση με το οριστικό καθεστώ. Παίρνουμε στα σοβαρά αυτές τις καταγγελίες. Κάναμε μάλιστα και μία πρόταση για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Εδώ και πολλούς μήνες είχαμε πει το εξή. Το σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών λειτουργεί ω εξή. Ο, ο, θα πρέπει να, κατα... να υποβάλει μια αίτηση, να αιτηθεί να λάβει το καθεστώς της ε, Εμείς, από την άλλη μεριά, προτείναμε στο Υπουργείο Εσωτερικών να καθιερώσει ένα σύστημα αυτόματης ε, εγγραφής. Δηλαδή, όποιο εγγραφεί να παίρνει αυτόματα το καθεστώς. Οπότε να αντιστραφεί το βάρος απόδειξης. Το Υπουργείο Εσωτερικών, σε αυτή την περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, θα έπρεπε να έχει συγκεκριμένα στοιχεία για να απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα. Δηλαδή να πει ξέρω εγώ ότι στην πραγματικότητα εσύ κύριε λες ψέματα δεν έχεις, ε, δεν είσαι μόνιμος κάτοικος της, του Ηνωμένου Βασιλείου για πάνω από πέντε χρόνια. Οπότε με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε μια αυτόματη οριζόντια 100% συμμετοχή ε, με αποκλεισμό μόνο όσων το Ηνωμένο Βασίλειο, οι υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου θεωρούσαν ή απεδείκνυαν ότι δεν αξίζουν το καθεστώς. Εξακολουθούμε και στο τελευταίο μας ψήφισμα νομίζω, την Ολομέλεια, να πιέζουμε το Ενώμενο Βασίλειο να κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση της αυτόματης της αυτοματοποιημένης χορήγησης του καθεστώτος ε, εγκατάστασης στους Και γι' αυτό δεν χρειάζεται αλλαγή της ε, συμφωνίας αποχώρησης, έτσι. Δεν ζητούμε αλλαγή τη συμφωνία υποχώρηση. Ε, συζητάμε απλώς το τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστεί αυτή. Εκεί κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις βελτίωση. Μετά. Στην περίπτωση no deal, δηλαδή εξόδου χωρίς συμφωνία. Έτσι κι αλλιώ η συμφωνία αποχώρηση δεν έχει εγκριθεί μέχρι τώρα, δεν είναι σαφές, αν θα, δεν είναι σαφές ακόμα αν θα εγκριθεί μια τέτοια συμφωνία. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση ε, το ερώτημα τι θα γίνει αν δεν έχουμε μια συμφωνία, οποιαδήποτε, ούτε αυτή ούτε κάποια άλλη. Σε περίπτωση λοιπόν αποχώρησης χωρίς συμφωνία, Οι πολίτε εκατέρωθεν, μάλλον οι Ευρωπαίοι πολίτες του ΕΒ Βασίλειο, θα πρέπει να καταθέσουν αίτημα και πάλι για να τους χορηγηθεί καθεστώς εγκατάστασης. Το θέμα όμως τι γίνεται. Αν δεν έχουμε τη συμφωνία αποχώρησης, η κατάσταση αλλάζει. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν θα αποτελέσουν ε, προστασία προστατευτικές διατάξεις. Για παράδειγμα, μεταβατική περίοδος. Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περίοδου δεν υπάρχει καμία αλλαγή με τη συμφωνία, ενώ αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος. Οπότε αμέσως ε, θα πέσουμε στο οριστικό καθεστώς, αυτό που θα προβλεφθεί τελικά ε, κανονικά μετά από μια μεταβατική περίοδο. Χωρίς συμφωνία δεν υπάρχει μεταβατική περίοδος. Επίσης, χωρίς συμφωνία δεν υφίσταται προστασία επί τη βάση των διεθνών συνθήκων, γιατί όλα όσα είπαμε ε, βασίζονται σε μια διεθνή συμφωνία που θα υπογραφεί μεταξύ, Ηνωμένας, ε, μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν καταλήξουμε στη συμφωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο μόνο μερός μπορεί να αλλάξει το σύστημά του ε, και τον τρόπο με τον οποίο χορηγείται το καθεστώς της εγκατάστασης. Αύριο μπορεί το νομικό Βασίλειο να το αλλάξει μέσω υιοθέτηση ενό νομοθετικού κειμένου, αλλά να αλλάξει του όρου, τι προποθέσει, τα πάντα. Δεν υπάρχει καμία διεθνή συμφωνία η οποία να το κατοχυρώνει. Ε, ε, Επίσης δεν υπάρχει προστασία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία. Άρα ε, οποιαδήποτε προσφυγή μπορεί να γίνει μόνο εσωτερικά στο Ηνωμένο Βασίλειο ως ε, διοικητική νομική εξέταση. Επίσης δεν υπάρχει ανεξάρτητη αρχή παρακολούθησης ε, που να παρακολουθεί τη σοβαρότητα με την οποία εφαρμόζεται το σύστημα. Θα υπάρχουν πιο σύντομες προθεσμίες ε, ως προς τις ε, ε, τήσεις για χορήγηση καθεστώτος εγκατεστημένου και για τις οικογένειες από αυτές που είχαμε στην Συμφωνία για την Αποχώρηση. Επίσης θα υπάρξει μια προστασία των προνομίων, το οποίο όμως περιγράφεται από τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου ε, σε γενικές γραμμές με τους ίδιους όρους ως τώρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι ακριβώς οι ίδιοι οι όροι όπως τώρα, είναι σε γενικές γραμμές οι ίδιοι. Δεν ξέρουμε ποιες παροχές δεν θα καλύπτονται σε ένα τέτοιο σενάριο χωρίς συμφωνία. Θα υπάρχει μια έλλειψη συντονισμού στην κοινωνική ασφάλιση σε αυτή την περίπτωση. Είναι ξεκάθαρο λοιπόν ότι σε περίπτωση που δεν έχουμε συμφωνία θα έχουμε το σενάριο που θα δίνει στους Ευρωπαίους πολίτες το καθεστώς των κατεστημένων, αλλά χωρίς τις εξασφαλίσεις και τις προστασίες που θα έδινε μια ε, συμφωνία. Και σίγουρα χωρίς τις παροχές, ε, ε, καθώς δεν θα υπάρχει ο συντονισμός ε, στην κοινωνική ασφάλιση. Δεύτερον, θα υπάρχουν και επιπλέον ανησυχίες ως προς, υπάρχουν ανησυχίες ως προς τους πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι θέμα εθνικής αρμοδιότητας. Είναι διαφορετικά τα συστήματα στο κάθε κράτος μέλος, 27 κράτη-μέλη που προσπαθούμε να τα συντονίσουμε και θα συνεχίσουμε να προσπαθούμε να τα συντονίζουμε στο μέγιστο δυνατό. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σύστημα θα είναι το ίδιο ισότιμο και στα 27 κράτη-μέλη. Επίσης, όπως ξέρετε, στο ψήφισμά μας ζητήσαμε μέτρα τα οποία θα παράσχουν την νομική βεβαιότητα που θέλουν όχι μόνο οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και οι ε, πολίτες τη Μεγάλης Βρετανίας ε, που θα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και να έχει, με συμφωνία χωρίς, θα συνεχίσουμε εμείς ως ομάδα εργασίας να πιέζουμε το ομάδα εργασίας για το Brexit στο Συμβούλιο είναι κάτι παρά, συνήθως κάτι παράλληλο με το δικό μας, αλλά δεν είναι όπως είναι η διευθυντική ομάδα. Ε, ε συνήθως ε, εμείς δουλεύουμε και αυτοί καθοδηγούν, ε, σε αυτή την περίπτωση όμως πρέπει να δουλέψουν. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα δεν γίνονται πάντοτε με τον τρόπο που λέγονται. Επίσης, σε περίπτωση χωρίς, ε, που δεν θα έχουμε συμφωνία, οι περισσότερες χώρες θα δώσουν μια περίοδο χάριτος, όπως λέγεται, κατά την οποία τα περισσότερα δικαιώματα των πολιτών του, Μαγα... του Ηνωμένου Βασιλείου στη χώρα που τους φιλοξενεί θα παραμένουν τα ίδια. Μετά όμως από την περίοδο χάριτος θα πρέπει να ζητήσουν καθεστώς ε, παραμονής. Μάλλον αυτό θα γίνει στις περισσότερες χώρες. Όπως και να έχει λοιπόν, προσπαθούμε να πιέσουμε τα 27 κράτη-μέλη να πάνε όσο πιο μακριά γίνεται. Και εδώ επανέρχομαι στο θέμα του τι μπορεί να γίνει σε περίπτωση που δεν θα υπάρχει συμφωνία. Είπε ο κόσμος, τι θα κάνουμε. το κομμάτι στη συμφωνία της αποχώρησης ε, που μιλάει για τα δικαιώματα των πολιτών ε, θα το προσπίσουμε με μια διαφορετική συμφωνία που θα το διασφαλίζει ακόμα περαιτέρω. Το Ηνωμένο Βασίλειο δεν είναι πολύ ενθουσιώδης ε, ως προς αυτό το σημείο. Δεν θέλουν αυτό και δεν το θέλουμε κι εμείς γιατί δεν θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο ε, να επιλέγει ό,τι του αρέσει και να κάνει μια χωριστή συμφωνία γι' αυτό. Α, υπάρχει θέμα με τους πολίτες, κάνουμε εκεί μια συμφωνία. Υπάρχει θέμα με τις μεταφορές, ναι, ναι, να κάνουμε μια συμφωνία γι' αυτό. Α, και παρεπιπτόντος, για τα ψάρια υπάρχει ένα θέμα, να κάνουμε και εκεί μια συμφωνία. Και πριν το καταλάβουμε δεν έχουμε πια την ε, ε, δομημένη αυτή συμφωνία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις, αλλά έχουμε ένα πληθωρισμό μικρότερων συμφωνιών, όπου το Ηνωμένο Βασίλειο επιλέγει τα πλεονεκτήματά του χωρίς να έχει τις υποχρεώσεις. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε έναν τρόπο να προασπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών χωρίς να τα προασπίσουμε μέσω μιας έξτρα συμφωνίας και από τις δύο πλευρές να υπάρχει μια μονομερής δέσμευση είναι ο καλύτερος τρόπος. Μην το πείτε συμφωνία. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να πει, όχι να συμφωνήσει, να δηλώσει ότι θα καλύψει, ακόμα και σε περίπτωση έλλειψης συμφωνίας, ε, τα δικαιώματα, ως προβλέποντας τη συμφωνία αποχώρησης και μετά να το ε, εφαρμόσει ακριβώς όπως εμείς θέλουμε, δηλαδή να μην γίνονται μεμονωμένες αιτήσει. Και οι 27 μετά να κάνουν ακριβώς το ίδιο. Να πούν δηλαδή ο καθένας από την πλευρά του ότι μονομερός δεσμεύεται να σεβαστεί κάτι τέτοιο. Αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Μπορεί κάποιος να πει αυτό δεν είναι έτσι λίγο υπεκφυγή, να μην το λέμε ε, συμφωνία αλλά ε, δήλωση. Το σημαντικό είναι να υπάρχει μονομερής δήλωση και να καλύπτει τα δικαιώματα που προβλέπονται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Και η εφαρμογή να γίνεται καλύτερα από ό,τι γίνεται σήμερα για να αποφύγουμε αυτόν τον πληθωρισμό των mini deal, των μικρότερων συμφωνιών που κατά κάποιο τρόπο είναι ένα, μια μέθοδος να μπορεί το Ηνωμένο Βασίλειο να επιλέγει πλεονεκτικές συμφωνίες ε, στη μελλοντική του σχέση με μας. Αυτά έχω να πω. Συγγνώμη που μακρηγόρησα. Συνόψισα έτη εργασίας. Η κυρία Χιούμπνερ και ο κύριος Σταγιάννη ενεπλάκησαν και αυτοί σε αυτή την ε, συζήτηση Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Η κυρία Χιούμπνερ φαντάζομαι ότι θέλει και αυτή το λόγο. Είναι σχεδόν αδύνατο να προσθέσω οτιδήποτε αφόσον έχει μιλήσει ο Γκί. Αλλά υπάρχουν δύο-τρία πράγματα που θέλω να υπογραμμίσω γιατί είναι σημαντικά. Το no deal δεν είναι ο τελικός προορισμός ε, για το Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως και να έχει, στο μέλλον θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε κάτι. Επειδή η προσέγγιση λοιπόν χωρίς συμφωνία ε, δεν είναι λύση ούτε για τους πολίτες, ούτε για τα δημοσιονομικά, ούτε για το θέμα των συνόρων με την Ιρλανδία, Ιρλανδία καλό είναι ως προϋπόθεση πριν ξεκινήσουμε τη συζήτηση για την επόμενη συμφωνία, να έχουμε κάτι στο μυαλό μας για τους πολίτες. Το δεύτερο, που δεν ξέρω αν είναι ήταν ξεκάθαρο από αυτά που είπε ο Γκί, ενδεχομένως έμεσα να φάνηκε, έχει να κάνει με το γεγονός ότι έχουμε μόνο προφορικές υποσχέσεις από το Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν υπάρχει νομικό κείμενο από τον Δεκέμβρη του 2018 που ξεκίνησαν αυτά τα θέματα. Υπάρχουν μόνο πολιτικά κείμενα. Ε, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει ε, κάποιος νέος νόμος ε, για τη μετανάστευση. Ε, όπως ακούμε πολύ συχνά από Βρετανούς φίλους, ότι και να έχουμε δεν θα είναι δεσμευτικό για την επόμενη κυβέρνηση ή το επόμενο κοινοβούλιο. Αυτό μας ανησυχεί λοιπόν κάπως. Και επίσης είναι σημαντικό να πούμε ότι ίσως να μην είμαστε τέλειοι στην πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίπτωση της έλψης συμφωνίας, γιατί όπως είπαμε ότι είναι εθνικό το ζήτημα, αλλά από την πρώτη μέρα υπήρχε πίεση και από εμά και από την Κομισιόν ε, τα κράτη-μέλη να παράσχουν την πιο έτσι γενναιόδορη λύση ε, ως προς τους πολίτες ε, του, της Βρετανίας που ζουν στο έδαφος τους. Και υπάρχει και κάτι άλλο που θέλω να κρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί όλοι μας έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις με όλους τους ενδιαφερόμενους από το Ηνωμένο Βασίλειο και πρόσφατα Είχαμε και κάποια συνάντηση με ανθρώπους ε, που ενδιαφέρονταν για την αμοιβαία αναγνώριση των ε, επαγγελματικών προσόντων. Αυτό και πάλι θα είναι κάτι που θα εναπόκειται στην εθνική αρμοδιότητα και δικαιοδοσία. Πρόσφατα λοιπόν συζητήσαμε για το επάγγελμα του γιατρού. Η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν ήδη περάσει, δεν ξέρω αν έχουν οριστικοποιήσει μια συμφωνία η οποία έχουν εξετάσει ή δεν έχουν οριστικοποιήσει μια συμφωνία η οποία έχει να κάνει με την αμοιβαία αναγνώριση των προσόντων του γιατρού. Επίσης, δεν ξέρω προσωπικά ο καθένας σας πόσο πολιτικά εμπλέκεστε στο θέμα, αλλά στην πατρίδα σας καλό θα ήταν να δείξετε το θέμα των φοιτητών που ξεκινάνε στο Ηνωμένο Βασίλειο να σπουδάζουν και μετά επανέρχονται στις χώρες μας ε, με κάποια προσόντα. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Uh, mm, Συγγνώμη που μίλησα στα ισπανικά. Στην Επιτροπή ΑΦΚΟ την επόμενη εβδομάδα θα διοργανώσουμε μία ακρόαση με τον Οργανισμό των Ευρωπαίων Πολιτών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς πολίτες που ζουν στην Ευρώπη. Είστε προσκεκλημένοι και εσείς, το Προεδρείο και βεβαίως η συζήτηση είναι ανοιχτή για όλα τα μέλη, αλλά ήθελα να σας προσκαλέσω, να προσκαλέσω την Πρόεδρο της Επιτροπής ΠΕΤΗ, και τα άλλα μέλη του Προεδρείου. Πιστεύω ότι είναι ένα ισχυρό μήνυμα από την ΑΦΚΟ στους Ευρωπαίους πολίτες, γιατί θέλουμε να ενδυναμώσουμε τα δικαιώματά τους, τα δικαιώματα των α, Ευρωπαίων που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, 3,6 εκατομμύρια περίπου, αλλά και ένα εκατομμύριο περίπου Βρετανοί που ζουν στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα αυτό, ούτω ώστε να ξέρετε, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, υπάρχουν πολλά προβλήματα στην ε, Βόρεια Ιρλανδία. Πολλά άτομα που προέρχονται από τη χώρα αυτή ζουν στη Βόρεια Ιρλανδία. Θέλουμε να ακουστούν οι φωνές τους, οι φωνές των οργανώσεων αυτών, των ατόμων αυτών, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών, τα δικαιώματα των Βρετανών πολιτών είναι προτεραιότητα για μας. Επομένως η ακρόαση αυτή είναι πολύ σημαντική. Και επίσης πιστεύω ότι και η ακρόαση σήμερα εδώ στη δική σας την Επιτροπή είναι ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Όλοι στο κοινοβούλιο αυτό θέλουν να προστατεύσουν τους πολίτες στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ευχαριστούμε πολύ. Πάντοτε λέμε όχι ως Επιτροπή πέτει ότι είμαστε γέφυρα εμείς μεταξύ των πολιτών και των ε, θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό λοιπόν και λαμβάνουμε πολλές αναφορές, ε, ανησυχούν οι πολίτες σε σχέση με τον Brexit. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα ανοίξαμε τη συζήτηση αυτή και στη συνέχεια έχουμε και άτομα που θα παρουσιάσουν τις αναφορές τους από όλη την Ευρώπη που μας ζητάνε να τους βοηθήσουμε. Επομένως σας ευχαριστούμε πραγματικά τώρα ε, δίνουμε το λόγο στα μέλη της Επιτροπής αυτής. Η κυρία Κύρτον πρώτη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, λέει. Και ευχαριστώ πολύ και στους ο, τρεις σας που είστε σήμερα εδώ. Δουλεύουμε ήδη πριν από το δημοψήφισμα. Ήδη κυρίως ό,τι αφορά τα δικαιώματα ψήφου που είναι ένα από τα βασικά ζητήματα που εκκρεμούν. Και με 30 μέρες δυνητικά μπροστά μας και ένα Brexit χωρίς συμφωνία, το επίπεδο ανησυχίας σε σχέση με τον Brexit πραγματικά εντατικοποιείται. Και η πολιτική αστάθεια στη Βρετανία αυτή τη στιγμή δεν βοηθάει και θέλω να θέσω επιτάπητος επίσης ότι και η ρητορική και ο τόνος α, της κυβέρνησης όταν μιλάνε για ελεύθερη μετακίνηση και όταν μιλάνε και για τα δικαιώματα των πολιτών επίσης δεν βοηθάει το επίπεδο αγωνίας των πολιτών σε σχέση με το τι συμβαίνει επί της ουσίας. Έχοντας λοιπόν αναφέρει όλα αυτά, πιστεύω ότι παρουσιάσατε πολύ αποτελεσματικά όλα τα πιθανά σενάρια και έχω ένα σχόλιο για σας και στη συνέχεια θα παρουσιάσω και μία από τις αναφορές σε ένα από τα επόμενα σημεία της ατζέντα μας. Θέλω λοιπόν να αναφερθώ σε αυτό ακριβώς το σημείο και όχι στις δικές μου ανησυχίες. Σε τι αναφέρομαι. Τα δικαιώματα των πολιτών που δεν μπορούν να είναι μια επιμέρους συμφωνία. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων αυτών δηλώνει ότι οι πολίτες που έχουν στηρίξει την εμπιστοσύνη τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχουν αξιοποιήσει την ελεύθερη μετακίνηση, που έχουν δείξει την επιθυμία τους να, να επωφεληθούν από όλα όσα τους προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν θα πρέπει να τιμωρηθούν από την κατάσταση αυτή στην οποία βρίσκονται άθελά τους είτε πρόκειται σε ό,τι αφορά την ψηφοφορία στο δημοψήφισμα, είτε ήταν κάτοικοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκτός Ηνωμένου Βασιλείου είτε ζούσαν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά τα άτομα θα πρέπει να είναι η ηθική μας πηξίδα. Ο προσανατολισμός μας θα πρέπει πάντοτε να έχει κατά νου τα άτομα αυτά γιατί επί τη ουσία εδώ δεν έχουμε τεχνικές αποφάσεις, έχουμε τη συγκεκριμένη ζωή των ανθρώπων και η αγωνία που τους καταβάλει αυτή τη στιγμή τους πολίτες αυτούς είναι πραγματικά ιδιαίτερα υψηλή. Ανησυχούν, ανησυχούν και πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη μας. Αναγνωρίζω ότι υπάρχει πρόοδο σε ό,τι αφορά την προστασία των δικαιωμάτων τους. Θα ήταν καλύτερα αν στο Στρασβούργο από κοινού ως κοινοβούλιο είχαμε αναφερθεί στην προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών αυτών για τους συγκεκριμένους λόγους. Ανησυχία μου είναι ότι η πρόταση για μονομερείς δηλώσεις, συμφωνίες είναι κάτι το οποίο τελικά δεν λαμβάνει υπόψη τους πολίτες. Αν λάβουμε υπόψη μας τα 3 εκατομμύρια που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, το πρόβλημα τους είναι ότι οι μελλοντικέ κυβερνήσεις θα επιβαρύνουν τις συνθήκες διαβίωσής τους δεν θα υπάρξει κάτι σε μια μονομερή πρωτοβουλία που να επιλύει τις διαφωνίες αυτές. Πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα πλαίσιο που να εξασφαλίζει ότι ε, μια μελλοντική κυβέρνηση, για παράδειγμα, θα μπορούσε να αλλάξει τελείως τα δεδομένα. Αυτό είναι ένα ερώτημα που έχω για σας. Και από την άλλη μεριά, σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς τις χώρες της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, βλέπουμε ένα μείγμα διαφόρων μεθόδων, διαφορετικής μεταχείρισης. Θα ήταν ένα ισχυρό σήμα από πλευρά Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν μπορούσαμε να πούμε ότι θα πρέπει να εναρμονιστούν όλες αυτές οι μέθοδοι. Θα ήταν ένα σήμα ότι όντως στηρίζουμε τα άτομα που έχουν επωφεληθεί της ελεύθερης μετακίνησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ερωτευτούν, να κάνουν τις οικογένειές τους, να σπουδάσουν, να δουλέψουν. Πρέπει να γιορτάσουμε αυτό το ευρωπαϊκό ιδανικό, αντί ε, να συμβαίνει αυτό που βλέπουμε. Τα άτομα που επωφελήθηκαν των δυνατοτήτων αυτών τώρα βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου πραγματικά έχουν να αντιμετωπίσουν ένα τεράστιο βαθμό αγωνία σχετικά με το τι μελγενέστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μοράλες, έχετε το λόγο. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε και την Επιτροπή Αναφορών για τη συζήτηση αυτή με τους συναδέλφους μας. Ε, με ενδιαφέρει πραγματικά γιατί έχω βρεθεί σε πολλές από τις συνεδριάσεις της ε, παρούσας ε, Επιτροπής αλλά και της ΛΥΜΠΕ. Και πιο συγκεκριμένα, σε σχέση με όλα όσα είπε ο κύριος Φαγιάν και ο κύριος Βερχόφσταπ, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να ζητάμε ένα ξεκάθαρο σύστημα. Η κυρία Κέρτιν αναφέρεται σε μελλοντικά δυσάρεστα σενάρια. Αν θέλουμε να είμαστε δίκαιοι, ο Γκίβερ Χόφστα καταλαβαίνει αυτή την, την ιδέα της εθνικότητας. Αν δεν έχουμε όμως ένα σύστημα εγγραφής και δήλωσης και δεν στηρίξουμε το σύστημα αυτό με πραγματική νομοθεσία, τότε μπορεί να προκύψουν προβλήματα κακοδιαχείρισης. Επομένως, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ακροάσεις σχετικά με το Brexit, συζητήσεις σχετικά με το Brexit έχουν στόχο να βελτιώσουν τη θέση των πολιτών, τα δικαιώματα των πολιτών για τα τρία εκατομμύρια άτομα που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και για τους Βρετανούς που ζουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και θέλω να επαναλάβω αυτό που είπε ο Βερχόφστατ, γιατί θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το κρατήσουμε στο μυαλό μας. Το ζήτημα που προκύπτει για μας είναι πολυμερές και η Κέρν αναφέρθηκε στο σημείο αυτό. Πρώτα απ' όλα, η διαρκής δυσκολία που αντιμετωπίζουν τα 3 εκατομμύρια Ευρωπαίοι στο Ηνωμένο Βασίλειο και οι Βρετανοί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιε είναι οι παρούσε δυσκολίε που αντιμετωπίζουν στο τρέχον σύστημα εγγραφής, στο πρόγραμμα εγκατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτοί είναι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμη είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα περάσω στη, στο σενάριο no deal Brexit, αλλά προς το παρόν δεν θα πρέπει να ενδυναμώνουμε φόβους, αλλά και να ενισχύουμε αυτή τη ρητορική στην οποία αναφέρθηκε και η συνάδελφος. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε το σημείο αυτό, γιατί η ρητορική είναι σε τόσο κακό χρονικό σημείο σε ό,τι αφορά την ελεύθερη μετακίνηση που έχει πραγματικά άμεσο αντίκρισμα στο πώς αισθάνονται όλα αυτά τα άτομα. Υπάρχει μια απτή αλλαγή στο πώς αισθάνονται όλα αυτά τα άτομα. Κάτι το οποίο με φέρνει και στο τελευταίο σημείο που θέλω να, να θίξω. Δεν θέλω να εκμεταλλευτώ το χρόνο γιατί ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν. Το ζήτημα λοιπόν που εμένει είναι πώς θα προστατέψουμε τους Βρετανούς, τους Ευρωπαίους πολίτες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και όσους ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένως, θέλω να εγγραφεί επισήμως. Αποδέχομαι ότι όταν συζητάμε τη Συμφωνία Αποχώρησης και όταν συζητάμε όλα αυτά τα πράγματα με το Ηνωμένο Βασίλειο, αυτή η ιδέα του να επιλέγονται επιμέρους συμφωνίες ήταν κάτι το οποίο είχε προκύψει. Αλλά σε ό,τι αφορά το ζήτημα αυτό της προστασίας σε ενδυνάμωσης των δικαιωμάτων των πολιτών, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Και ξέρω ότι είναι κάτι για το οποίο είναι πεπισμένη και η Επιτροπή για το Brexit. Το ζήτημα της νομοθεσίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε ακούσει όλοι και το Windrush, ο Γκίβερ Χόφσταντ έχει αναφερθεί στο ζήτημα αυτό πάρα πολλές φορές. Γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί δεν υπάρχει νομική προστασία και ποιο είναι τώρα το ηθικό ζήτημα που προκύπτει. Αν ενδυναμώσουμε τα δικαιώματα αυτά, τότε θα έχουμε και την ανάλογη νομική προστασία. Να έχουμε ένα ανεξάρτητο σώμα εποπτείας, για παράδειγμα, γιατί αν δεν έχουμε το αυτό, τότε τι έχουμε. Είναι κάτι το οποίο μπορεί να εξασφαλίσει σιγουριά για το μέλλον, για, για τα μέλη της κάθε οικογένειας. Αυτό είναι κάτι το οποίο έχει συμβεί σε πολλα κάτι κράτη-μέλη της Ευρώπης, ιδίω αυτά που, που είχαν άλλοτε απικίες και έχουν αντιμετωπίσει το ζήτημα της επανένωσης οικογενειών κτλ. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την ενδυνάμωση των δικαιωμάτων, την προστασία των δικαιωμάτων, έχουν γίνει συζητήσεις και σε διάφορα εθνικά κοινοβούλια και πραγματικά το εκτιμώ ότι κάνετε μια προσπάθεια εδώ να μιλήσουμε και για μονομερίσα μονομερείς πρωτοβουλίες, αλλά αυτό που θα έλεγα εγώ είναι ότι χρειαζόμαστε προστασία από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί στο μέλλον θα πρέπει να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα. Και αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι με δεδομένο τη ρητορική στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι ανάγκη να επιμείνουμε σε αυτό το θέμα. Σας εγκαλώ λοιπόν να το, να το σκεφτείτε περισσότερο. Είναι μια μαρτυρία το γεγονός ότι σε αυτό εδώ το κοινοβούλιο βασιζόμαστε στα δικαιώματα των πολιτών. Και γι' αυτό το λόγο σας ζητώ να εξετάσετε και πάλι αυτό το ζήτημα της απόλυτης προστασίας. Ξέρω ότι η πρόθεσή σας, στην καρδιά σας το καταλαβαίνετε, αλλά έχετε αυτό το φόβο των επιμέρους συμφωνιών. Πρόεδρε, λοιπόν, θέλω πραγματικά να σας πω ότι μπορεί να καταλήξουμε σε, μια, ένα Brexit χωρίς συμφωνία υπάρχουν πάμπολοι πολίτες που θέλουν, περιμένουν από το Κοινοβούλιο να τους δώσει μια λύση, γιατί έχει γίνει τόσο μεγάλη προσπάθεια προστασίας των δικαιωμάτων τους μέχρι στιγμής. Ευχαριστώ. Ο, ο λόγος του κυρία Φομβάισε. Για 22 χρόνια ε, έζησα ως Γερμανίδα στον Βασίλειο και στο τέλος ε, έλαβα και την υπηκότητα, οπότε τώρα εκπροσωπώ το Ηνωμένο Βασίλειο. Καταλαβαίνω λοιπόν πολύ καλά τι σημαίνει η ανασφάλεια των αλλοδαπών πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο σήμερα. Ε, εγώ όλα αυτά τα χρόνια όχι, ήμουν ελεύθερη, όχι μόνο ήμουν ελεύθερη να κυκλοφορώ, αλλά αναγνωρίστηκαν και τα επαγγελματικά μου προσόντα. Κατάφερα λοιπόν να κάνω τη ζωή μου στο Ηνωμένο Βασίλειο και τα τελευταία χρόνια αντελήφθη ότι Οι σχέσει ε, με το Υπουργείο Εσωτερικών γινόντουσαν όλο και πιο δύσκολες ε, γραφειοκρατικά ενώ ε, άργησα χρόνια να καταφέρω να βγάλω διαβατήριο, βρετανικό διαβατήριο για την κόρη μου που γεννήθηκε στον Ηνωμένο Βασίλειο και είναι κόρη δύο Ευρωπαίων πολιτών. Υπάρχουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στον Ηνωμένο Βασίλειο σε μια ανασφαλή κατάσταση. Ε, εκτιμάται ότι 40% των όσων ε, έκαναν αίτηση για καθεστώς εγκατάστασης έλαβαν το προσωρινό καθεστώς. Ε, αυτοί, περισσότεροι από αυτούς ζουν στον Βασίλειο πάνω από 20 χρόνια. Αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ανασφάλεια και άγχος στους Ευρωπαίους πολίτες. Ο Μπόρις Τζόνσον υποσχέθηκε ότι θα εξασφαλίσει απόλυτη σαφήνεια για το καθεστώς τους. Παρ' αυτά, όπως και με άλλες υποσχέσεις του δεν φαίνεται να την υλοποιεί ούτε αυτήν. Χαίρομαι που ο Κίφερ Χόφστατ είναι εδώ, αντί να διαβάζει αυτό το έγγραφο το οποίο από ό,τι φαίνεται έφτασε από τη Βρετανική κυβέρνηση και προτείνει κάποια καινούρια υποτιθέμενη λύση. Δεν γνωρίζουμε προφανώς το αποτέλεσμα, το περιεχόμενο. Δυστυχώ, ο κύριος Φώσταν μιλάει εκτός μικροφώνου, δεν τον ακούμε. Ας υποθέσουμε ότι αυτό το καινούριο έγγραφο δεν θα είναι και κάποια επανάσταση για του Ευρωπαίου πολίτες, οπότε θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που είπαν οι προηγούμενες ομιλητρίες τα εξής. Η μόνη συμφωνία με τους 27 και που εγκρίθηκε από το Βρετανικό Κοινοβούλιο ε, δεν εφαρμόζεται. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, πολλοί αναφέροντες λένε ότι υπάρχουν κενά. Οπότε θα μπορούσε να μου πει η Κομισιόν για ποιο λόγο δεν έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα κενά. Επίσης θα ήθελα να στηρίξω το αίτημα της η, προστασία των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών να αποτελέσει αντικείμενο μιας πραγματικής συμφωνίας, επίσημης συμφωνίας, ε, έτσι ώστε να μην γίνουν πιόνια στην, σε, μια, σε ένα πολιτικό σκάκι. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κυρία Τόμ. Ευχαριστώ πολύ τα μέλη της διευθύνουσας ομάδας που είναι εδώ. Ε, δεν θα κάνω κάποια πολιτική δήλωση αυτή τη στιγμή. Επικρατεί έτσι κι αλλιώς μια ατμόσφαιρα νεκρικής ε, ε, ε ελκυδίας μάλλον. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια επικυρωμένη συμφωνία. Βρισκόμαστε στο πεδίο των διμερών συμφωνιών μόνο. Κάτι που προφανώ δημιουργεί πολλέ ανησυχίε. Ε, είναι ολιστήρο έδαφο. Δεν ξέρουμε πόσο μακριά θα μπορεί κανεί να πάει με διμερείς συμφωνίες. Ακούγεται ότι και στην Εστονία έγιναν κάποιες συναντήσεις με τους Βρετανούς. Δεν είμαστε μόνοι μας λοιπόν εμείς. Δεν ξέρω τι μέτρα θα πρέπει να λάβουμε έτσι ώστε να μείνουμε ενωμένοι και να έχουμε μία ενιαία αντιμετώπιση εμείς ως υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν ξέρω ε, αν θα υπάρχει σημείο επιστροφής από τις ε, διμερείς συμφωνίες αν αυτές προχωρήσουν. Δεν θέλω να είμαι απεσιόδοξη, απλά πιστεύω ότι είναι σημαντικό να, το, να σας ρωτήσω αν έχετε κάποιο άλλο εναλλακτικό σχέδιο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ντανούκα. Η κυρία Στανόκα, συγγνώμη. Ήμουν στη Λίμπε και ο, ο Κλοντ Μωράης θα θυμάται ε, υπήρχε και, η, η, και άλλη προηγούμενη έκθεση του Κατάνη ε, και οι δικοί μου και οι άλλοι απέτυχαν ως προτάσεις Είναι καθήκον μας να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε αυτά τα προβλήματα για τα οποία μιλάμε. Και πώς θα τα αποφύγουμε, με την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, η οποία θα δίνει αυτόματα δικαιώματα και δεν θα είναι μια απλή αυτόματη προέκταση της εθνικής υπηκότητας. Δεν πιστεύω σε μονομερείς ή διμερείς συμφωνίες. Ούτε σε μονομερείς δεσμεύσεις, σε διμερείς συμφωνίες. Στην, ε, πριν από 15 χρόνια, όταν προσχώρησαν η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία, είχαμε συζητήσει για το θέμα της, ε, του φόβου να βρεθούν οι πολίτες χωρίς καμία ηθαγένεια. Από τότε δεν έχει συμβεί τίποτα για την ευρωπαϊκή ηθαγένεια. My Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρουίτε Μέσα. Συμμετέχω σήμερα με διπλό ρόλο αντικαταστάτης ε, στην Επιτροπή Αναφορών αλλά και μέλος, τακτικό μέλος της Επιτροπής Συνταγματικών Θεμάτων. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή Αναφορών που διοργάνωσε αυτή την συνεδρία και είναι πολύ χρήσιμο που έχουμε μαζί μας τρία από τα μέλη της διευθύνουσας ομάδας συμπεριλαμβανομένου και του Προέδρου της, του κ. Φερχόφστατ, τον οποίο ευχαριστώ για την πολύ λεπτομερή και εκτενή παρουσίαση των πρακτικών πτυχών του Brexit, ιδιαίτερα του σκληρού Brexit για τα δικαιώματα των πολιτών μας. Δεύτερον, μια και έχουμε παρόντες κάποιους αναφέροντες, θα ήθελα καταρχήν να τους ευχαριστήσω και να τους εκφράσω την αλληλεγγύη μου, όπως και την αλληλεγγύη προς όλους τους ε, πολίτες μας που βρίσκονται στη Βρετανία και τους Βρετανούς ε, πολίτες που βρίσκονται στα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Και το λέω αυτό γιατί έχουμε όλοι εκλεγεί στη χώρα του ο καθένας. Δεν έχουμε διεθνείς εκλογικές περιφέρειες, αλλά Παρόλο που έχουμε εκλεγεί ο καθένα στη χώρα του, εκπροσωπούμε τα συμφέροντα όλων των πολιτών τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω εκλεγεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά έχω τι ίδιε ανησυχίες που έχουν οι Βρετανοί Ευρωβουλευτές για του Βρετανού πολίτε. Θα ακούσουμε λοιπόν και του αναφέροντε. αλλά χωρίς να μπω στη λεπτομέρεια των ετοιμάτων τους, θα ήθελα να επαναλάβω πως το δημοψήφισμα ήταν ε, κακή ιδέα και όχι μόνο το ίδιο το δημοψήφισμα αλλά και το αποτέλεσμα. Λέω το δημοψήφισμα όμως γιατί αναλύουμε αυτή τη στιγμή τα προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν οι πολίτες εξαιτία του Brexit. Και αυτό είναι αποτέλεσμα της σύγκρουσης δύο αρχών. Η αρχή των δικαιωμάτων και με την αρχή της πλειοψηφίας. Όλοι γνωρίζουμε τις βάσεις τα θεμέλια της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Το, η φιλελεύθερη δημοκρατία δεν ε, βασίζεται μόνο στην πλειοψηφία. Βασίζεται ταυτόχρονα και σε μια χάρτα δικαιωμάτων τα οποία καμία πλειοψηφία δεν μπορεί να παραβεί ή να αποφασίσει να καταργήσει ε, ή να περιορίσει. Τι έγινε με το Brexit, με το δημοψήφισμα του Brexit. Η πλειοψηφία, μια ε, περιορισμένη πλειοψηφία, αποφάσισε όλοι να χάσουν τα δικαιώματά τους ως ε, ε, Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί η, το καθεστώς του μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, αυτόματα συνεπάγεται συγκεκριμένα δικαιώματα για τους πολίτες της συγκεκριμένης χώρας. Ιδιαίτερα δε σε μια χώρα στην οποία δεν υπάρχει σύνταγμα, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Το ίδιο θα συνέβαινε με ένα δημοψήφισμα, όπως αυτό που συζητείτο για την απόσχηση της ε, Καταλωνίας από την Ισπανία. Ε, θα, μια τέτοιου είδους απόφαση θα αποτελούσε πλήγμα στα δικαιώματα πάρα πολλών πολιτών. Οπότε τα δικαιώματα των πολιτών δεν θα έπρεπε να επηρεαστούν από μια απόφαση που αποτελεί αποτέλεσμα ενός δημοψηφίσματος, μιας εκλογική διαδικασία. Επίσης, δεν ελήφθη καθόλου υπόψη το εξή. ότι το αποτέλεσμα αυτό του δημοψηφίσματος ερχόταν σε σύγκρουση με την Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής που ρύθμισε το καθεστώς στην Ιρλανδία. Μεταξύ της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Οπότε και εμείς ως Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με το άρθρο 50. Το άρθρο 50 είναι σχετικά καινούριο. Ε, ήταν άρθρο που προέκυψε με τη συνθήκη της Αβώνας. Δεν είμαι σίγουρος ήταν καλή ιδέα. Αυτό το άρθρο δεν προέβλεψε το, τα προβλήματα τα οποία θα δημιουργούνται με την εφαρμογή του. Επίσης, σε ό,τι αφορά το θέμα της προάσπισης και εξασφάλισης των δικαιωμάτων των πολιτών, το ονομαζόμενο ring fencing, Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης ή της διαχείρισης μιας συμφωνίας δεν θα πρέπει να διολυστήσουμε προς την κατεύθυνση των πολλών μικρών συμφωνιών. Σωστό αυτό, αλλά ίσως πρέπει να κάνουμε μία εξαίρεση και αυτή θα ήταν για τα δικαιώματα των πολιτών. Μία παράλληλη, διπλή, μονομερή δέσμευση, ας πούμε, ίσως θα μπορούσε να αποτελέσει λύση. Σίγουρα δεν μπορούμε να εξισώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών με την αλληλεία, με τις μεταφορές ή με άλλους τομείς που είναι σημαντικοί αλλά όχι παρόμοιοι. Γιατί αυτό που πραγματικά μας ενώνει όλους είναι το άρθρο 2 της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ añadiría una cosa de lo que Θα πρόσθετα το εξή, όχι μόνο δεν υπάρχει πολιτική πλειοψηφία στην Καταλωνία για γίνει ένα δημοψήφισμα, πολύ περισσότερο ότι δεν υπάρχει δικαίωμα διοργάνωση δημοψηφίσματος εκ μέρους της Καταλωνία στην Ισπανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ σημαντική και ευχαριστώ που δίνετε το λόγο σε έναν από τα τρία εκατομμύρια. Είμαι Γάλλος πολίτης και εκπροσωπώ την ε, Σκοτία εδώ ως Ευρωβουλευτής και θα ζήσω κι εγώ αυτό τον ε, φιάλτη που είναι το Brexit. Ε, σας ευχαριστώ καταρχάς όλους για την αλληλεγγύη σας, αλλά δεν μου αρκεί η αλληλεγγύη. Όπως ακούσαμε, αυτό που ζητούμε είναι η... τα τρία εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν στην ε, Βρετανία και οι Βρετανοί στην Ευρώπη. Αυτό που ζητούν είναι κάτι παραπάνω από αλληλεγγύη. Θα συνεχίσω στα αγγλικά, παρόλο που δεν είναι τόσο καλά σε τα γαλλικά μου των 35 ετών. Νομίζω ότι αυτό το καθεστώς του εγκατεστημένου δεν είναι ε, αρκετό για μας. Ε, δεν θα κάνω τέτοια αίτηση, αρνούμε να την κάνω. Ξέρω ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να μείνουμε στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2020, αν δεν υπάρξει συμφωνία και παραπάνω αν υπάρξει. Εγώ δεν θέλω ούτε συμφωνία ούτε ε, έλλειψη συμφωνίας. Θέλω να μείνει το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό θέλω από την πλευρά μου. Νομίζω όμως ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τις επόμενες μέρες, αν όχι εβδομάδες, να δείξουμε κάτι παραπάνω. Όχι απλώς αλληλεγγύη προς τους πολίτες ε, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρώπη και, τον, και στους άλλους πολίτες της Ευρώπης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Εδώ και 3,5 χρόνια υποφέρουμε. Έχω το δικό μου παράδειγμα, αλλά το κάθε παράδειγμα είναι διαφορετικό. Κάθε κατάσταση σε κάθε οικογένεια είναι διαφορετική. Εγώ θέλω επέκταση ένα ή δύο χρόνια για να λυθεί το θέμα του Brexit και ε, ίσως και να μην φύγει ε, το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ό,τι γίνει όμως δεν πρέπει να είναι εις βάρος των ανθρώπων ε, και των οικογενειών στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το ring fencing λοιπόν είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να είναι στο πρωτογενές και όχι στο δευτερογενές, στο παράγωγο δίκαιο αυτή η προάσπιση με επιπλέον συμφωνία. Αυτό ε, που έκανα εγώ όταν πήγα στο Ηνωμένο Βασίλειο, έκανα τρία παιδιά και τέσσερα εγγόνια, πήγα να βρω τη γυναίκα μου. Όταν το έκανα αυτό, κάτι σήμαινε για μένα. Κάτι πρέπει να σημαίνει λοιπόν για μένα, για τα τρία εκατομμύρια. Ο κόσμος μας παρακολουθεί. Πρέπει να προσέξουμε τους πολίτες μας πρέπει να γίνει με νομοθεσία και ζητώ από τον Γκίφερος Φέρχοφσταντ και όλους τους υπόλοιπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να μην κοιτούν τον Μπόρις Τζόνσον για τη λύση. Να βρουν τη λύση τώρα μέσα στην νομοθεσία ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματά μας και να μην πρέπει να κάνουμε αίτηση για ε, καθεστώς εγκατεστημένου. Να έχουμε μια πιο απλή διαδικασία. Εμείς ξέρουμε και πρέπει να ξέρουμε, χρειαζόμαστε να ξέρουμε ότι θα είναι τα δικαιώματά μας προστατευμένα ό,τι και να γίνει. Ο κύριος Η κυρία Απορίτ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μια πολύ συγκινησιακή είναι αυτή η συζήτηση. Υπάρχουν άνθρωποι σε αυτή τη διαδικασία. Όπως είπε και ο συνάλφος, υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα για την εγκατάσταση, γιατί αν έχεις πάει κάπου και ζεις εκεί, καλή την πίστη εδώ και δεκαετίες, είναι πραγματικά προσβολή να πρέπει να επαναδιατυπώσει το δικαίωμά σου να βρίσκεσαι εκεί ούτως ή άλλως. Να θυμόμαστε επίσης ότι όλα αυτά συνέβησαν μέσα στα πλαίσια μιας συνεχούς διάβρωσης των δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των ε, Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το δημοψήφισμα και μετά. Αλλά και πριν το δημοψήφισμα υπήρχαν άνθρωποι που δεν είχαν δικαίωμα τελικά να ψηφίσουν και να επηρεάσουν και αυτό που ψηφίστηκε επηρεάζει πλέον τη ζωή τους. Πολλοί από αυτούς δεν μπόρεσαν καν να αποφανθούν στις ευρωπαϊκές εκλογές με την ψήφο τους. Και τώρα υπάρχουν και άλλα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν ε, διαπιστωθεί και για, με το πρόγραμμα εγκατάστασης. Δεν είναι ωραίο να ζεις σε ένα περιβάλλον που δεν αισθάνεσαι ευπρόσδεκτος. Και είναι πολύ σημαντικό να ξέρει κανείς και να αναγνωρίζει ότι το περιβάλλον στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχώς επιδεινώνεται. Πριν από λίγο καιρό, ένα ε, ζευγάρι Ισπανών που ζούσε στην επόμενη γωνία από το σπίτι μου, μου είπαν ότι πάνε πίσω στη Μαδρίτη, γιατί δεν αισθάνονται πια ευπρόσδεκτοι. Και τώρα έχουμε τον Υπουργό Εσωτερικών που γιορτάζει το τέλος της ελεύθερης κίνησης και διακίνησης ανθρώπων. Ε, σαν να είναι κάτι σπουδαίο, ενώ δεν είναι κάτι που πρέπει να γιορτάζουμε. Η κυρία ε, Κίτον μίλησε για το θέμα. Ε, μιλάμε για ανθρώπους εδώ, μιλάμε για τις ζωές τους. Είναι πολλά τα παραδείγματα που δείχνουν πόσο δύσκολο είναι να ζήσουν μέσα σε αυτή την βεβαιότητα. Όσοι πεπισμένοι λοιπόν Ευρωπαίοι εμείς, ανεξάρτητα από το ποια είναι η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει κάτι να κάνουμε. Πρέπει να κάνω και ποιες ερωτήσεις και στον Γκί. Ανάφερες μια περίοδο χάριτος. Αυτό αν δεν υπάρχει συμφωνία... Και αν έτσι είναι τα πράγματα, φοβάμαι ότι αυτή είναι άλλη μία ιδέα που δεν έχει καθοριστεί έτσι επακριβώς, ενώ είμαστε μόλις ε, λίγες εβδομάδες πριν να συμβεί. Και τι θα γίνει μετά. Μιλάτε με μια κυβέρνηση η οποία δεν μπαίνει σε επικοδομητικές διαπραγματεύσεις. Είναι ανησυχητικός δείκτης αυτός. Μπορεί τελικά να έχουμε περισσότερη αβεβαιότητα και λίγο, λίγη πρόοδο για τους ανθρώπους που θα επηρεαστεί η ζωή τους. Επίσης αναρωτιέμαι γιατί η Βρετανική κυβέρνηση ως τώρα δεν θέλει να προσυπογράψει την αυτόματη κατα... εγγραφή. Πώς αυτό επηρεάζει την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επίσης, αυτό που φαίνεται ούτως ή άλλως και τονίζεται είναι ότι αυτά τα ζητήματα δύσκολα αντιμετωπίζονται. Τώρα λοιπόν να πιέσουμε για μονομερείς δηλώσεις, ανεξάρτητα με το τι θα συμβεί ε, με τη, σχετικά με την επέκταση της περίοδου πριν τη συμφωνία κτλ. Η κυρία Ρόι. Νομίζω ότι ο αριθμός των αναφορών που βλέπουμε προκύπτει από το γεγονός ότι υπάρχουν πάρα πολλά χαρακτηριστικά σε αυτή την κατάσταση που υπάρχει αυτή, στο, αυτή τη στιγμή στο Ενωμένο Βασίλειο που είναι ανησυχητικά. Και αυτά ισχύουν είτε έχουμε συμφωνία είτε όχι. Υπάρχουν τουλάχιστον τρία πράγματα για τα οποία δεν υπήρξε δημοκρατική εντολή, ακόμα και αν κανείς σεβαστεί το δημοψήφισμα, που δεν θα πρέπει μάλλον το σεβαστούμε. Δεν είχαμε ψηφοφορία σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο εχθρικό περιβάλλον σαν αυτό που έχει τώρα και το πανηγυρίζει η κυβέρνησή μας και ο Υπουργός Εσωτερικών υπό την Τερέζα Μέη. Δεν είναι κάτι που μας ζήτησε η πατρίδα μας ποτέ να προσυπογράψουμε. Επίσης δεν μας ρώτησαν Ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές που πρέπει να μπουν μέσα στην συμφωνία της Τερέζα Μέη. Έβαλε την ελευθερία των κινήσεων ως ένα κομμάτι αυτών των κόκκινων γραμμών χωρίς να συμβουλευτεί τους πολίτες της. Και αυτή η κυβέρνηση τώρα που δεν έχει νομιμοποιηθεί από πλειοψηφία κατά τη γνώμη μας γιατί παίρνει τα δικαιώματά μας, ε, τα, μας τα αφαιρεί χωρίς να έχει το δικαίωμα. Ε, πολλά από τα πανηγυρικά που κάνεις αυτό βασίζονται. Επίσης υπάρχουν ε, πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και Βρετανοί πολίτες που ζουν στην Ευρώπη. Για αυτούς είναι σημαντικό να σκεφτούμε ότι δεν πρέπει να αφήσουμε στο έλεος μιας κυβέρνησης ε, που δεν έχει πολιτική ε, αυτούς τους ανθρώπους. Αν αφήσετε αυτούς στο έλεος της κυβέρνησης θα αφήσετε και εμάς στο έλεος της μοίρας μας που δεν έχουμε να πού να πάμε. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που το σπίτι τους είναι στο Ηνωμένο Βασίλειο εδώ και πάρα πολλά χρόνια θα πρέπει να πάνε πίσω στο πρώτο σπίτι τους. Εμείς όμως που δεν έχουμε κάποιο άλλο σπίτι να πάμε, για όλους αυτούς λοιπόν τους πολίτες υπάρχει απώλεια δικαιωμάτων και δεν υπάρχει και προστασία. Η σενιόρ Ντάνς. Ο κύριος Ντάνς. Συμφωνώ με όλα όσα υπόθηκαν μέχρι στιγμής. Έχουμε μια ευρεία συνένεση, διακομματική. Δεν βλέπω κανέναν από τους συναδέλφους που στηρίζουν τον Brexit εδώ και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν θέλουν να ακούσουν τις αναφορές που παρουσιάζονται. Το, το επιχείρημα όμως που παρουσιάζουμε για την προστασία των δικαιωμάτων, για την προάσπιση του ιδανικού των Ευρωπαίων πολιτών δεν είναι κάτι στιγμιαίο. Είναι κάτι το οποίο στηρίζουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ήδη από το 2017. Ο κύριος Βερχόφστα είπε ότι θα εξετάσει την πιθανότητα του ring fencing, της προστασίας και της ενδυνάμωσης. Οι περιορισμοί του μοντέλου του, του κράτους μέλους και τα δικαιώματα των πολιτών που προκύπτουν ως τρίτοι πολίτες. Τα καταλαβαίνω όλα αυτά και βεβαίως εκτιμώ τους περιορισμούς. Παρόλα αυτά όμως πιστεύω ότι πρέπει να δώσει ένα ισχυρό σήμα το Κοινοβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τα άτομα που βρίσκονται εδώ σήμερα είναι άτομα που ήταν ήδη εδώ το 2017. Είναι άτομα που εξακολουθούν να, να ζουν την καθημερινή ζωή τους, ε, μπορεί να σπουδάζουν, μπορεί να έχουν αποφυτίσει, μπορεί να αγοράζουν σπίτια και να πρέπει να πληρώσουν υποθήκες. Ε, αυτά τα σημεία αναφορά στη ζωή του καθενός δεν μπορεί να μετακινηθεί. Παρ' όλα αυτά όμως η αβεβαιότητα εμένει και υπάρχουν άνθρωποι που στην καθημερινή τους ζωή δεν έχουν καταφέρει να βγουν από αυτό το στάδιο λίμπο στο οποίο βρίσκονται για ένα πραγματικά σύλληπτο χρονικό διάστημα. Υπάρχει ένα γενικό αίσθημα ότι θα μπορούσαμε να είχαμε δείξει περισσότερη αλληλεγγύη, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε στείλει ένα πολύ πιο ισχυρό ε, σήμα όπου η ευρωπαϊκή ηθαγένεια δεν προκύπτει μόνο από την γεωγραφία, από το που βρίσκεται κάποιος σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Δεν είναι μια πραγματικά παρουσία σε ένα συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αν σημαίνει κάτι παραπάνω, πράγμα για το οποίο έχετε παλέψει συνεπώς εδώ και πάρα πολύ καιρό, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προσπαθήσουμε να δώσουμε το στίγμα του τι σημαίνει να, να εγγράψουμε τους νόμους των πολιτών τρίτης χώρας για τις 27 χώρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχουν περιορισμοί και δυσκολίες. Δεν μπορώ όμως να σας πω πόσο φρικτό είναι για μια σειρά από πολίτες να αισθανθούν ότι τους έχουν αφήσει την τύχη τους, όχι μόνο οι χώρες τις οποίες ζουν, αλλά και αυτό το ίδιο το ιδανικό του πολίτη, το οποίο βρίσκονται σε μια κατάσταση όπου το, το στερούνται άνευ λόγω και αιτίας. Είναι πραγματικά ένα φρικτό πράγμα αυτό που συμβαίνει. Σας ευχαριστώ, λέει η πρόεδρος ο κύριος, η πρόεδρος ο κύριος Βερχοφστατ ή... αν θέλει να μιλήσει, θέλω να επιστρέψω, λέει ο κύριος Βερχοφστατ, σε κάποια σχόλια που έγιναν, αν μου επιτρέπετε. Το πρώτο είναι για την κυρία Τούμ. Αυτό που θα ζητούσα από τις υπηρεσίες θα ήταν να σας δώσουν μία σειρά από τις διμερείς συμφωνίες που εμείς τουλάχιστον έχουμε υπόψη μας, ως ε, κοινοβούλιο. Μια, μερά, μια ε, σειρά από τις α, διμερείς συμφωνίες αυτές έχουν ε, γίνει μεταξύ διαφόρων κρατών μελών. Μπορούμε να σας παρουσιάσουμε τις ε, διμερείς αυτές συμφωνίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιοι εκπρόσωποι του Brexit. Εδώ έχουμε και τη δική μας συνάντηση σε λίγη ώρα. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να θίξω είναι ότι υπάρχουν δύο διαφορετικά πράγματα. Το πρώτο, αν υπάρξει συμφωνία αποχώρησης, τότε ναι, πρόκειται να εφαρμόσουμε αυτό το πρόγραμμα εγκατάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, το Κοινοβούλιο θα πρέπει να πει, ναι, έχουμε ένα εργαλείο στα χέρια μας, πρέπει να εγκρίνουμε το πρόγραμμα αυτό εγκατάστασης και η δική μου ιδέα είναι ότι αν είναι να συμφωνήσουμε θέλω να είμαστε σαφείς στις συνθήκες υπό τις οποίες θα ισχύει. Άρα θα μπορέσουμε να επιστρέψουμε στο ζήτημα της αυτόματης εγγραφής, της δήλωσης ξένων πολιτών κτλ. Γιατί όντως, ναι, δεν είναι φυσιολογικό ε, για μια σειρά από πολίτες που έχουν κάνει αίτηση εγκατάστασης και έχουν λάβει την άδεια για κάποιους που θεωρούνται pre-settled, ήδη προεπιλεγμένοι. Δηλαδή, εγώ προσωπικά έχω ακούσει μια σειρά από παραδείγματα ατόμων που ζουν ε, σε μια χώρα 10 χρόνια και περισσότερο, στη Βρετανία, για παράδειγμα. Επομένως, μπορεί να θεωρηθούν pre-settlers. Αυτοί οι άνθρωποι είναι εγκατεστημένοι εκεί. Θα επιστρέψουμε, λοιπόν, άπαξ και έχουμε μία συμφωνία αποχώρησης μεταξύ των διαπραγματευόμενων μερών. Θα υπάρξει μια μεταβατική περίοδος και σε αυτή τη μεταβατική περίοδο ακριβώς αυτά τα πράγματα θα κάνουμε. Θα τη χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε ότι οι Βρετανικές αρχές θα εφαρμόσουν με τρόπο σαφή και σοβαρό όλη αυτή την ε, δήλωση εγκατεστημένων, την αυτόματη εγγραφή κτλ. Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Αυτό όμως άπαξε και υπάρξει μια συμφωνία. Αν έχουμε σκληρό Brexit, αν έχουμε no deal, δεν θα ξαναπώ τα ίδια που είπα και πριν, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι δύο πράγματα τα οποία θα πρέπει να εξασφαλίσουμε που πηγαίνουν ε, επί της ουσίας πέρα από τις ε, μονομερείς δεσμεύσεις εκ μέρους μας στους Βρετανούς πολίτες, στις Βρετανικές αρχές, ε, στους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι ένα νομοθετικό σύστημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά. Όπως βλέπουμε και στις επιμέρους συμφωνίες αυτό κατ' εμέ είναι ουσιώδες. Είναι κάτι το οποίο δεν είναι πέρα από αυτό που εγώ τουλάχιστον αποκαλώ μονομερή δέσμευση. Εμείς λοιπόν ως steering group θα θέσουμε επιτάπητος και πάλι στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα αυτό. Να πούμε ότι δεν υπάρχει επίσημα ring fencing, αλλά πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα. Και υπάρχει ένα δεύτερο σημείο, σας το είπα από την αρχή, το δεύτερο σημείο είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μονομερής αλλαγή στο σύστημα μετέπειτα. Αυτά είναι τα δύο σημεία, θεωρώ, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ως steering group. Αυτό θα πρέπει οι συνάδελφοι να, να θέσουν υποδιαπραγμάτευση. Να πούμε πώς θα εξασφαλίσουμε όλα αυτά που θέλουμε. Ότι υπάρχει νομοθετική κάλυψη και ότι υπάρχει και η βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει μονομερής ε, αλλαγή, περιορισμός των δικαιωμάτων αυτών. Ότι δεν θα είναι δυνατόν στην Συμφωνία Αποχώρηση. Αυτά είναι τα δύο σημεία που εγώ ήθελα, στα οποία ήθελα να αναφερθώ. Και θα ήταν ίσως σκόπιμο ίσως με την Επιτροπή ΠΕΤΗ, ίσως με τη Λίμπε, ίσως με την ΑΦΚΟ να επιστρέψουμε στο θέμα αυτό, γιατί για μένα είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. Αυτά ήθελα να πω. Ευχαριστούμε, λέει η Πρόεδρος. στον διευθυντή της ομάδας για τον Brexit. Είμαι σίγουρη ότι θα σας ξαναδούμε. Είτε σε άλλες επιτροπές, είτε και σε αυτήν εδώ την επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ γιατί ξέρω ότι έχετε σε... και τη δική σας ε, συνεδρίαση σε... στις 5.30. Και το επόμενο σημείο της σημερινής διάταξής μας είναι όλες οι αναφορές για τον Brexit. Θέλω να, να προσθέσω κάτι σε σχέση με αυτό που είπε ο Κλοντ, ότι υπάρχει μια τεράστια μετρήσιμη αλλαγή στη συμπεριφορά των πολιτών. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση σταδιακά χάνει την αιτία ύπαρξή της, ίσως όχι και τόσο σταδιακά. Επομένως, το τι μπορεί να είναι αποδεκτό για την κυβέρνηση. Και όλη αυτή η αβεβαιότητα μπορεί να είναι κάτι το οποίο διαρκώς εντείνεται. Παρόλο θα συμφωνώ με όλα όσα είπε ο Γκί και είμαι σίγουρη ότι μιλάω και εκ μέρους των συναδέλφων της ομάδας για το Brexit. Η πόρτα μας είναι ανοιχτή αν λοιπόν υποπέσει την αντίληψή σα το οτιδήποτε που θεωρείτε εσεί ότι εμεί πρέπει να ξέρουμε ή ότι θα πρέπει να το περάσουμε στην ομάδα του Περνιέ ή <laughs> άμα βρείτε και λύση, λέει ο Γκίβερ Χόφστατ, πάρτε μα ένα τηλέφωνο να μα την πείτε και εμά. Να σας προσκαλέσουμε πρόεδρε στην επόμενη συνεδρία στη ΣΑΦΚΟ όπου θα γίνει μια ακρόαση με τους εκπροσώπους των Ευρωπαίων και Βρετανών πολιτών ακριβώς για το ίδιο πρόβλημα. Τώρα θα δούμε τι έγινε με την επιστολή που έστειλε ο κύριος Μπόρις Τζόνσον στον πρόεδρο της Κομισιόν, τον κύριο Γιούνκερ. Έκανε κάποια, κάποιες προτάσεις εναλλακτικές του backstop. Είναι λίγο πιο ελαστικά αυτά που προτείνει. Ε, δεν είναι σαφές όμως τι προτείνει. Για μας είναι πολύ σημαντικό να προσπίσουμε τα δικαιώματα των πολιτών. Και γι' αυτόν τον λόγο θα ήθελα να σας προσκαλέσω να συμμετάσχετε. Είναι μια κρόση ανοιχτή σε όλα τα μέλη της ΠΕΤΗ και κυρίως βέβαια στην Πρόεδρο. Ευχαριστώ κύριε Ταγιάννη εκ μέρους της Επιτροπής 5. Προφανώς θα αποστείλουμε μια αντιπροσωπεία με μέλη μας. Σας θέλω να σας συγχαρώ για την εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η διευθυντική ομάδα, η διευθύνουσα ομάδα ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όλους αυτούς τους μήνες ε, διότι πραγματικά είχατε πάντοτε στο μυαλό σας ε, τις πραγματικές ανησυχίες, τα πραγματικά προβλήματα των Ευρωπαίων πολιτών. ποτέ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα αμελήσει το καθήκον του σε σχέση με όλους και τον καθένα από τους Ευρωπαίους πολίτες. Συνεχίστε αυτή τη δουλειά που κάνετε. Εξαιρετική. Περνάμε στο σημείο 16. Συνεχίζουμε για τον Brexit. Διάφορες αναφορές. Ορισμένοι από τους ε, αναφέροντες είναι εδώ. 0307 του 17 της Φιώνα Γκότφρι, η 0470 του 17, η 0627 του 18, η 926 του 18, η 97 του 19 και η 826 του 19. Όλοι οι αναφέροντες είναι πολίτες που ανησυχούν με τον Brexit. Θα δώσουμε καταρχήν το λόγο στα μέλη της Επιτροπής. Καταρχήν θα δώσω βέβαια το λόγο στον κύριο Στόκ γιατί βιάζεται, αν μου επιτρέπετε. Και μετά θα δώσω το λόγο στις υπόλοιπες πολιτικές ομάδες ε, για να ολοκληρώσουμε με τους αναφέροντες. Thank you for admitting my petition and for giving me the opportunity. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου την ευκαιρία να μιλήσω αν λάβει χώρα το Brexit, οι Βρετανοί πολίτες θα χάσουν την ευρωπαϊκή τους ηθαγένεια. Για πολλούς αυτό έρχεται σε αντίθεση με τις επιθυμίες τους. Κάτι παρόμοιο ε, θα προκαλούσε αγανάκτηση αν συνέβαινε αλλού στον κόσμο. Θα πρέπει να βρούμε λύσεις για τους ε, πολίτες που εκατέρωθεν ζουν σε, στην αντίθετη περιοχή. Θα πρέπει να εξασφαλιστούν το, τα δικαιώματα διαμονής και εργασίας των Ευρωπαίων πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνεται η υποστήριξη του, της ε, παραμονής. Αυτό είναι αποτέλεσμα της ανησυχίας πολλών. Πολλοί νιώθουν να τους κλέβει η ίδια τους η κυβέρνηση την ταυτότητά τους. και πολιτιστικά και πρακτικά και συναισθηματικά τα δικαιώματα μας θα περιοριστούν. Έχω δει τη μεγάλη αγωνία. Με τα δικά μου μάτια, ιδιαίτερα σε εμά στην Ιρλανδία, που έχουμε λίγο διαφορετική γεωγραφία και ιστορία από την υπόλοιπη Ευρώπη. Όλο αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό να βλέπουμε, να κοιτάμε του άλλου Ευρωπαίου στα μάτια και να του δηλώνουμε ότι είμαστε και εμεί τμήμα του ευρωπαϊκού project. Για τη λύση αυτού του είναι σαφέ ότι η δική μα κυβέρνηση δεν έχει προτείνει τίποτα το ουσιαστικό τα τελευταία τρία χρόνια. Είμαστε αόρατοι. Η καθημερινή ρητορική για τη θέληση του λαού δεν έχει καμία σχέση με τι δικέ μα επιθυμίες. Όπω είπε κάποιο, μα έχουν διαγράψει το ίδιο μα το μέλλον. Με άλλα λόγια, η Βρετανική κυβέρνηση δεν ξέρει τι να μα κάνει. Είναι προφανέ ότι και η καινούργια κυβέρνηση ενδιαφέρεται ακόμα λιγότερο από την προηγούμενη. Είναι επίσης σαφές ότι οι Βρετανοί που είναι υπέρ του Brexit επίσης δεν ενδιαφέρονται για μας. Για αυτούς είναι μια νίκη χωρίς αρνητικές πτυχές. Εγώ ζω στην εκλογική περιφέρεια του Υπουργείου, Εσωτερικών, του Υπουργού Εσωτερικών και βλέπω το μίσος που πολλοί από αυτούς που είναι υπέρ του Brexit εκφράζουν εναντίον μας. Όμως ε, δεν θα έπρεπε να πληγεί η ζωή των πολιτών της, του Ηνωμένου Βασιλείου από τον Brexit. Όμως αυτό θα συμβεί εξαιτία των δρατοπράξεων μιας μειοψηφία. Δεν θα έπρεπε η ευρωπαϊκή κοινότητα, κοινότητα των Ευρωπαίων να το δεχτεί αυτό. Ακόμα και αν συμβεί το Brexit και το Ηνωμένο Βασίλειο γίνει τρίτη χώρα, δεν θα έπρεπε να ε, αναγνωριστεί η μείωση των δικαιωμάτων. Θα έπρεπε η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσει ένα ειδικό καθεστώς που θα περιλαμβάνει ακριβώς τους Βρετανούς πολίτες που θα ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα τους δίνει σχεδόν πλήρη αν όχι πλήρη δικαιώματα σαν να ήταν Ευρωπαίοι πολίτες. Γι' αυτό το λέω πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό. Δεν θα πρέπει να πληγούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών ούτε στην Βρετανία ούτε το αντίστροφο, αλλά αυτό μπορεί να γίνει και μονομερός εν ανάγκη. Αν η Βρετανία δεν θέλει να πράξει το ίδιο. Ε, θα ήθελα ένα σύστημα τέτοιου τύπου να μην ε, πλήξει τους Βρετανούς που έχουν χαμηλά εισοδήματα, οπότε δεν θα πρέπει να, είναι, ε, να έχει ψηλό κόστος. Όλες αυτές οι διαδικασίες δεν έχουν καμία σχέση με την κυβέρνηση του Βρετανίου, της Μεγάλης Βρετανίας. Ε, Εγώ έχω δουλέψει στο εκπαιδευτικό σύστημα στη Βρετανία και σας λέω ότι ένα τέτοιο σύστημα θα είναι σημαντικό γιατί πραγματικά θα βοηθήσει πάρα πολύ να διατηρηθεί η συνείδηση των Βρετανών και η ταυτότητά τους. Ε, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαμε να συμφιλιώσουμε στο μέλλον τους Βετανούς ε, πολίτες με την υπόλοιπη Ευρώπη και να αποφύγουμε μια διολίσθηση της ε, κοινωνίας μας. Κάτι τέτοιο θα ενθάρρυνε τον μέρ Βασίλειο να ξαναενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Thank Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα η Τζέιν Κόλτι από το ε, British Europe δεν είναι εδώ και η κυρία Κίτον θα μας διαβάσει την παρέμβασή της. Ευχαριστώ πολύ. Θα κάνω μια δήλωση εκ μέρους του British in Europe των 1,2 εκατομμυρίων Βρετανών που ζουν στην Ευρώπη. Τρία εκατομμύρια είναι οι Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι δύσκολο να πιστέψει κανείς ότι η θέση αυτών των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται σε βεβαιότητα εδώ και τρία χρόνια θα μπορούσε να είναι ακόμα πιο αβέβαιη από την τελευταία φορά που είχαμε έρθει στην Επιτροπή σας τον Ιανουάριο. 30 μέρες μέχρι τις 31 Οκτωβρίου απομένουν και είμαστε στην, στα πρόθυρα μιας συνταγματικής κρίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρουμε καν ποια είναι η συμφωνία που ζητά το, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου. Δεν, αν δεν υπάρχει συμφωνία θα είναι μια καταστροφή. Θα έχουμε 29 μονομερείς ε, συμφωνίες ε, για θέματα όπως η κοινωνική ασφάλεια, η υγειονομική περίθαλψη, η αναγνώριση των προσόντων, που είναι ζωτική σημασία. Πρέπει να πάμε στην αρχή, να δούμε τι είχαν υποσχεθεί στους πολίτες τον Μάιο του 2017. Μισελ Μπαρνιά είπε στη Φλωρεντία και αναφέρω το επίπεδο της προστασίας που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία δεν πρέπει να φθήνει το Brexit δεν πρέπει να αλλάξει την καθημερινή ζωή των πολιτών. Τέλος της παράθεσης, οι βασικές αρχές ε, για τα δικαιώματα των πολιτών ε, το 2007 έλεγε ότι θα πρέπει να προστατευτούν ε, οι πολίτες του Ηνωμένου Βασιλείου και η οικογένειά τους που είχαν δικαιώματα ελεύθερης κίνησης την ημέρα που μπήκε σε εφαρμογή η αποχώρηση από το, του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων όλα αυτά δεν τηρήθηκαν και έγιναν παραχωρήσεις. Υπάρχουν ε, κάποιες ε, προστασίες ε, που δεν, βάζουν, δεν προστατεύουν ούτε καν τα βασικά δικαιώματα της διαβίωσης. Υπάρχουν επιλογές ζωής που έχουν γίνει με βάση τα δικαιώματα και όχι το ανάποδο. Δεν πρέπει λοιπόν να προστατέψουμε το lifestyle αλλά τα δικαιώματα. Όταν δεν υπάρξει συμφωνία, αυτά τα δικαιώματα που είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα προστατεύσει θα χαθούν στον αέρα και θα έχουμε όλα αυτά τα εκατομμύρια πολιτών που είχαν ασκήσει τα δικαιώματα ελεύθερης κίνησης ε, που θα πρέπει μέσα σε μια νύχτα να επανέλθουν ε, στην ε, πρώτερη κατάσταση χωρίς προστασία του προηγούμενου καθεστώτος τους. Δεν πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας τις προσδοκίες των πολιτών αυτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά διλήμματα. Οι πεπισμένοι Ευρωπαίοι που έχουν ασκήσει και ενεργοποιήσει τα δικαιώματά τους ως Ευρωπαίοι πολίτες τώρα αντιμετωπίζονται με τρόπο ε, περίεργο γιατί δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ηθαγένεια. Ε, είναι περίεργο το πώς αντιμετωπίζεται η ηθαγένεια αυτή. Επίσης υπάρχει κυριότητα της εσωτερικής αγοράς που, που εξετάζεται. Ποιο είναι όμως το νόημα να προστατεύει αυτό το, η Ευρωπαϊκή Ένωση αν δεν προστατεύει την απτή άσκηση της ε, ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το καθήκον να προστατέψει τους πολίτες της. Είναι πολύ σημαντικό για τα 3,6 εκατομμύρια πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σύντομα μπορεί να ζουν σε τρίτη χώρα. Ακόμα και αν ε, ήταν τέλεια η διαδικασία εγκατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο και 3 εκατομμύρια μας λέει ότι δεν είναι. Οι άνθρωποι αυτοί θα χρειάζονταν την προστασία μιας διεθνούς συνθήκης. Χωρίς αυτή την προστασία τα δικαιώματά τους μπορούν να ε, φύνουν με τον καιρό και σιγά σιγά χάνονται τα δικαιώματα αυτά ε, σε και, και κλεισμένων το θυρών με το δευτερογενές δίκαιο της του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς διεθνή συνθήκη να προστατεύει τα 3 εκατομμύρια, τα δικαιώματά του σίγουρα θα μειωθούν από αυτή την κυβέρνηση. Είμαστε λοιπόν στο άγνωστο. Θα έχουμε 27 διαφορετικές λύσεις. Το καθεστώς ε, θα βασίζεται ε, το πού θα ζουν ε, οι Βρετανοί πολίτες που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα υπάρχει μια ενιαία λύση για όλους. Και για τις δύο ομάδες, μια τη διεθνή συνθήκη, τα σημαντικά αμοιβαία ζητήματα όπως οι συντάξει, η υγειονομική περίθαλψη, τα επαγγελματικά προσόντα, απλώς δεν θα καλύπτονται. Ούτε θα υπάρχει ε, τήρηση των αρχών της ε, έλλειψης διακρίσεων και της ίσης μεταχείρισης. Δεν ξέρουμε καν τι θα συμβεί μετά την 31η Οκτωβρίου ή πριν από αυτήν. Αν συμφωνηθεί κάτι, θα πρέπει να υπάρξει μια δέσμευση ότι θα υπάρξει το ring fencing με το που θα ξεκινήσει η επέκταση. Συχνά ε, μας λένε ότι το ring fencing είναι δυνατό μόνο την τελευταία στιγμή. Όμως δεν είναι γιατί και το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βρετανία θα πρέπει να συμφωνήσουν σε αυτό, να τα κυρώσουν τα κοινοβούλια και να υπάρχει και μια νομοθεσία που θα περάσει από το Κοινοβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου πριν την ημερομηνία εξόδου. Και δεν μπορεί να γίνει υπό το άρθρο 50 γιατί θα προκύψουν θέματα αρμοδιότητας και η κύρωση από τα 27 κοινοβούλια συν τα περιφερειακά κοινοβούλια θα απαιτείται. Αντί για Γι' αυτό λοιπόν πρέπει άμεσα να αποφασίσουμε το ring fencing πριν μόλις δοθεί η επέκταση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει μια χαλαρο, μια ηρεμία όταν ε, οι νομοθέτες δουλεύουν τα κείμενα. Στην Βρετανία υπάρχουν 3 εκατομμύρια πολίτες. Δεν ζητούν κάποια επαναδιαπραγμάτευση, ζητούν αυτό που έχει ήδη συμφωνηθεί να διατηρηθεί και όχι να χαθεί πρέπει να προστατεύσετε 5 εκατομμύρια από τους πιο αφοσιωμένους πολίτες σας. Τα δικαιώματα τους δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν υποβληθεί σε παζάρια ή στο τίποτα δεν είναι συμφωνημένο μέχρι να συμφωνηθεί. Υπάρχει αυτό το καθήκον φροντίδας που η Ευρωπαϊκή Ένωση αφήνει στους πολίτες της. Μην αφήσετε 5 εκατομμύρια ανθρώπους από τα 17 εκατομμύρια να απογοητευτούν λόγω αυτής της άνευ προηγωμένου κατάστασης. Τώρα δεν είναι η ώρα να υποσκάψουμε τις πεπιθήσεις. Έχουμε τους πιο αφοσιωμένους πολίτες. Δηλώνω το δικό μου ενδιαφέρον. Έχω Βέλγο σύζυγο, παιδί με τον Βέλγο σύζυγό μου και είμαι εδώ για να υπερασπιστώ τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων που ε, είναι στην ίδια θέση με μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για αυτή την συναισθηματικότατη έκκληση για όλους εμάς που πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τώρα ο Άντωνι Βάλκερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου για την εκλογή τους και σας ευχαριστώ που με προσκαλέσατε σε αυτήν εδώ την ακρόαση σήμερα. Μαζί με την συνάδελφό μου σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μία σειρά από αναφορές, μία από τις οποίες σχετίζεται με την ανεπάρκεια δυστυχώς της προστασίας που προβλέπεται στη Συμφωνία Αποχώρησης. Το περιεχόμενο της Συμφωνίας Υποχώρησης, Αποχώρησης, με συγχωρείτε, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, δυστυχώς δεν στέκεται στο ύψος των αιτήσεων, των απαιτήσεων των Ευρωπαίων πολιτών. Αυτό που θέλουμε λοιπόν είναι την προστασία των δικαιωμάτων και όσων ορίζονται στο πρωτογενές δίκαιο το δικαίωμα, έτσι όπως θα έπρεπε να ορίζεται σε μια συμφωνία αποχώρησης, θα έπρεπε να ορίζει το ίδιο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων, έτσι ακριβώς όπως περιγράφεται στο πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς όμως το περιεχόμενο της συμφωνίας αποχώρησης δεν ανταποκρίνεται σε αυτούς τους στόχους και πιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά το άρθρο 50 της Επιτροπής. Θα πρέπει να εξηγήσει αυτήν εδώ την ομάδα για ποιο λόγο υπάρχουν αυτά τα κενά και ποια είναι τα κενά αυτά. Πρώτα απ' όλα σε ό,τι αφορά τα παιδιά. Όλοι γνωρίζετε την απόφαση Ζαμπρούλινγκ του α, Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παιδιά Βρετανοί που γεννιούνται από μη Ευρωπαίους γονείς θα έχουν το δικαίωμα παραμονής και το δικαίωμα ηθαγένειας ή γονεί στη χώρα των παιδιών. Δυστυχώς δεν υπάρχει, δεν εξασφαλίζεται η προστασία αυτή στη συμφωνία αποχώρησης που να εξασφαλίζει ότι το άτομο που φροντίζει τα παιδιά θα μπορεί να παραμείνει στη χώρα. Και αυτό είναι κάτι που θα μπορούσε ενδεχομένως να επηρεάσει δεκάδες χιλιάδες παιδιά στη Βρετανία, αν όχι περισσότερα. Αν το σκεφτούμε, το 2017 περίπου 200.000 παιδιά γεννήθηκαν στη Βρετανία από έναν τουλάχιστον πατέρα που δεν ήταν Βρετανός υπήκος. Ένα άλλο κενό σε ό,τι αφορά τους Βρετανούς που επιστρέφουν στη χώρα τους μετά από την εξάσκηση του ελεύθερου δικαιώματός τους για την μετακίνηση δεν υπάρχει προστασία των δικαιωμάτων τους, να εξασφαλίσει ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες που επιστρέφουν στη χώρα τους έχοντας ζήσει σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν μπορούν να επιστρέψουν μαζί με ε, συνοδευόμενοι από ένα μη Βρετανό πολίτη, μέλος άλλης χώρας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε ό,τι αφορά τώρα την κατάσταση των Βρετανών πολιτών, δεν θα έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης μετακίνησης θα είναι περιορισμένοι στη χώρα διαμονής τους τη στιγμή που θα γίνει το Brexit. Επίσης δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις σε ό,τι αφορά τις εξουσίες που θα έχει η ανεξάρτητη αρχή που θα πρέπει να εγκατασταθεί στο Ηνωμένο Βασίλειο για να εξασφαλίσει ότι εφαρμόζονται οι περιορισμοί και οι κανόνες της συμφωνίας της αποχώρησης. Για παράδειγμα, το δικαίωμα παρέμβασης εκεί όπου δεν παρέχονται, δεν παράγονται αποφάσεις. Υπάρχει γίνει, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση σε ό,τι αφορά αυτήν την ανεξάρτητη αρμόδια αρχή. Πολλά από τα μέλη του κοινοβουλίου αυτού και πολλές περισσότερες φορές έχουν αναφερθεί στο γεγονός των λεγόμενων settled staters, των ατόμων που θεωρούνται εγκατεστημένοι σε μια χώρα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι ήταν η ίδια επιτροπή που α έθιξε αυτό το θέμα στις διαπραγματεύσεις με τις αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, της εγκατάστασης, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Εγκατάστασης. Το να αλλάξουμε λοιπόν το σύστημα αυτό, το πρόγραμμα εγκατάστασης σε μια αυτόματη εγγραφή, πάνω να πει ότι θα πρέπει να επανεκκινήσουμε τις διαπραγματεύσεις και αυτό είναι κάπως ληστηρό έδαφος για να, να δουλέψουμε. Θα ήταν πολύ καλύτερα να υποχρεώσουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να αποσύρει την προθεσμία για την εγγραφή στο πρόγραμμα αυτό εγκατάστασης, γιατί με αυτό τον τρόπο θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι θα αντιμετωπίσουμε το ζήτημα αυτό εγκατάστασης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ένα τελευταίο σημείο. Ο πρόεδρος του steering group ο Γκίβερ έκανε λόγο για ένα σκληρό ή πιο ήπιο Brexit. Αυτοί όμως που θα υποφέρουν περισσότερο αν δεν εξασφαλίσουμε τον ring fencing, το ring fencing των δικαιωμάτων θα είναι οι Βρετανοί πολίτες. Οι Βρετανοί πολίτες θα πρέπει να αντιμετωπίσουν 27 διαφορετικές νομοθεσίες που θα ποικίλουν από καμία απολύτως αλλαγή όπως συμβαίνει στην Ιρλανδία, και από τεράστιες αλλαγές όπως συμβαίνει στην Ιταλία αλλά και σε πολύ πραγματικά ε, περιοριστικές νομοθεσίες όπως ε, θα συμβεί στο Βέλγιο. Μέχρι το τέλος προθεσμίας ξέρουμε τι, τι πρόκειται να γίνει εδώ μετά, κανείς δεν ξέρει τι πρόκειται να συμβεί. Επομένως, θα πρέπει να σκεφτούμε πάρα πολύ σοβαρά να υιοθετήσουμε ένα μονομερές όργανο που να εξασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, των Βρετανών πολιτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας και λυπάμαι που καταχράστηκα το χρόνο Ευχαριστώ. Ο λόγος στην Λούσι Ναβίγιο. Λουσίνα Ναμπιζού. Δεν είναι εδώ. Εδώ είναι. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσω που δίνετε την ευκαιρία στη Haringey Welcome Organization, την οποία εκπροσωπώ, να σας παρουσιάσει την αναφορά μας. Εισαγωγικά, θα ήθελα να σας περιγράψω εν συντομία ποιοι είμαστε. Τις ανησυχίες μας επίσης για τα δικαιώματα των ε, μεταναστών και των ετουμένων ασύλου στο Ηνωμένο Βασίλειο και το πώς μπορεί το Κοινοβούλιο να βοηθήσει. Η Χάριγκεϊ ε, έχει έδρα στο βόρειο, ε, είναι μια περιοχή στο βόρειο Λονδίνο με πολλούς αλλοδαπούς από τα τέσσερα σημεία του πλανήτη. Από, μερικοί από αυτούς είναι από τους πιο φτωχούς στην, στην Ευρωπαϊκή, στην, στο Βασίλειο. Η Hurricane Welcome είναι ένα, μια ομάδα που, ανθρώπων που ζουν εκεί. Ξεκινήσαμε το 2015 με την εκστρατεία να πείσουμε τις ε, τοπικές αρχές να επανακαταστήσουν στην κοινότητά μας οικογένειες ε, σύρων ε, μεταναστών και προσφύγων. Προσπαθούμε να διαμορφώσουμε τοπικές υπηρεσίες και τοπικές πολιτικές πιο φιλικές προς τους πρόσφυγες και ιδιαίτερα να βοηθήσουμε τους πιο φτωχούς από τους συμπολίτες μας. Επίση, ε, κάνουμε εκστρατεία για να σταματήσουμε αυτό που η Βρετανική κυβέρνηση ε, δημιουργεί και που είναι ένα εχθρικό περιβάλλον, ένα σύνολο πολιτικών, αρνητικών πολιτικών που δημιούργησαν ένα ε, ολόκληρο σύστημα εσωτερικών συνόρων με συλλήψεις και επαναπατρισμούς ατόμων που δεν έχουν χαρτιά. Ε, όλα αυτά ξεκίνησαν το 2012 ε, με υπουργό εσωτερικών Τερέζα Μέη και ε, κατέληξαν σε βάρβαρη εκδίωξη και συμπεριφορά σε άτομα τα οποία είναι από το, προέρχονταν από το Commonwealth και δεν ήταν Βρετανοί. δεν του ε, κατέσχανε του τους του αρνούνταν να του χορηγήσουν άδειε οδήγηση, στέγαση κλπ. Πολύ συχνά πολλοί από αυτούς ε, ε, συνελήφθησαν, έμειναν σε καταβλισμούς και στρατόπεδα και μετά εκδιώχθηκαν από τη χώρα μας. Πολλοί από αυτούς έχανε και τη ζωή τους. Όλο αυτό το σύστημα δεν έχει καταργηθεί παρόλε τι ε, αντιρρήσει που έχουν εκφραστεί. Το, η Βρετανία δεν μπορεί λοιπόν να προστατεύσει ούτε καν τα δικαιώματα των δικών τη πολιτών. Πολίτε που είναι ακόμα Ευρωπαίοι πολίτε. Με το Brexit να είναι ε, πρώτον πυλών, έχουμε σημαντικέ ανησυχίε ε, για την ενδεχόμενη διεύρυνση αυτού του καθεστώτο και ε, για στους ε, Ευρωπαίους μη Βρετανούς μόνιμους κατοίκους του Ηνωμένου Βασιλείου. Ε, οι, αυτοί οι άνθρωποι δεν έλαβαν αυτόματα το καθεστώς ε, της εγκατάστασης και δεν υπάρχει κανένα σύστημα που να βοηθάει ε, τους, ε, αυτούς που είναι οι πιο απομονωμένοι στο να αποκτήσουν πρόσβαση στο μηχανισμό χορήγησης αυτού του καθεστώτος. Οπότε ορισμένοι από αυτούς τους Ευρωπαίους πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορεί να πέσουν στην κατάσταση που αντιμετώπισαν αυτοί οι πολίτες του Commonwealth ε, για τις οποίες σας μιλούσα προηγουμένως. Μετά τον Brexit, από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου δεν σκοπεύει ε, να ε, επιτελέσει το, να τηρήσει τις υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που βρίσκονται στο έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ό,τι αφορά την επανένωση των οικογενειών. Έχει πει ότι μετά το Brexit δεν θα επιτρέψει επανένωση οικογενειών σε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο, ούτε καν για παιδιά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συγγενείς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτές οι οικογένειες θα έπρεπε να μπορούν να επανενωθούν και να παραμείνουν, να διαμείνουν μαζί στο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit μέσω χορήγησης θεωρήσεων και συγκεκριμένων διαδικασιών επανένωσης. Ε, η, το η κυβέρνηση λοιπόν του Ηνωμένου Βασιλείου προ, προτιμά να αγνοήσει τις υποχρεώσεις της ε, και την προστασία των δικαιωμάτων που έχουν καταγραφεί στην, ως θεμελιώδη δικαιώματα για τους ε, ε Βρετανούς πολίτες. Το Ηνωμένο Βασίλειο όμως είναι ακόμα πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνεπώς με αυτόν τον τρόπο παραβαίνει το πρωτογενές δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συνεπώς Παροτρύνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να λάβει μέτρα έτσι ώστε να εξασφαλίσει την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τα οποία έχουν χορηγηθεί σε όλους τους πολίτες ε, και τα οποία η Βρετανική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή δεν προστατεύει. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα μπορούσαμε να συγκεντρώσουμε τα σχόλιά μας σε μια παρέμβαση κομισιόν. Πέστε μου εσείς ποιος από τους τρεις θέλει να πάρει το λόγο, αλλά ένας από τους τρεις παρακαλώ. Στέφαν Τερέκ. Εκπροσωπώ την ομάδα του Μισελ Μπαρνιέ. Έχουμε και άλλους ανθρώπους από την Κομισιόν, από την DG Δικαιοσύνης και DG Εσωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστώ πολύ τους ε, ε, αναφέροντες για το πάθος τους, για τον ενθουσιασμό τους, για το συναισθηματισμό τους. Καταλαβαίνω την αγωνία, καταλαβαίνω το, τη συναισθηματική φόρτιση. Κανένας δεν είναι εδώ ε, από επιλογή. Θα θέλαμε να, είχα, να είχε ρυθμιστεί το Brexit πιο νωρί. Δυστυχώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Στο προηγούμενο σημείο τη μέση διάταξη, ο Γκίφ Βερχόφστατ είπε ότι, έχουμε, ότι Κοινοβούλιο και Κομισιόν συνεργάστηκαν πάρα πολύ στενά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Σε τρία τέταρτα περίπου ο Μισελ Μπαρνιέ θα συναντηθεί με την ομάδα, με τη διευθύνουσα ομάδα και θα συζητήσει και το θέμα αυτό. Ε, Καθώ επίση και το θέμα τη Ιρλανδίας και τη Βόρειας Ιρλανδίας, όπου η κατάσταση του Brexit δημιουργεί ιδιαίτερη αγωνία για του πολίτε. Ε, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την εφαρμογή τη ε, συμφωνία μεγάλη παρασκευή που αποτελεί και τμήμα τη συμφωνία απόχώρηση στην οποία αναφέρθηκε ο Βερχόφστατ προηγουμένω. Ο κ. Βερχόφστατ είπε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έσπρωξε την Κομισιόν προκειμένου να δώσει, δικαιώματα, ε, να δώσει προτεραιότητα στα δικαιώματα των πολιτών. Μα άρεσε αυτό. Πρόκειται για 3 εκατομμύρια Βρετανών στην Ευρώπη, με αντιπροσώπους των οποίων συναντηθήκαμε επανειλημμένως και ο κ. Μπαρνιέ και, το, και η ομάδα του. Πρέπει να προστατεύσουμε τις επιλογές ζωής ε, των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών των 27 χωρών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις ε, για την συμφωνία αποχώρησης με τις Βρετανικές Αρχές στην αρχή του 2018, ε, τα ουσιαστικά δικαιώματα, τον τρόπο άσκησής τους, ε, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα, τις διοικητικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της εφαρμογή. Εξασφαλίσαμε την απλότητα του συστήματος, συζητήσαμε τα θέματα του κόστους, και το πώς ε, το κόστος θα αποτελέσει άχθος κλπ. Τώρα, κάποιοι από τους αναφέροντες έδειξαν πολύ συγκεκριμένα ζητήματα, θα ήθελα να επανέλθω αυτά. Ένα σημείο το οποίο δεν συζητήθηκε ε, είναι η μελλοντική σχέση και η δήλωση για αυτήν. Συμφωνήσαμε με τη Βρετανική κυβέρνηση σε μια δήλωση για τη μελλοντική σχέση, η οποία θα καθοριστεί μετά από διαπραγματεύσει. Είναι σαφέ ότι η σημερινή Βρετανική κυβέρνηση θέλει να αλλάξει ε, την δήλωση αυτή του Νοεμβρίου ε, του 2018. Ε, σε κάθε περίπτωση όμως με την κυβέρνηση της Τερέζα Μέη είχαμε καταλήξει στο ότι η Βρετανία θέλει να σταματήσει την ελεύθερη κυκλοφορία. Δεν θα είναι λοιπόν δυνατόν οι Ευρωπαίοι πολίτες των 27 να κινούν, να ε, εισέρχονται στην στο Μεγάλη Βρετανία ελεύθερα. Και το αντίστροφο. Το ίδιο θα γίνει και με, γενικότερα και με την ενιαία εσωτερική αγορά και με, τις, ε, με την κυκλοφορία των αγαθών και των υπηρεσιών. Αυτό προφανώς επηρεάζει πάρα πολλά πράγματα σε ό,τι αφορά αυτά που είπαν οι αναφέροντες. Επηρεάζει την ελεύθερη κυκλοφορία και το, την ελεύθερη διαμονή ε, των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και την ελεύθερη επαγγελ, άσκηση επαγγελματο. Όλα αυτά θα πρέπει να βασίζονται στην αμοιβαιότητα και στην αρχή της ε, μη διάκρισης μεταξύ των 27 ε, όταν καθοριστεί το οριστικό καθεστώς. Ε, ο όρος περίκλειστος χρησιμοποιήθηκε από ένα από τους αναφέροντες, έχει δίκιο. Οι Ευρωπαίοι πολίτες έχουν πολύ συγκεκριμένα δικαιώματα. Υπάρχει ένα κεκτημένο λοιπόν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει και συγκεκριμένα δικαιώματα στους Βρετανούς πολίτες ως πολίτες τρίτων χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποιοι αναφέροντες αναφέρθηκαν σε αδυναμίες και κενά το σημειώνουμε. Γνωρίζουμε αυτές τις θέσεις γιατί έχουμε συζητήσει με πολλούς από αυτούς που είναι εδώ αλλά και εκτός της αιθούσης. Για παράδειγμα, ανησυχία σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Θαγένεια. Ε, η Συμφωνία Αποχώρησης εστιάζει στην ελευθερία, στα δικαιώματα κυκλοφορίας. Ε, ο κ. Στοκ αναφέρθηκε σε αυτό, δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά ε, αυτή τη στιγμή ο κανόνα είναι ότι πρέπει κανεί να είναι Ευρωπαίο πολίτη για να έχει ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. Αν πρέπει να το συζητήσουμε αυτό, θα μα το πει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. σω θέλετε να το δείτε εσεί και να το προτείνετε. Αν θέλουμε κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτό. Επίση, οι εθνικέ αρχέ μπορούν να επιβάλλουν συγκεκριμένε υποχρεώσει ε, σε ό,τι αφορά του πολίτε που ασκούν το δικαίωμα τη ελεύθερη κυκλοφορία ε, δεν θα προσθεθεί κάτι σε αυτό. Επίσης υπάρχει το δικαίωμα προστασίας στους Ευρωπαίους πολίτες οι οποίοι επιστρέφουν από τρίτη χώρα. Ε, υπάρχει ένα ισχυρό σύστημα εφαρμογής της ε, Συμφωνίας Αποχώρησης, το ανέφερε και ο Κίφερ Χόφστατ, άμεση εφαρμογή. Οπότε οποιοδήποτε μπορεί να προσφύγει στο δικαστήριο, βρετανικά δικαστήρια ή το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα υπάρχει και μια εθνική ανεξάρτητη αρχή που θα παίζει το ρόλο που παίζει η Κομισιόν ε, ως θεματοφύλακα δηλαδή της ε, συμφωνίας ε, αποχώρησης. Με τη συμφωνία αποχώρησης, η συμφωνία αποχώρησης έχει κλείσει τον Νοέμβριο του 2018 από το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο, δεν πρόκειται να ξανανοίξει η διαπραγματεύσή τη. Το μόνο το οποίο συζητάμε αυτή τη στιγμή με τη Βρετανία είναι η κατάσταση και το σύστημα που θα διέπει την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία. Προσπαθούμε να βρούμε μια νομικά διαχειρίσιμη και λειτουργική λύση για τον backstop. Τώρα, για το ring fencing, την περιχαράκωση, την προστασία των δικαιωμάτων, στην οποία αναφέρθηκαν πολλοί. Δεν είναι δική μας προσέγγιση να περιχαρακώσουμε τα δικαιώματα των πολιτών μέσω της Συμφωνίας Αποχώρησης. Σκεφτείτε τι θα γινόταν στην κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ο, Κίφερ ε, Χόφστατ ε, είπε ότι δεν θα δεχτούμε τον βομβαρδισμό από πολλές μικρές μήνυ συμφωνίες. Υπάρχει ένα ολόκληρο πακέτο δικαιωμάτων που έχουν σχέση με το τμήμα 5 της εφαρμογής της Συμφωνίας Αποχώρησης, ε, οπότε δεν είναι δυνατόν να διαλέξουμε ένα κομμάτι από αυτά και να τα βάλουμε σε μια, ε, στη Συμφωνία ε, του ring fencing. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ε, απαρνείται την Συμφωνία Αποχώρησης. Οτιδήποτε θα υπέσκαπτε ε, την Συμφωνία αυτή ε, δεν μπορεί να γίνει δεκτό. Υπάρχει μια σαφής πλειοψηφία στο Βρετανικό Κοινοβούλιο εναντίον της άτακτης εξόδου. Οπότε κάποια στιγμή θα πρέπει να γίνει μια ψηφοφορία για να ληφθεί απόφαση. Έφτακτο ή άτακτο Brexit. Εκτό και αν εντωμεταξύ έχουμε συμφωνήσει. Αλλά πάντως εμεί μέχρι τότε ε, θα πρέπει να επιμείνουμε και να σταθούμε πίσω από τη συμφωνία αποχώρηση που έχουμε ε, συνάψει, στην οποία έχουμε καταλήξει. Καταλαβαίνω την αγωνία σα, αλλά αυτό είναι ο μόνο τρόπο να είμαστε αποτελεσματικοί και να έχουμε αποτέλεσμα. Πρόεδρο. ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Παρακαλώ πολύ εν συντομία, γιατί έχουμε ακόμα τρεις αναφορές και στις 6.30 θα διακοπεί η διερμηνία. Δεν θα ήθελα οι αναφέροντες να μην έχουν το δικαίωμα να μιλήσουν τη γλώσσα τους. ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μιλήσω ουγγρικά. Νομίζω ότι Έχουμε ε, σε έτσι, έντονους συναισθηματικούς τόνους κάνει αυτή την ακρόαση. Όλοι όσοι ήρθαν εδώ με μία αναφορά έπρεπε να πάρουν τη διασφάλιση ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτή την αναφορά τους με τον υψίστο σεβασμό και επίσης είδαμε και την ε, απάντηση του Κίχη Φεροστάτ και των άλλων ευρωβουλευτών, οπότε από όλα όσα μας είπαν και από όσα μας είπε η Κομισιόν είναι κάτι που πραγματικά βγαίνει ως συμπέρασμα και είναι ξεκάθαρο. Ο Μισελ Μπαρνιά έχει προσφέρει πολλά στη συζήτηση και γενικά τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κάνει τα πάντα ώστε να αντιδράσουν σωστά στο Brexit, το οποίο σίγουρο, σίγουρα θα συμβεί. Και οι πολίτες βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Είναι απαράδεκτο να χάνουν οι πολίτες τα δικαιώματά τους. Όμως, από την πρώτη στιγμή προσπαθήσαμε να βρούμε λύσεις για τους πολίτες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο και τους Βρετανούς που ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή το Brexit θα γίνει ούτως ή άλλως, ε, πονάει περισσότερο. Και είναι δύσκολο ε, για μας, γιατί δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε και να δούμε πόσο καιρό θα διαρκέσουν όλα αυτά. Ο πόνος λοιπόν γίνεται ακόμα μεγαλύτερος. Εδώ στην Επιτροπή μας δεν μπορούμε να κάνουμε στην πραγματικότητα πολλά, μπορούμε απλώς να παρακολουθήσουμε αυτά που συμβαίνουν και μπορούμε να προωθήσουμε λύσεις οι οποίες είναι οι καλύτερες για τους πολίτες. Ε, το θέμα είναι να κρατήσουμε ανοιχτές ε, τις αναφορές, αυτό μπορούμε να κάνουμε εμείς, όμως ε, για την ε, συμφωνία χρειάζονται και οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μια επικοδομητική στάση. Τώρα πρέπει και το Ηνωμένο Βασίλειο να έρθει με μια καλή λύση ώστε να χάσουν όσο λιγότερα γίνεται οι πολίτες. Δεν θέλουμε λοιπόν περιπτώσεις περιπτώσεις ε, παραβίασης του δικαίου και δεν θέλουμε και περιπτώσεις ε, που μειώνονται τα δικαιώματα των πολιτών. Τις επόμενες εβδομάδες, λοιπόν, θα ακούσουμε πολλά για το Brexit και πραγματικά πονάει όταν κανείς ε, πρέπει να ασχοληθεί με τα δικαιώματα των πολιτών. Ο κύριος Ρουίντε Μέσα έχει το λόγο. Ευχαριστώ. άκουγα την διερμηνία. Ήθελα να την ακούσω μέχρι το τέλος. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τα σχόλια σας προηγουμένως. Ας πάμε τώρα στο θέμα που μας απασχολεί. Θα προσπαθήσω να μιλήσω τη γλώσσα των αναφερόντων. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για τη δέσμευσή σας και μια, ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ ε, στο Τζουτ Ντάρλινγκ που το έκανε προτεραιότητα και μου θύμισε το πόσο σημαντικό είναι να βρισκόμαστε σήμερα εδώ η κυρία Κέλλη μας ε, έδειξε και τη σημασία των σοσιαλδημοκρατών γιατί γίνατε ο εκπρόσωπος ε, ενός εκ των αναφερόντων. Αυτό που είπε ο πρόεδρος Μονσεράτε για την οικονομία και τη χρήση του χρόνου, εμείς εκ μέρους των σοσιαλδημοκρατών υποστηρίζουμε τους αναφέροντες και τις αναφορές ε, των Φιώνα ή Ιαν Σκότ, Άντωνη, Βάλκε και τη Μικαιόπικου Είναι πολύ σημαντικό διότι αυτή τη στιγμή βλέπουμε πως το Brexit ε, πλήττει ιδιαίτερα τους ανθρώπους που μας χρειάζονται περισσότερο στην κοινωνία. Τους μετανάστες ε, του ετούντες άσυλο. David Neville Smith και άλλος ένας αναφέρον που δεν βλέπω το όνομά του ήταν μεταξύ αυτών των αναφορών που ήρθαν σε εμά και που θεωρούμε ότι είναι ιδιαίτερα σχετικές ως προς την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα θέλαμε λοιπόν να παραμένουν ανοιχτές αυτές οι αναφορές και υποστενή παρακολούθηση και εποπτεία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να υποστηρίξω στεναρά τις αναφορές που ακούσαμε, ειδικά την αναφορά του Αντώνη Βάλκε και να σχετικά με την οικογένεια Ζαμπράνο. Να πω ότι αυτή μπορούσε να είναι η οικογένειά μου. Ο μόνος λόγος που δεν είναι, είναι ότι ήμουν αρκετά τυχερή και μπόρεσα να πληρώσω για το ε, διαβατήριο, βρετανικό διαβατήριο. Δεν είναι σωστό η Βρετανία να χρεώνει πέντε φορές παραπάνω από άλλες χώρες για ένα διαβατήριο. Πέντε φορές παραπάνω από το μέσο όρο όλων των 27 χωρών. Γιατί το κάνουν αυτό, γιατί δεν θέλουν αυτούς που δεν μπορούν να δώσουν ε, μεταξύ 1.500 και 1.700 Βρετανικών λιρών για το διαβατήριο. Αν δικαιούνται αυτό το διαβατήριο θα πρέπει να το πάρουν. Και πρέπει αυτό να το έχετε στο μυαλό σας όταν εξετάζετε την κατάσταση των Ευρωπαίων πολιτών στην ε, Βρετανία. Το κόστος της νομιμοποίησης είναι 250 με 300 ευρώ στην Ευρώπη και στις άλλες χώρες. Ε, αυτό το ποσό κατά μέσο όρο τηρείται. Νομίζω λοιπόν ότι καλό θα ήταν να έχουμε μια αμοιβαιότητα ως προς το κόστος του να γίνεις πλήρες μέλος ε, αυτής της ε, κοινωνίας και του δικαιώματος να μπορείς να ψηφίσεις στη χώρα που κατοικείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Μπανλόκα, η κυρία Μπανλόκα. Η κυρία Μπανλόκα. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω κι εγώ να στηρίξω τις αναφορές, ιδίως την κυρία Κύρτον που ήταν τόσο συναισθηματική Είμαι βαθύτατα ανήσυχη από τις αποφάσεις της ε, Κομισιόν, καθόλου ικανοποιημένη. Και θέλω λοιπόν να απευθυνθώ σε εσά. Αν εμείς πρέπει να αναλάβουμε τις ευθύνες μας και πρέπει να προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε με κάποιο τρόπο τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να βρεθούν οι διάφοροι πολίτες Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε εξετάσει διαφορετικές πιθανότητες. Από τότε που βρισκόμαστε σε αυτό το παράδοξο καθεστώς μη πολιτών. Και ξέρουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και να το προωθήσουμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο χωρίς να αλλάξουμε τις συνθήκες. Για παράδειγμα, η οδηγία αυτή για τους μόνιμους κατοίκους τρίτων χωρών που διαμένουν σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν κάποιος κατορθώσει να λάβει το καθεστώς στο κράτος μέλος όπου διαμένει, τότε μπορεί να μετακινηθεί σε άλλο κράτος μέλος. Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο σε μια σειρά από κράτη-μέλη, συμπεριλαμβανομένου και του δικού μου, να μπορέσουν να αποκτήσουν αυτό το καθεστώς. Έχουμε μόλις... Έχουμε λιγότερους από 200 κατοίκους, από 250.000 ξένους που, που ζουν εκεί, γιατί στην ίδια την οδηγία γράφεται, αναγράφεται ότι τα κράτη-μέλη μπορούν να βάλουν επιπλέον κριτήρια. Για παράδειγμα, καλή χρήση της γλώσσας. Γιατί αν θες να μετακινηθείς από το ένα στο άλλο κράτος μέλος, γιατί πρέπει να περάσει αυτές τις εξετάσεις γλώσσας Επομένως, η οδηγία αυτή δεν μ' αρέσει καθόλου εν ολίγης. Και πιστεύω ότι πρέπει να βελτιωθεί και η Κομισιόν μπορεί να το κάνει. Κάτι άλλο τώρα. Σας προτείνω να αναλογιστείτε το ακόλουθο. Είπα ότι δεν πιστεύω σε μονομερείς δεσμεύσεις. Αλλά στην περίπτωση της Λευκορωσίας πιστεύω ότι εφαρμόζουμε κάτι που θα μπορούσε να είναι και χρήσιμο και για το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλώσεις διευθύνσεως σε διάφορα κράτη-μέλη. Τι κάνουμε στη Λευκορωσία. Λετωνία, με συγχωρείτε. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε ίσως να κάνει κάτι ανάλογο. Μόνο και μόνο για να θεωρήσουμε ότι θα πρέπει οι πολίτες που ζουν, σε, οι Βρετανοί πολίτες που ζουν σε άλλα, σε άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να θεωρούνται ως μόνιμοι κάτοικοι. Θα πρέπει να θεωρούνται, να τους μεταχειρίζονται ως Ευρωπαίους πολίτες. Και κατά αναλογία, τα κράτη-μέλη αυτά μπορούν να ζητήσουν από το Ηνωμένο Βασίλειο να θεωρήσουν ότι οι πολίτες που έχουν μόνιμη διεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Ηνωμένου Βασιλείου. Υπάρχουν ε, βήματα που μπορούμε να κάνουμε. Αλλά εσείς ως υπεύθυνοι για τις αναφορές και εμείς ως πολιτικοί πρέπει να βάλουμε τα δυνατά μας για να μπορέσουμε να προωθήσουμε τέτοιου τύπου λύσεις. Αυτά είναι ένα-δύο παραδείγματα που σας έδωσα. Υπάρχουν όμως πάμπολες ενέργειες που μπορούμε να, να κάνουμε. Σας εύχομαι το καλύτερο δυνατό στην προσπάθειά σας και θα είμαστε ε, στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Για να κλείσουμε αυτό το θέμα, θα ήθελα να ζητήσω από τους αναφέροντες ε, εν συντομία να κάνουν κάποιες τελικές παρατηρήσεις. Ο λόγος του κύριου Άντωνη Βάλκια καταρχήν. Και μετά στον Άντωνη Βάλκε και στην Λούσινα Μπιζού. Εν συντομία όμως παρακαλώ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι ότι πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα ε, στην περίπτωση ανυπαρξίας συμφωνίας χωρίς ε, να απαρνηθούμε την ανάγκη μιας συμφωνίας νομικά. Ένα από τα πράγματα που μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο μερός είναι να υιοθετήσει ένα ενιαίο νομικό κείμενο που θα προστατεύει τα δικαιώματα των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση στην περίπτωση εξόδου χωρίς ε, συμφωνία και δεδομένου ότι θα είναι μονομερής αυτή η προσέγγιση θα παροτρύνει την Βρετανία να κάνει το ίδιο. Έτσι κι αλλιώς, είτε υπάρχει συμφωνία είτε δεν υπάρχει, θα πρέπει η Βρετανία να έχει ένα είδου καθεστώ για του πολίτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό ξεκίνησε ήδη από τον Απρίλιο του τρέχοντο έτου. Ε, κάποιο καθεστώ ε, δεν είναι αρκετό, δεν θα είναι πλήρε. Πάντω η ύπαρξη κάποιου καθεστώ είναι καλύτερη από τη μη ύπαρξη. Ακόμα και στην περίπτωση που λάβει η χώρα το Brexit. Και εγώ ακόμα ελπίζω ενδόμηχα να μην γίνει. Αλλά ακόμα και αν γίνει, θα ήθελα να σκεφτούν τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκδοθεί ένα ενιαίο νομικό κείμενο για, τους 27, για τις 27 χώρες σε ό,τι αφορά το καθεστώς των Βρετανών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λούση Ναμπιτζού. Δεν είμαι νομική, δεν είμαι νομικός. Χαίρομαι που μας επιτρέψατε να σας μιλήσω. Ε, ήταν συγκινητικό για μένα. Στο Haringey είμαστε άνθρωποι που ήδη έχουμε επηρεαστεί βαθιά από την ε, προοπτική του Brexit. Εμείς δουλεύουμε με πάρα πολλούς μετανάστες, ιδιαίτερα τους ευάλωτους και αυτοί είναι που έχουν τις μεγαλύτερες ανησυχίες. Παρακαλώ πολύ κάντε ό,τι μπορείτε για να προστατεύσετε τα ανθρώπινα δικαιώματα αυτών των ευαίσθητων, των ευάλωτων ανθρώπων. Ήταν πολύ συγκινητική αυτή η συζήτηση. Ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους αναφέροντες, τη διευθύνουσα ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οπότε θα προφανώς θα διατηρήσουμε ανοιχτές όλες αυτές τις αναφορές. Και θα παρακολουθήσουμε στενά την κατάσταση. καθώς επίσης και την εφαρμογή της, ε, του συστήματος εγγραφής των Ευρωπαίων πολιτών στα Μητρώα Μονιμοκατοίκων του Νομού Βασιλείου. Η, στο 18 Σεπτεμβρίου 2019, το Κοινοβούλιο επανέλαβε ότι επιθυμεί μια έφτακτη έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου με διατήρηση των δικαιωμάτων και εκτιμένων δικαιωμάτων των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασιλείο. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας. Περνάμε στο σημείο 17. Αναφορά 12-11 του 17, 09-23 του 18, 09-25 του 18 και 09-27 του 18. Έχουν σχέση ε, για με την εφαρμογή της οδηγίας 2004 ε, 38 της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκ μέρους της EU Rights Clinic. Υπάρχει ως για όλες αυτές ε, αναφέρον είναι ο Βιτόριο Φαμπρίτσιο. Α, και οι δυο σας είσαστε εδώ. Για τον ίδιο λίγο που σας εξήγησα πριν, σε 15 λεπτά δεν θα έχουμε διαρμηνία. Έχετε 5 λεπτά ο καθένας σας παρακαλώ πολύ αν είναι δυνατόν να συντομεύσετε κιόλα. Αν χρειάζεστε το χρόνο σας, τον έχετε. Απλά σε 15 λεπτά πια δεν θα έχουμε πλέον η Ευχαριστώ. Δύο φορές μιλάμε. Μία φορά παρουσιάζουμε και μία απαντάμε. Εκτός μικροφώνου η παρέμβαση. Ε, η πρόεδρος διευθύνει τη συζήτηση εδώ πέρα. Ε, εγώ του έδωσα το λόγο. Έδωσα το λόγο στον κύριο Αντώνη Μπάλκε. Οπότε έχετε το λόγο. Και παρακαλώ πολύ, κλείστε το μικρόφωνο σας. Σβήστε το μικρόφωνο σας. Ναι, παρακαλώ κύριε Μπάλκε. Um, the... Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο γρήγορος γίνεται. Οι αναφορές αφορούν μια δια... σειρά ζητημάτων σε διάφορα κράτη-μέλη και όλα έχουν να κάνουν με την ε, κακή εφαρμογή της οδηγίας 2047 ε, 438 ε, στην Σουηδία, το Βέλγιο και πρόκειται για ένα θέμα που υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Αυτό το πρώτο, η πρώτη αναφορά είναι το 2007 και η Επιτροπή ε, έχει ξεκινήσει το θέμα από το 2007. Δεν έχει υπάρξει βέβαια κάποια διορθωτική δράση ουσίας έκτοτε. Βλέπετε ότι έχει υπάρξει μια λύση συμβιβαστική ε, που έδωσε η Κομισιόν και οι Σουηδικές Αρχές ε, είναι ο αριθμός συντονισμού, όχι το αφημί. Ε, δυστυχώς αυτό δεν λύνει τίποτα, ούτε πρόκειται. Δημιουργεί μια δεύτερη κατηγορία Ευρωπαίων πολιτών που ζουν στην Σουηδία και δεν έχουν πρόσβαση στην πλήρη γάμα των ιδιωτικών και δημόσιων υπηρεσιών που περνούν μέσα από το ΑΦΜΗ. Επίσης, τα συστήματα πληροφορικής των ιδιωτών δεν αναγνωρίζουν αυτόν τον αριθμό συντονισμού της Σουηδίας, γιατί οι αριθμοί είναι το έτος, ο μήνας και η ημέρα γέννησης των ανθρώπων, ενώ ε, στον αριθμό συντονισμού υπάρχουν κάποια επιπλέον ψηφία. Το σύστημα λοιπόν βγαίνει λάθος. Αν κάποιος ε, γεννηθεί στις 30 ε, ας πούμε Ιουνίου του 1972 και το νούμερο είναι 90, ξεκινάει με 90. Έτσι, το σύστημα δεν αναγνωρίζει το νούμερο. Επιπλέον κόστος λοιπόν δημιουργείται για τις επιχειρήσεις η έκθεση του 2018 εκτιμά ότι το κόστος της δημόσιας αρχές από την εφαρμογή του αριθμού συντονισμού θα είναι 22 εκατομμύρια ε, κορώνες, 2 εκατομμύρια ευρώ το έτος μέχρι το 2022. Ενώ το κόστος αλλαγής μιας απλώς πρότασης στην προβληματική νομοθεσία είναι ελάχιστο αν το συγκρίνουμε πρέπει να αλλάξουμε τον παράγραφο 3 του αντίστοιχου νόμου για τον πληθυσμό της Σουηδίας. Υπάρχουν επίσης προβλήματα σε σχέση με τις ε, συνεχείς περιοριστικές πρακτικές των Σουηδικών αρχών. Δεν έχουν φύγει, δεν έχουν ε, μείνει στην άκρη τα προβλήματα παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει πολλές ουσιαστικές αλλαγές. Υπάρχουν καθυστερήσεις ε, στην κάρτα ε, κατοίκου στην Σουηδία. Υπάρχουν επίσης αρνήσεις έκδοσης. Στη Σουηδία χρειάζεται δύο χρόνια για να βγάλεις ε, μια κάρτα για τα μέλη της οικογένειας, ενώ σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Νόμο αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε έξι μήνες. Άρθρο 10 και 20 της οδηγίας 2014/38 Οι γαλλικές αρχές αυτή τη στιγμή δεν έχουν πλήρως εφαρμόσει την ε, οδηγία 2438 μάλλον. Ε, και de facto δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση από την πλευρά των ε, Ευρωπαίων πολιτών να εγγραφούν στην Γαλλία. Έχουν όμως αυτή την επιλογή αν θέλουν ε, το ίδιο γίνεται και με τους Βρετανούς πολίτες, όμως τώρα δεν ε, τους επιτρέπεται αυτό και αυτό θα έχει σοβαρά προβλήματα. Σε κάποιους που έκαναν ένταση, αίτηση τώρα, τους είπαν «Ελάτε ξανά τον Ιούνιο του 2020». Υπάρχουν εξαιρετικές λοιπόν καθυστερήσεις και προβλήματα και είναι κάτι που μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι δεν έχει γίνει κάτι, ε, κάποια διαδικασία παραβάση για αυτές τις χώρες. Θυμηθείτε τι έγινε το 2007-2008 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ιρλανδία. Η Κομισιόν είχε απειλήσει ότι θα πάει στο δικαστήριο αν δεν επιλύθει το θέμα και σε ένα χρόνο λύθηκε το ζήτημα. Γιατί αυτή η κατάσταση παραμένει εκεί στην Γαλλία και τη Σουηδία. Η συστηματική επίσης ε, επιβεβαίωση των δικαιωμάτων ε, ε, κατοικίας και προμονής από τις βελικές αρχές είναι ένα άλλο ζήτημα. Υπάρχει μια ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι πολίτες στο Βέλγιο που έχουν πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης για τα οποία έχουν συνεισφέρει με εισφορές αν, αν πάντων υπάρχουν τα στοιχεία του εκεί, θα πρέπει να πάνε τα στοιχεία του κατευθείαν στις αρχές μετανάστευση και να δουν αν ε, υφίσταται αυτό το άτομο και να σηματοδοτηθεί αυτός που ψάχνει δουλειά, αυτός που έχει χάσει τη δουλειά του. Το 2014-2016 το Γραφείο Μετανάστευσης λοιπόν είχε πρόσβαση σε δεδομένα σε περισσότερες από 9.000 περιπτώσεις. Είχαμε περίπου 2.000 αποφάσεις ε, που τερμάτιζαν το δικαίωμα παραμονής. 44% του συνόλου των ε, αποφάσεων αποπομπής από τη χώρα. Έτσι λοιπόν υπάρχει το πρόβλημα ότι το σύστημα αυτό ε, είναι σύστημα καταρχάς το οποίο είναι προβληματικό και ε, δυστυχώς φαίνεται ότι ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί πως οι βελικές αρχές έχουν το δικαίωμα να το κάνουν. Το θέμα είναι ότι οι βελικές αρχές θεωρούν πως όταν δεν έχεις δικαίωμα στις παροχές κοινωνικής ασφάλισης, ε, δεν έχεις δικαίωμα και παρανομής, παραμονής. Και πρέπει να φύγεις από τη χώρα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα τέλειωσε ο χρόνος μου. Θα δώσω το λόγο στο συνάδελφο που θα μιλήσει για τα προβλήματα στη Σουηδία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ελπίζω άλλη φορά να έχω περισσότερο χρόνο. Είναι δυνατόν σε δύο λεπτά να τα πείτε. Ναι, απλώς δύο σχόλια. Πρώτον, ο αριθμός συντονισμού στη Σουηδία και η πρόταση που έγινε από την Σουηδική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως είπε ο Άντωνη, ε, έχουν ε, αξιολογηθεί από μια έκθεση του Scott Worker που είναι ε, μια έκθεση η οποία αναφέρει πως υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα ως προς αυτό τον αριθμό συντονισμού. Το θέμα είναι και με την έκδοση και με τις αλλαγές. Αυτή τη στιγμή οποιαδήποτε αλλαγή στο σύστημα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Αυτή την άποψη την επιβεβαίωσε και η Σουηδική κυβέρνηση το Σεπτέμβριο του 2019 λέγοντας ότι ναι, εργαζόμαστε επί του προβλήματος, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε κάποια αλλαγή στο σύστημα του αριθμού συντονισμού για να επιτρέψουμε στους Ευρωπαίους πολίτες να εγγραφούν με τον ίδιο τρόπο που εγγράφεται όποιος έχει αφήμη. Το δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με τη διαδικασία επί παραβάση που ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εναντίον της Σουηδίας για την ε, οδηγία που αφορά στην επανένωση των οικογενειών. Αυτή η διαδικασία επί παραβάση αναφέρει στην απάντησή της η Κομισιόν ότι ο νόμος που προκαλεί τόσα προβλήματα στην Σουηδία που έχει να κάνει με τον μητρό τον του πληθυσμού ε, είναι προβληματικός διότι έχουμε πολίτες τρίτων χωρών που έχουν τεράστια αναμονή για την έκδοση αφημί και το γεγονός ότι το Σκέτερ ζητά από αυτούς τους ανθρώπους να περιμένουν 12 μήνες ή παραπάνω για να πάρουν το φημί τους είναι παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Η ερώτησή μου στην Επιτροπή είναι γιατί αυτή, αυτό το ενδιαφέρον επιχείρημα έγινε για πολίτες τριών χωρών και ξεκίνησε διαδικασία επί παραβάση και γιατί δεν γίνεται τίποτα ή σχεδόν τίποτα για τους Ευρωπαίους πολίτες και τη παραβίαση της δικής τους ας πούμε δυνατότητας για ίση μεταχείριση. Ευχαριστώ για τα 49 δευτερόλεπτα. Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Η Επιτροπή έχει, Η Επιτροπή έχει το λόγο τώρα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Καθώς και όλους τους θέλω να ξεκινήσω με τις αναφορές σε σχέση με την Σουηδία. Συμμεριζόμαστε τις ανησυχίες. Προσπαθήσαμε να λύσουμε το ζήτημα αυτό με τους Σουηδικές αρχές, όχι όμως με την ταχύτητα που θα θέλαμε. Είμαστε εδώ ακριβώς για να συζητήσουμε για το αφημί αυτό, το τον αριθμό mid-row, είναι πάρα πολύ δύσκολο το σύστημα για, τους, ε, για, του, για τις IT να το χρησιμοποιήσουν. Μετά από την αναφορά ήρθαμε σε επαφή με τις Σουηδικές Αρχές και επιμείναμε ε, στο ότι ο αριθμός αυτός συντονισμού θα πρέπει να λύσει τα προβλήματα όλων αυτών των πολιτών τόσο για δημόσιες αρχές όσο και για ιδιωτικούς φορείς το, η Επιτροπή ζήτησε ε, μία αναφορά για την πρόοδο του ζητήματος. Έχουν γίνει βήματα, αλλά πραγματικά δεν έχουμε φτάσει εκεί που θα θέλαμε και πρέπει να αναλογιστούμε ποια είναι τα επόμενα ζήτημα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ασφάλιση υγείας, η Σουηδική κυβέρνηση άλλαξε τις κατευθυντήριες γραμμές. Περισσότερες ιδιωτικές ασφάλειες γίνονται αποδεκτές και ε, εκτιμάται κατά περίπτωση το σύστημα της ασφάλειας της υγείας, ούτω ώστε να μπορούν να αποφασίζουν ποιο έχει το δικαίωμα, ποιο έχει το δικαίωμα της ε, μόνιμης παραμονής. Δεν έχουμε λάβει παράπονα για αρκετό καιρό. Πολύ πολύ πρόσφατα μας ήρθαν κάποια παράπονα και από την δική σας την μεριά. Ε, και εμείς ε, επικοινωνήσαμε τις ειδικές Αρχές για να συζητήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εντοπίσουμε πού ακριβώς βρίσκονται τα προβλήματα. Είμαστε σε επικοινωνία με τις ειδικές Αρχές. Σε ό,τι αφορά τώρα την καθυστέρηση στην έκδοση αδειών παραμονής, είναι δεδομένο ότι οι Σουηδικές αρχές είχαν ένα πρόβλημα εξαιτία της μεταναστευτικής κρίσης από το 2015 και μετά. Ε, πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν αυξημένο αριθμό ατόμων που έρχονται στην χώρα. Είχαμε μια ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις στατιστικές, σε ό,τι αφορά τα νούμερα. Υπήρξε μια βελτίωση, αλλά όχι όσο ελπίζαμε. Επομένως, ναι, και πάλι έχουμε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας με τις Σουηδικές Αρχές και περιμένουμε να ακούσουμε τα νέα τους αυτόν το μήνα. Σε ό,τι αφορά τώρα τις α, ανησυχίες σχετικά με την Γαλλία. Οι πολίτες δεν έλαβαν κάρτα παραμονής. Ίσως ε, θα πρέπει να πούμε ότι γιατί για μια περίοδο μεταξύ τριών και πέντε μηνών δεν υπάρχει τέτοιου τύπου έγγραφο, αλλά η Γαλλία βασίζεται σε έναν εθνικό νόμο, σύμφωνα με τον οποίο μπορεί κάποιος να λάβει την άδεια παραμονής κατόπιν αίτησης. Υπήρχε μια αύξηση των αιτήσεων για τέτοιου τύπου έγγραφα. Είμαστε σε επαφή με τις α, γαλλικές αρχές, ούτως ώστε να α εξασφαλίσουμε ότι οι κανόνες εφαρμόζονται και πιο συγκεκριμένα για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι πολίτες ή πιο συγκεκριμένα οι Βρετανοί πολίτες θα μπορούσαν να λάβουν τέτοιου τύπου έγγραφα, δεν θα επηρεαζόταν η νομιμότητα της παραμονής του σε ένα σενάριο σκληρού Brexit ή Brexit κατόπιν συμφωνίας. Σε ό,τι αφορά το Βέλγιο τώρα, οι ανησυχίες των αναφερθέντων, των αναφερόντων, έχουν να κάνουν με τα άτομα που ενώ έχουν κάποιους πόρους διαβίωσης, παράλληλα κάνουν αίτηση για κοινωνικά επιδόματα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να οδηγήσει σε αντικρουόμενα μηνύματα, δηλαδή έχει κανείς τα μέσα για να ζήσει ή έχει ανάγκη από κοινωνικά επιδόματα. Η εξέταση των αιτήσεων διαρκεί τρεις μήνες περίπου και υπό αυτό το πρίσμα θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όντως ένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να χρειάζεται να επαληθεύει συστηματικά την νομιμότητα α, της άδειας παραμονής ενός πολίτης. Αν όμως από την άλλη μεριά η υπάρχουν σημάδια ότι ένα κράτος μέλος δεν συμμορφώνεται με την οδηγία και πρέπει να κάνει τέτοιου τύπου επαληθεύσεις. Η οδηγία δηλώνει επίσης ότι η αίτηση για κοινωνικό επίδημα δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αυτόματη επαλήθευση της νόμιμης παραμονής. Στην περίπτωση όμως που κανείς θεωρείται ότι εκμεταλλεύεται τα κοινωνικά επιδόματα, τότε η ιδιαίτερη κατάσταση του συγκεκριμένου τόμου θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη, να εξετάζεται, καθώς επίσης και ο βαθμός της βοήθειας που έχει λάβει. Το σύστημα που χρησιμοποιείται επιτρέπει στο κράτος μέλος να λειτουργήσει κατά αυτόν τον τρόπο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι δεν εμποδίζεται, δεν θα πρέπει να εμποδίζεται ένα κράτος μέλος να ελέγχει τη νομιμότητα της άδεια παραμονής ενός ατόμου αν θεωρούν ότι υπάρχουν συνθήκες, προϋποθέσεις που να πληρούν τέτοιου τύπου ελέγχου. Σας ευχαριστώ πολύ. Sí, Presidenta, lamento interrumpir. Me gustaría preguntarle si usted va a abandonar